Καθίστε σιγά σιγά. Monsieur Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω όλους στην 33η Ολομέλεια της Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Υπάρχουν αντιρρήσεις στην ημερήσια διάταξη που σας έχει κοινοποιηθεί. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Άρα εγκρίνεται. Το ίδιο ισχύει και για τα πρακτικά της εκατοστής ης Ολομέλειας του Δεκεμβρίου πέρσι. Υπάρχουν σχόλια, όχι. Άρα εγκρίνονται τα πρακτικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, τις, ε, οι τελευταίες εβδομάδες ε, ήταν τραγικές. Σκέφτομαι τον δήμαρχο του Γκτάνσκ, τον Πάβελ Αβραμοβίτς, ο οποίος ε, δυστυχώς μαχαιρώθηκε μέσα στα πλαίσια μιας εκδήλωσης και μετά την επόμενη ημέρα υπέκυψε στα τραύματά του. Το ίδιο αφορά την 11η Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο με την τρομοκρατική ενέργεια. Μεταξύ των θυμάτων είχαμε δύο δημοσιογράφους, έναν Ιταλό και έναν Πολωνό, με τους οποίους είχαμε συνεργαστεί μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών. Δεν ξεχνάμε και τον Βιτσέντε Άλβαρες Ρίσες, που ήταν πρόεδρος των Αστουριών και τον Γιούρι Πιλ Εσθονό και αντιδήμαρχο, τους οποίους χάσαμε. Θα ήθελα να τηρήσουμε στη μνήμη τους ενός λεπτού σύγκρισης, Merci. Σας ευχαριστώ. Chers Αγαπητοί συνάδελφοι, εξ ονόματός σας θα ήθελα να ε, χαιρετήσω μία αντιπροσωπή από το Γκτάνσκ υπό την κυρία Ντούλκεβιτς η οποία ασκεί καθήκοντα δημάρχου και τον αδελφό του Πάβελ Αντάμοβιτς, τους οποίους χαιρετίζω θερμά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία για να τιμήσουμε τη μνήμη του Πάβελ και να υπογραμμίσουμε τη σημασία της μάχης κατά της μυσαλλοδοξίας καθώς και την υπεράσπιση των μειονοτήτων και των ε, διαφόρων σεξουαλικών μειονοτήτων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, ε, αντιδήμαρχο της, ε, του Γκτάνς και μετά τον, ε, στον Εσθονό αντιδήμαρχο. During the communist era,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 Ο κύριος Βοσνιακ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, ήταν ε, μεγάλη απώλεια όχι μόνο για την ε, πολωνική αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών ολόκληρη η Ευρώπη υπέστη μια απώλεια η Ευρώπη η οποία βασίζεται στις κοινέ αξίες μας μέχρι πρόσφατα ο Πάβελ ήταν εδώ μαζί μας σε αυτήν εδώ την έδρα όπου τώρα βλέπετε τη φωτογραφία του και τα λουλούδια. Την μοιραία μέρα της 13ης Ιανουαρίου μαχαιρώθηκε, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης που οργανώνεται κάθε χρόνο που στόχο έχει να συγκεντρωθούν λεφτά για να αγοράσουν ε, ιατρικό εξοπλισμό για τις μονάδες νεογνών στα πολωνικά νοσοκομεία. Χιλιάδες ε, εθελοντές ε, βγαίνουν στους δρόμους για να μαζέψουν λεφτά από τους Πολωνούς και οπωσδήποτε και ο Πάβελ Αντάμοβιτς ήταν εθελοντής και εκείνη τη μέρα κατά τις 8 η ώρα συνήθως έδινε το ποσό που είχε συγκεντρωθεί από την εκδήλωση. Το ίδιο συνέβη και στο Γκτάνσκ λοιπόν. Ο Πάβελ ήταν στη σκηνή, ευχαριστούσε τον κόσμο για την γενεοδορία του και μόλις είπε αυτά τα λόγια, του επιτέθηκε ο δολοφόνος. Το έγκλημα αυτό, οπωσδήποτε, έχει πολιτική χρειά και πλαίσιο, είναι σαφές για όλους μας, ε, για δύο λόγους. Αφού μαχαίρωσε τον Αντάμοβιτς, ε, ο δολοφόνος μας είπε ε, γιατί το έκανε. Είπε ότι ήθελε να εκδικηθεί το κόμμα του γιατί ο Αντάμοβιτς ήταν ε, μέλος του κόμματος της Πλατφόρμας Πολιτών. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο το λέμε. Εδώ και μήνες ο κύριος Αντάμοβιτς έκανε μια εκστρατεία για να κατέβει στις επόμενες εκλογές και ε, δεχόταν επιθέσεις από τα ΜΜΕ και διάβαζε κανείς διάφορες ε, ψευδείς κατηγορίες εις βάρος του με σαφή στόχο. να μην ε, κερδίσει τις εκλογές. Και να το πούμε αυτό, γιατί το πολιτικό πλαίσιο αυτού του φρικτού εγκλήματος πρέπει να το θυμόμαστε. Σήμερα λοιπόν έχουμε έρθει εδώ για να τιμήσουμε τον κύριο Ντάμοβιτς, αλλά νομίζω πως ο κύριος Στρούγκ ε, είναι σε καλύτερη θέση ε, για να μας τα πει, γιατί είναι Περιφερειάρχης Πομερανίας και πρωτεύουσα της Πομερανίας είναι το Γκτάνσκ. Θα ήθελα λοιπόν να του δώσω τον λόγο πριν από αυτό να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο για τα συλληπιτήριά σας, για την παρουσία σας στην κηδεία. Ευχαριστώ όλους όσους μας συλληπίθηκαν για τα λόγια σας, για τις χειρονομίες σας και τα καλά σου λόγια για τον ε, κύριο Ανταμόβιτς. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κρατήσετε τη μνήμη του ζωντανή. Είναι και πάντα θα είναι πολύ σημαντικό μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη μαρτυρία, κύριε Βοσνιάκ, και το λόγο έχει ο κύριος Στρούκ. Szanowne koleżanki i koledzy, staję dziś przed Państwem, by uczcić pamięć naszego kolegi, przyjaciela. Θα θέλαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του Πάβελ Αντάμοβιτς όλοι το δήμαρχο του Γκτάνσκ κάτι το οποίο έγινε και κατά τη διάρκεια μίας συναυλίας που έγινε για καθαρά φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στόχος ήταν να βοηθήσουμε τους πιο αδύναμους. Το θύμα ήταν ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, ο οποίος εργάστηκε δημοσία για να αντιμετωπίσει τη μυσαλλοδοξία και τη ρητορική μίσους. Τον είδαμε και εδώ στις Βρυξέλλες λίγο καιρό πριν συμμετείχε στις συζητήσεις της Ολομέλειας και πριν είχαμε συζητήσει ειδικά σχέδια για το Γκντάνσκ για τη νέα του θητεία η οποία είχε και μόλις αρχίσει. Μιλούσε για την αγαπημένη του πόλη, την ε, κατονόμαζε ως πόλη της ελευθερίας και της αλληλεγγύης, κάτι τον οποίο, το οποίο τον απασχόλησε από τα νεανικά του χρόνια μέχρι και την πρόσφατη θητεία του ως δήμαρχος. Και το έλεγε αυτό όχι επειδή γεννήθηκε η Σολινταρνόσκ στο Γκτάνσκ, το κίνημα αυτό της αλληλεγγύης, αλλά και γιατί θεώρησε ότι το Γκτάνσκ είναι μια πόλη ελευθέρων πολιτών, ανεξάρτητα από το θρησκευμά τους ή τις απόψεις των πολιτών. Θεωρούσε ότι η αλληλεγγύη βρίσκεται στο κάθε βήμα αυτής της πόλης, όπου κανένας δεν αποκλείεται από τον κοινωνικό αυτό ιστό. Χάρη στο Πάβελ, το Πτάνσκ είναι μια ελεύθερη πόλη, ελεύθερη αλληλέγγυα και στα πλαίσια της ε, λειτουργίας μέσα στην ισότητα. Ο αντιδήμαρχος τώρα έχει αναλάβει καθήκοντα. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτές οι αξίες υπάρχουν στη, στο Gdansk και θα υπάρχουν όσο υπάρχει ζωή. Ο Παύλ Ανταμόβιτς είχε υποστηρίξει τους μετανάστες, τις μειονότητες, ήταν δραστήριος στην ανατολική εταιρική σχέση και στην Επιτροπή μας είχε ταχθεί υπέρ μίας ε, δυνατής κοινωνίας των πολιτών για τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Η δολοφονία του μας σημάδεψε γιατί είχε δεχτεί πολλές επιθέσεις κατά τους τελευταίους μήνες της ζωής του από δημόσια μέσα και από πολιτικά κόμματα. Αυτό το βλέπουμε στην Πολωνία σε καθημερινή βάση, κάτι το οποίο οδηγεί σε τραγικά αποτελέσματα σε αυτή την τραγική εποδό. Γι' αυτό αύριο πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα σε σχέση με την αντιμετώπιση της ρητορική μίσους και ελπίζω αυτή να είναι η απαρχή δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να δώσουμε τέλος σε αυτές τις κατηγορίες, σε αυτό το κατηγορητήριο που υπάρχει στην καθημερινή μας ζωή. Πάβελ, θα ήθελα να σε αποχαιρετήσω σήμερα στην Επιτροπή των Περιφερειών και θα ήθελα να επαναλάβω λέξεις που είχαμε ακούσει πολλές φορές από το δικό σου στόμα. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το δήμαρχο του Γκτάνσκ και η δράση του θα μας καθοδηγεί πάντα. Αύριο θα αρχίσουμε τις εργασίες μας με ένα ψήφισμα κατά της ρητορική μίσους και τα, κρίμα και τα εγκλήματα ρητορική μίσους. Θα είναι ένα στεναρό μήνυμα και προς τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στις 10 Απριλίου στην επόμενη Ολομέλεια θα οργανώσουμε μία εκδήλωση, επίσημη εκδήλωση, έτσι ώστε το φουαγέ ε, του πέμπτου ορόφου να μετονομαστεί. Να γίνεται λόγος για χώρο Πάβελ Αντάμοβιτς και φυσικά θα υπάρξει και ένα ε, μνημείο υπομορφή μιας τιμητικής ε, πλάκας. Θα καλέσουμε του συγγενείς του Πάβελ καθώς και τους εκπροσώπους της πόλης του Γκτάνσκ καθώς και εκπροσώπους της πολωνικής κοινωνίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα ήθελα να ξαναβρεθούμε στις 10 Απριλίου και όλοι μπορείτε να υπογράψετε το βιβλίο συλληπιτηρίων που βρίσκεται στην είσοδο της αίθουσας αυτής. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα επανερχόμαστε στις εργασίες μας ευχαριστώντας τον Επίτροπο Ναύρα γιατί παρευρέθηκε και στο πρώτο μέρος αυτής της εκδήλωσης, εκδήλωσης μνήμης. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην Ολομέλειά μας καταδεικνύοντας τη σημασία που προσδίδουμε στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Πέρυσι ε, πανηγυρίσαμε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμού με τη συμμετοχή 6.000 πολιτών. Η Επιτροπή, η Επιτροπή μας ήταν πολύ δραστήρια και χαιρόμαστε για αυτή την επιτυχία που διαιωνίζει αυτή την παράδοση όπως είχε εγκριθεί πέρσι το Δεκέμβριο και που αναγνωρίζει και την εδαφική συνεισφορά. Ήδη εξ αρχής η Επιτροπή μας θεώρησε ότι φέτος θα πρέπει ο πολιτισμός και η εκπαίδευση να είναι δύο βασικοί πυλώνες της δυναμικής πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρσι το Μάιο μιλήσαμε για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω του πολιτισμού. Αυτό το θέμα παραμένει επίκαιρο εν ώψη της διάσκεψης στο Σιμπίου και των ευρωεκλογών γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί πλήρως. Υπάρχει μία νέα πρόταση για το Εράσμους με χρηματοδότηση 30 δις για να τριπλασιάσουμε τον αριθμό συμμετεχόντων. Επίσης θα δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης μέχρι το 2025, μια πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν σύνορα στην εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα. Σημεριζόμαστε αυτό το στόχο και η Επιτροπή των Περιφερειών είναι υπέρ της Creative Europe μέσα στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς για να φτάσουμε στα 2 δις ευρώ για μια εγκάρσια προσέγγιση του πολιτισμού και τον ορισμό των άλλων ευρωπαϊκών, των συναφών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να θεωρηθεί ένα στρατηγικό πόρος για την Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να προωθεί τα αναδυόμενα οικοσύστηματα των πόλεων μας μέσα στα πλαίσια της, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής. Η Επιτροπή δέχεται την πρωτοβουλία ανακάλυψε την Ευρωπαϊκή Ένωση Discover EU έτσι ώστε οι νέοι να ανακαλύψουν τις ε, ευρωπαϊκές χώρες. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας στην πρόταση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και τη νέα στρατηγική υπέρ της νεολαίας. Στα πλαίσια αυτά τασόμαστε υπέρ μιας πολιτικής για την νεολαία που να εντάσσεται σε όλες τις πολιτικές οριζόντια μέσα στα πλαίσια της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας. Οι δύο γνωμοδοτήσεις για το έρασμους και την Δημιουργική Ευρώπη που θα εγκρίνουμε στη συνέχεια υπογραμμίζει την θέληση των περιφερειών να συμμετέχουν σε έναν ευρωπαϊκό χώρο για την εκπαίδευση και τη νέα ατζέντα του πολιτισμού μας. Αυτό το επιβεβαιώνει και η σημερινή συζήτηση. Τώρα θα ήθελα να σας δώσω το λόγο κύριε Επίτροπε. Thank you, President. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε από τα μέλη της Επιτροπής κυρίες και κύριοι. Η επένδυση στους ανθρώπους, ειδικά τους νέους, στην εκπαίδευσή τους, στην δημιουργικότητά τους, έχει κέρια σημασία για να φτιάξουμε μια συνεκτική και ανθεκτική Ευρώπη για το μέλλον. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερο για το ότι η Κομισιόν ε, το έχει θέσει αυτό στην καρδιά της πρότασής της για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προπολογισμό μετά το 2020. Αυτό αφορά ιδιαίτερω δύο μελλοντικά προγράμματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Την Δημιουργική Ευρώπη και το Εράσμου. Αναμένω την συζήτησή μας και θα ήθελα ήδη να σας ευχαριστήσω για την στήριξή σας συγκεκριμένα να ευχαριστήσω τον Άνταμ Κοράτσο και την κυρία Ολίκα Χίλερ τους εισηγητές η εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι ξανά στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκαθάρισαν ότι θέλουν να δουν περισσότερα πράγματα εδώ και χάρηκα που είδα αυτές τις προτάσεις ε, κατά το 2018. Προτάσεις που στόχο έχουν να φέρουν μια αλλαγή στην συνεργασία μας ε, και να καταφέρουμε να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Οι προτάσεις για τη μελλοντική δημιουργική Ευρώπη και τα προγράμματα Εράσμους που υποβάλαμε πέρσι βασίζονται σε αυτό. Θέλουμε η Ευρώπη να ωφεληθεί πλήρως από τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και να υπάρχει μια ευρωπαϊκή περιοχή εκπαίδευσης μέχρι το 2025 για να παραμείνει η Ήπειρός μας ανταγωνιστική και να υπάρχει ενότητα μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών, των κοινοτήτων και των ανθρώπων. Να ξεκινήσω από τη Δημιουργική Ευρώπη. Προτείνουμε να αυξηθεί ο προπολογισμό κατά το 1 τρίτο σε 1,85 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το έχουμε σχεδιάσει ώστε να στηρίξει πλήρως τις πολιτικές προτεραιότητες που παρουσιάζει η νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον πολιτισμό που εγκρίθηκε πέρσι. Βασικό βασικός μας στόχος είναι το πρόγραμμα αυτό να είναι ευέλικτο. Χρειάζεται καλύτερη ισορροπία μεταξύ της οικονομικής, της κοινωνικής και της διεθνούς πτυχής του πολιτισμού, ενώ θα υπάρχει οπωσδήποτε και περιθώριο για δημιουργία και καινοτομία. Θέλουμε επίσης να εισαχθούν καινοτομίε που θεωρούμε ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Συγκεκριμένα, έχουμε προτείνει την στήριξη των καλλιτεχνών που θέλουν να πάνε στο εξωτερικό και έχουμε περιλάβει και νέες τέχνες όπως η μουσική. Αυτό κάποιους σας ανησυχεί αλλά σας παρακαλώ και σας διαβεβαιώ. Τα περισσότερα χρήματα θα πάνε σε οριζόντιες δράσεις που καλύπτουν όλους τους κλάδους. Όμως, οι διαπραγματεύσεις επί του προπολογισμού είναι δύσκολες Περισσότερο από ποτέ, ο υπολογισμό χρειάζεται συμμάχους στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσοι πιστεύουν στην δύναμη του πολιτισμού, στο να μετασχηματίσει τις ε, περιφερειές μας, ε, πρέπει να το δείξουν. Χαίρομαι λοιπόν που το κάνετε και βασίζομαι σε εσά ε, να με βοηθήσετε να πείσω τις κυβερνήσεις ότι είναι μια εξαιρετική επένδυση η χρηματοδότηση του πολιτισμού αποδίδει σε οικονομικούς και κοινωνικούς όρους η δημιουργική Ευρώπη θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην στήριξη των προτεραιοτήτων που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον πολιτισμό. Χαίρομαι για το ότι το σχέδιο γνώμοδότησης ε, καλωσορίζει την ατζέντα αυτή και χαίρομαι που στηρίζεται τους στόχους ε, της οικονομικής και της εξωτερικής πολιτικής και τις οριζόντιες δράσεις που περιλαμβάνουν κάποιες ε, πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να διαφυλάξουν την πολιτιστική κληρονομιά πέρα από το έτος 2018. Έχετε έναν κεντρικό ρόλο να παίξετε για να υλοποιηθούν αυτά. Παραδείγματος χάρη, όταν μιλάμε για τις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες και τον πολιτισμό. Τώρα, να αναφερθώ στο Εράσμους. Ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση Θεωρούμε όμως ότι μπορεί να γίνει πιο επιτυχημένο. Γι' αυτό την επόμενη περίοδο μετά το 2020 θέλουμε να διπλασιάσουμε τον προπολογισμό στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι θα τριπλασιαστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων ε, σε όλους τους κλάδους που καλύπτει το πρόγραμμα. Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Βεβαίω, ε, το θέμα δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Θέλουμε να φτάσουμε σε περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι ίσως συνήθως δεν συμμετέχουν σε τέτοια έργα ανθρώπους από μειονεκτικές περιοχές ίσως ή σε μειονεκτικά περιβάλλοντα. Θέλουμε λοιπόν το μελλοντικό Εράσμους να το επιτύχουμε αυτό. Είναι ένας απλός τρόπος έτσι ώστε οι νέοι να ερευνήσουν την πολιτισμική ποικιλομορφία της Ευρώπης, να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους και να καταλάβουν τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν να ανακαλύψουν την Ένωση και να την δουν να αναπτύσσεται. Γι' αυτό έχουμε προτείνει έναν προπολογισμό 700 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος 7 ετών. Έτσι, θα μπορέσουμε να δώσουμε σε 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους την ευκαιρία να δουν την Ευρώπη από πρώτο χέρι και να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες. Οι περιφέρειες, οι πόλεις ε, και οι τοπικές αρχές έχουν μεγάλο ρόλο να παίξουν εδώ. Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω άλλον έναν σημαντικό παράγοντα στις προτάσεις μας έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί το Εράσμος με κονδύλια από άλλα προγράμματα. Η συνέργεια με άλλα προγράμματα είναι πάρα πολύ σημαντική όταν μιλάμε για την αύξηση κονδυλίων επιτυχών προγραμμάτων που μπορούν να γίνουν μια τυποποιημένη πρακτική για μια χώρα ή για έναν κλάδο. Επίσης μπορεί έτσι ένα πρόγραμμα σαν το Εράσμος να γίνει πιο προσβάσιμο για τους ε, νεαρούς ε, από μειονεκτικές ε, ομάδες. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα της κοινή διαχείρισης και των διαρθρωτικών κονταλίων. Εδώ πέρα λοιπόν ηγετικό ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες και θα ήθελα να κατευθύνετε κάποια από αυτά τα κονδύλια ώστε να συμπληρώνουν τη στήριξη που δίνουμε με το Εράσμος. Κυρίε και κύριοι, σε τέσσερις μήνες οι πολίτες θα ψηφίσουν για την κατεύθυνση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της Υπήρου. Εάν λοιπόν πιστεύετε σε αυτήν την επιλογή θα πρέπει και εσείς να ζητήσετε από τους νέους να ψηφίσουν. Εμείς ήδη πιστεύουμε σε αυτό το μέλλον, επενδύουμε στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στους νέους. Θέλουμε να επενδύσουμε σε αντοχή, σε κοινότητες που θα βασίζονται σε κοινέ αξίες όπως η κατανόηση και ο σεβασμός. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με την συνεργασία. Χαίρομαι που θέλετε να λάβετε μέρος σε αυτή την προσπάθεια και αναμένω να συνεχίσουμε αυτή την κοινή πορεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα αυτά που μα δώσατε και για την παρέμβασή σα την συζήτηση. Να δώσουμε το λόγο στα μέλη μα τώρα και να ξεκινήσουμε καταρχά με τι πέντε πολιτικέ ομάδε και του πρώτου αντιπροέδρου. Και μετά θα πάρουν το λόγο οι συγητέ και μετά θα ακούσουμε και την παρέμβαση των ασκούμενων σε ό,τι αφορά μια ημερίδα για τα δικαιώματα των γυναικών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους ασκούμενους μας για την επιτυχία τους αυτή. Επίσης, έχουμε και τους μεμονωμένους ομιλητές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Εδώ να σας υπενθυμίσω ότι το ανώτατο όριο είναι δύο λεπτά και θα προσπαθήσουμε να τα ολοκληρώσουμε όλα αυτά στο προδιαγραμμένο χρονικό διάστημα. Και παρακαλώ να κοιτάτε τις ε, οθόνες ε, και γενικά να δείξετε αυτοσυγκράτηση το χρόνο ομιλίας. Είναι πιο ευχάριστο και για σας και για μένα να σταματάτε την ώρα σας και να μην χρειάζεται να σας διακόπτω. Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν το λόγο έχω, έχει ο κύριος Στιμάτε Κομισάρ, uh, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται να κοιτάξουμε το θέμα της ανεργίας των νέων. Είχαμε πολλές εμπειρίες από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κοινωνική ένταξη. Ε, είχαμε πολλά προγράμματα, ωστόσο τα ποσοστά της ανεργίας ε, είναι πάρα πολύ υψηλά. Εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ υψηλά σε ό,τι αφορά τους νέους σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τα προγράμματα αυτά, τα οποία έχουν αποδειχτεί επιτυχή, όπως για παράδειγμα το Erasmus+. Και προσβλέπουμε και χαιρόμαστε που διπλασιάστηκε ο υπερπολογισμό για τα προγράμματα αυτά. Και θα συνεχίσω στα ουγγρικά. Κύριε Επίτροπε, Η πολιτική εκπαίδευση ε, και παιδεία ε, των νέων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει συνεχώ να προωθήσουμε. Συνεχώ, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Το πρόγραμμα Erasmus και το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη Creative Europe βοηθούν για την εξέβρεση καινοτομικών τρόπων αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων, για παράδειγμα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πανευρωπαϊκή τέτοια τάση, αλλά αυτό συνήθω πλήττει πιο πολύ τι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη. Με αυτά τα προγράμματα λοιπόν υποστήριξη μπορούμε να κατακτήσουμε στρατηγικέ. Στρατηγικέ οι οποίε πραγματικά θα προωθήσουν τι γνώσει των νέων προκειμένου να έχουν δεξιότητες και ικανότητες που να χρειάζονται και οι χώρες τους οι πατρίδε του. Γι' αυτό επίση είναι σημαντικό να προωθήσουμε και το σκέλο τη ψηφιακή εκπαίδευση για την απόκτηση τέτοια γνώση και ανταλλαγή τέτοιων εμπειριών. Αυτό που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαμορφώσουμε με καλύτερο τρόπο είναι να εξοπλίσουμε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα σχολεία με ψηφιακό εξοπλισμό και στις περιοχές εκείνε όπου δεν έχει γίνει αυτό ακόμα. Γιατί στα νέα επαγγέλματα θα αυξηθούν οι θέσεις εργασία και στο μέλλον. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν για τα κρατημέλη τα οποία αντιμετωπίζουν στην παρούσα φάση ακόμα προβλήματα σε ό,τι αφορά την απασχόληση των νέων. τα τοπικά και περιφερειακά συμβούλια έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν εδώ, γιατί αυτά είναι που υποστηρίζουν τα σχολεία και τα σχετικά σχολικά δίκτυα. Είναι λοιπόν ανάγκη, έχουμε ανάγκη να δραστηριοποιηθούμε στον τομέα αυτό και να παίξουμε το ρόλο που μας αναλογεί. Το Erasmus τώρα ως πρόγραμμα πώς μπορεί να βοηθήσει με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με γνώσης, ε, παροχή γνώσεων μπορούμε να μειώσουμε τα χάσματα μεταξύ των περιοχών, των περιφερειών και θα πρέπει και στο μέλλον να λάβουμε σχετικές απαντήσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω σε ό,τι αφορά και τα προγράμματα εκπαίδευση online στο διαδίκτυο ότι αυτά θα πρέπει προφανώς να βοηθούν και τις απόμακρες περιοχές. Χρειαζόμαστε λοιπόν το πρόγραμμα Erasmus Plus προκειμένου η ομαδική αυτή εργασία η συνεργασία και όλα τα προγράμματα άσκησης να βοηθήσουν στην ένταξη των νέων. Εξ ονόματος λοιπόν του ΕΛΚ θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ζητήσω από τον Επίτροπο την υποστήριξή του. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλητρία, η Ουλίκη Χίλερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Επίτροπε, έχω μεγάλη χαρά και τιμή να κάνω μια, σύμβαση, μια σύντομη παρέμβαση εξ ονόματος της ομάδας μου και θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως για το γεγονός ότι σήμερα βάζουμε στο επίκεντρο το θέμα της εκπαίδευσης των νέων, το θέμα του αθλητισμού, το θέμα του πολιτισμού Ασφαλώς ε, είναι σημαντικά τα θέματα αυτά, γιατί η εκπαίδευση, οι νέοι είναι το μέλλον μα και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μα. Και θα επικεντρωθώ προφανώ στο πρόγραμμα Erasmus ε, γιατί κατήρτησα και την σχετική τροπολογία, συγγνώμη, τη σχετική γνωμοδότηση που θα ψηφίσουμε και διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει σημαντικά στο να καταστεί η Ευρώπη πιο βιώσιμη για πολλούς, στη μείωση των εμποδίων και την αύξηση της ποιότητα στον τομέα τη εκπαίδευση. Αυτό θεωρώ για όλους μα ότι αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία. Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Erasmus Plus 2017 καταδεικνύει ότι όχι μόνο συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό πιο πολύ παραπότε, 800.000, αλλά και ότι αυξήθηκε περαιτέρω ο αριθμός των ε, υποστηριζόμενων έργων και projects. Επίσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι το Erasmus Plus από το 2021 θα λάβει ε, μια σωστή συνέχεια, ένα καλό διάδοχο πρόγραμμα. Και καλωσορίζουμε ιδιαίτερο το γεγονό ότι διπλασιάζει, προτείνει διπλασιασμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προπολογισμού του προγράμματο και αυτό θα ωφελήσει όλους, από παιδιά μέχρι και νέους, να έχουν την ευκαιρία να βιώσουν με καλύτερο τρόπο την Ευρώπη. Την Αφορά αυτό φυσικώς και φοιτητές και μαθητές, αλλά και συμμετέχονται στα προγράμματα ενήλικης, ε, ενήλικων για διαβίωση Ένα σημαντικό επίσης στοιχείο είναι η φιλόδοξη της τριπλασιασμός. 12 εκατομμύρια συμμετέχοντες ε, αν απλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Γιατί αυτό μας το λένε χρόνια τώρα οι ε, οι συμμετέχοντες. Και στην Βρέμη το ακούσαμε, αλλά και εδώ στις Βρυξέλλες. Και σίγουρα εμποδίζονται κάποιοι από το να υποβάλουν αίτηση. Και αυτό ισχύει κυρίω για μικρέ οργανώσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρξει μια απλοποίηση στο σημείο αυτό, αλλά να υπάρχουν και δυνατότητε διαβούλευση. Γιατί είναι σημαντικό και στι εθνικέ υπηρεσίε να υπάρχουν άτομα τα οποία να μπορούν να υποστηρίξουν την όλη διαδικασία υποβολή έντασης και να βοηθήσουν και σε περίπτωση σύγκρουση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με τι εθνικέ υπηρεσίε. Και να πω και δύο λόγια τώρα για αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από δική μα πλευρά ε, είναι πολύ ευπρόσδεκτο το γεγονό ότι ανοίγει η οργάνωση και για άτομα με πιο περιορισμένες ευκαιρίε που δεν έχουν από την οικογένειά του την δυνατότητα να συμμετάσχουν. Είναι σημαντικό και αυτοί να μπορούν να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν την Ευρώπη, να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε και τους ε, νέους ό,τι αφορά και τις εξωσχολικέ δραστηριότητε, τις εθελοντικέ ε, δραστηριότητε, τι αθλητικές δραστηριότητε. Δεν κάνει οι χώρες ε, στην παρούσα φάση που διοργανώνουν και συμμετέχουν σε κοινέ αθλητικές δραστηριότητε. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε και τις πιο μικρές δραστηριότητε. Εγώ προσωπικά, θα το είδατε και στην γνωμοδέτηση, σε δύο σημεία υπερέβησα αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, στον τον τομέα της ε, κατάρτισης. Και εγώ ακολούθησα τεχνική, τέτοια κατάρτιση και ξέρω πόσο σημαντικό είναι να δουλεύει κανείς. Κλείνει το μικρόφωνο Σομιλητρία. ich bin interveniert, weil ich... Ναι, συγγνώμη, ε, παρενέβησα γιατί έχετε ξεπεράσει το όριο της ομιλίας σας ε, και με Παρακαλώ να τηρείτε τα όρια. Μάλιστα. Να πω ότι στον τομέα του Interrail και του Discover EU θα πρέπει να σκεφτούμε και τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι σημαντικό σκέλος και αυτό. Ευχαριστώ πολύ και το λόγο τώρα έχει ο συνάδελφος Τζακσούκου. Στιμάτε, Un Μία πρόσφατη μελέτη θεωρεί ότι ο πολιτισμός είναι πρόκριμα για την ανάπτυξη της Ευρώπης και τη βελτίωση της ζωής και του τρόπου διαβίωσης. Εδώ και 15 χρόνια ένας δήμαρχος της Ρουμανίας, της Ρουμανίας μια ε, πόλης με 15.000 ε, κατοίκους το αποδεικνύει αυτό. Το 2000 έκλεισαν 2.000 ε, ανθρακοριχεία, η ανεργία ε, έφτασε το 70% αλλά στη συνέχεια έγινε, μετατράπηκε σε μία τουριστική ζώνη και οι Ιάπωνες ε, είναι αυτοί που κατακλείζουν αυτή την πόλη. Η πολιτιστική κληρονομιά, τα ταμεία συνοχής και η χρηματοδότηση των ε, ευρωπαϊκών σχεδίων, καθώς και τα δύο μνημεία της UNESCO που βρίσκεται σε αυτή την περιφέρεια, οδήγησαν σε αυτή την ανωδική πορεία αυτής της μικρής πόλης. Γι' αυτό εκτιμώ ιδιαίτερα το Erasmus Sin γιατί η Επιτροπή ζήτησε να αυξηθούν οι πόροι για το Discover EU και μόνο εάν εκτιμήσουμε τον πολιτισμό θα μπορέσουμε στο μέλλον να υποστηρίξουμε την Ευρώπη και να παραμείνουμε ενωμένοι μέσα στη διαφορετικότητά μας. Υπάρχουν χώρες που θέλουν αποκλειστικές αρμοδιότητες στον τομέα του πολιτισμού. Μας πείσατε όμως κατά την τελευταία θητεία ότι υπάρχουν μέσα και διακόπτει ο μιλητής. Ναι. Γνωρίζω ότι έχω υπερβεί το χρόνο μου, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και όπως είπατε στην αρχή της θητείας σας, τα μέσα αυτά αν δεν έχουν ε, νομοθετικό χαρακτήρα δεν θα αποτελέσουν εφαλτήριο. Έκλεισε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμού και διαπιστώσαμε ότι εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά δυστυχώς η λέξη πολιτισμός δεν αναφέρεται ούτε μία φορά. Τι θα αφήσουμε πίσω μας όταν ολοκληρωθεί η δική σας θητεία. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue. Έχει ο συνάδελφος Κρυμπόφσκι. Szanowny panie komisarzu, koleżanki, koledzy, w imieniu Grupy Europejskich Konserwatywnych. Επιτροπέ, κυρίε και κύριοι. Μιλώ εξ ονόματο τη ε, ομάδα των συντηρητικών μεταρρυθμιστών. Θα ήθελα να σα καλωσορίσω εδώ στην αίθουσά μα και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο στοιχεία. Στο θέμα του αθλητισμού και τη νεολαία. Θα Ήθελα να πω ότι αναφέρατε την νεολαία, κύριε Επίτροπε. Χάρηκα ιδιαίτερα για τον ενθουσιασμό για τις νέε τεχνολογίε, την εκπαίδευση και το γεγονός ότι είναι στο επίκεντρο οι νέοι σε ό,τι αφορά και το πρόγραμμα Erasmus Plus. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Η Βαρσοβία Δέλτα σας λέει κάτι. Νομίζω ότι δεν ξέρετε τα ονόματα αυτά. Πρόκειται για μια, ένα ποδοσφαιρικό, ποδοσφαιρική ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του κ. Λεβαντόφσκι και τώρα είναι πλέον παγκόσμια φύσμη, ξακουστό ε, ποδοσφαιριστή. Ε. Έχουμε πολλέ τέτοιε αθλητικέ λέσχε ε, εδώ και εκεί. Και πολλά παιδιά ξεκινούν την καριέρα του εκεί. Πολλέ φορέ σε μικρά χωριά, σε κομμοπόλεις σε τέτοιε αθλητικές λέσχες όπου έχει την ευκαιρία κανεί και να γνωρίσει άλλου ενέργου ανθρώπου, αλλά και να εμποτιστεί με αξίες. Εκεί προετοιμάζονται οι νέοι λοιπόν με έναν δομημένο τρόπο για τη μετέπειτα ζωή του. Είναι σημαντικό λοιπόν να το τονίσουμε αυτό. Είναι άλλωστε και η πολιτιστική, του κληρονομιά. Στο χωριό που είχα γεννηθεί είχαμε μια αθλητική λέσχη με 100 χρόνια παράδοση, έναν αιώνα. Θα ήθελα λοιπόν στην επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, αγαπητέ Επιτρόπε, να αφήσουμε κατά μέρο ένα ποσό του προπολογισμού για τους εκπαιδευτές, για τους προπονητές. Και όχι μόνο για τους νεαρούς ανθρώπους ε, που ακολουθούν μια τέτοια ε, εκπαίδευση, αλλά και για υποδομές. Έχουμε κάνει πολλά λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή στην Πολωνία. Πολλά είναι τα έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί, αλλά στην τελευταία δημοσιονομική προοπτική δεν δώσαμε τη δέουσα σημασία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρω ότι έχει τελειώσει ο χρόνο ομιλία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, και Πρόεδρο. Επόμενο ομιλητή είναι ο συνάδελφο, η κυρία Φόρτ, μάλλον. Ευχαριστώ. Η εκπαίδευση απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση. Να ξεκινάει από την γέννα, την άτυπη εκπαίδευση εντός οικογένειας μέχρι το χώρο της εργασίας. Πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολλά κοινωνικά αλλά και υλικά εμπόδια που εμποδίζουν την πρόσβαση όπως λέω στην ε, σχετική μου γνωμοδότηση άλλωστε. Αυτά περιλαμβάνουν την ψηφιακή πρόσβαση και τις ειδικέ ανάγκες ε, σε επίσημο και άτυπο επίπεδο. Επίσης ε, απαιτείται φροντίδα υψηλή ε, ποιότητα σε εγκαταστάσει ε, διδακτικέ ε, και φροντίδα και βέβαια μην ξεχνάμε τη μετάβαση στην αγορά εργασία. Και υπάρχουν και άλλε προκλήσει για τα κορίτσια και τι γυναίκε για να αναπτύξουν αυτοσεβασμό, αυτοπεποίθηση και όλα αυτά αποτελούν μια συνέχεια από τα πανεπιστήμια στην δουλειά και στην διαβίου κατάρτιση. Επίσης μπορούν να δοθούν προγράμματα σε αγοριά και κορίτσια μέσω και των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Θετικά πρότυπα, ο ρόλος των επιχειρήσεων και η ερμηνεία του τι θα έπρεπε να είναι οι γυναίκες. Όλα αυτά βεβαίως γίνονται μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης και της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Και πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην έρευνα και την ανάπτυξη και τα κράτη-μέλη να βλέπουν το τι λειτουργεί. Υπάρχουν κάποια εξαιρετικά παραδείγματα όσων γίνονται στις κοινότητές μας. Τέλος, πρέπει να γίνουν κάποιες σοβαρές συζητήσεις για το τι μπορεί να γίνει με τους υφιστάμενους πόρους και το τι απαιτεί περαιτέρω χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο πρώτος αντιπρόεδρος Μάκου Μάκουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, αγαπητέ Τίμπορ, να πω με άλλα λόγια αυτό το οποίο είπατε κι εσείς. Με τα δικά μου τα λόγια, το μέλλον της Ευρώπης είναι οι νέοι Ευρωπαίοι και το πώς αισθάνονται για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, στις δράσεις τους και τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Είδαμε και στις συζητήσεις ε, με τους νέους πως οι νέοι κάτω των 30 στηρίζουν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα μαζί τους και για αυτούς ε, θα πρέπει να προγραμματίσουμε το μέλλον της Ένωσης. Για το θέμα αυτό, καθώς εσείς έχετε ασχοληθεί και με το Erasmus Plus και το έχετε φέρει σε ένα νέο επίπεδο, νομίζω ότι αυτό είναι το βήμα προς τα εμπρός ε, πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το ότι πριν από δυόμιση χρόνια σε συνεργασία του γραφείου του δικού σας με το δικό μου όταν ήμουν πρόεδρος προετοιμάσαμε ένα έγγραφο 10 σελίδων για το πώς ε, θα οργανώσουμε την συνεργασία με την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ για το πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε. Και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Γιατί βεβαίως ε, οι αρμοδιότητές σας υλοποιούνται σε επίπεδο πόλεων και περιφερειών. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία για διαβίου κατάρτιση. Και αυτό σχετίζεται τώρα στενά με την ψηφιοποίηση και αυτό το οποίο λέμε STEM θετικές επιστήμες, ε, μαθηματικά και μηχανική. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, αλλά να βάλουμε και τις τέχνες μέσα και να το λέμε STEAM. Για να έχουμε έτσι μια διεπιστημονική προσέγγιση. Γνωρίζω πως έχετε το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο της ε, Βουδαπέστης ε, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και τα είχατε πει όταν ήρθατε στο δικό μας ε, το πανεπιστήμιο στο ΕΣΠΟ στη Φιλανδία όπου βρήκαμε πολλές κοινέ δραστηριότητες που μπορούμε να μοιραστούμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή λοιπόν είναι η Ευρώπη που μπορούμε να οικοδομήσουμε και να βασιστούμε σε αυτήν. Συνεργασία Τονίσαμε επίσης την έξυπνη εξειδίκευση στο Κοινό Κέντρο Έρευνας. Ανοίξαμε σήμερα την έκθεση εδώ στο Κοινοβούλιο για την συνάντηση με τους επιστήμονες ε, και αύριο βέβαια οι επιστήμονες θα συναντήσουν και τις περιφέρειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριο Καρατζουνή. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Επίτροπε που ήρθατε και αναπτύξατε τις σκέψεις σας. Τους τελευταίους έξι μήνες είχα μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, αλλά βεβαίως είναι και μια ευθύνη. Ο τομέας αυτός ε, του πολιτισμού ε, με απασχόλησε. Κοίταξα το τι έχουμε κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια. Εξοικειώθηκα με το έργο της Κομισιόν, του Κοινοβουλίου και βεβαίω του Συμβουλίου και της Αυστριακής Προεδρίας και πρόσεξα ότι υπήρξαν διαφορετικές ε, προσεγγίσεις διαφορετικά έγγραφα. Η Κομισιόν πέρσι τον Μάιο έκανε την πρότασή της, μετά στο δεύτερο μισό ασχολήθηκε με την ε, πολιτική κληρονομιά, υπήρχαν πολλές εκδηλώσεις ε, μετά υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών και είχαμε και ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψεων και βεβαίως και η Αυστριακή Προεδρία. Μέχρι τον Δεκέμβριο έτρεχαν να κάνουν ό,τι μπορούν. Οργάνωσαν μια εκδήλωση για τους Υπουργούς Πολιτισμού για να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση. Οπότε, όσον αφορά το τι έκανα εγώ. Κοίταξα τις λεπτομέρειες της πρότασης της Κομισιόν και βεβαίω πρέπει να δούμε το πλαίσιο 2021-2027 να αυξηθεί ο προπολογισμός του πολιτισμού γιατί τελικά αν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η ορμή που υπάρχει απαιτείται να αυξηθεί και η χρηματοδότηση δεν γίνεται αλλιώ. και χαίρομαι που η θα εγκρίνει το πρόγραμμα για την δημιουργική Ευρώπη και να το επεκτείνει. Θέλουμε να υπάρχει και συνέργεια. Βεβαίως σημειώνουμε ότι την σήμερα ημέρα ο πολιτισμός ε, είναι δραστηριότητα και των περιφερειών και των δήμων και τέλος θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα σημαντικά βήματα που νομίζω ότι πρέπει να γίνουν από τον Οκτώβριο πέρσι, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Έτος ε, Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ένα σημαντικό βήμα δηλαδή προς την σωστή κατεύθυνση. Και στην ε, σημερινή Ολομέλεια καταθέσαμε κάποιες ε, τροπολογίες και εγώ έχω καταθέσει μια τροπολογία όπου καλωσορίζω το ότι ανέφερε το γεγονός αυτό ο Επιτροπός Ναύρατσιτ στην Βιέννη. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει κυρία Σάριο που εκπροσωπεί τους ε, ασκούμενους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα, που μου δίνετε τη δυνατότητα να αποτανθώ σε εσά σήμερα. Αν κοιτάξετε γύρω σας, βλέπετε ότι οι γυναίκες αποτελούν μειοψηφία σε αυτό το πολιτικό σώμα και το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Οι γυναίκες σήμερα υποεκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα λήψης πολιτικών αποφάσεων συμπεριλαμβανόμενου και του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου. Εάν οι κυβερνήσεις δεν αντικατοπτρίζουν την κοινωνία μας, πώς μπορούν οι πολιτικές μας να ε, απασχοληθούν με τα ζητήματα των πολιτών. Γι' αυτό δημιουργήσαμε οργανώσαμε αυτή τη διάσκεψη για το ρόλο των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαμε 200 ε, συμμετέχοντες και 300 παρακολουθούσαν online για να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί η κοινωνία και το βλέπετε και στο δελτίο που σας διανύμαμε σήμερα. Έχουμε ένα διπλό μήνυμα μην ε, υποτιμάτε το ρόλο, το δικό σας ρόλο ως πολιτικοί εκπρόσωποι για την ισότητα των δύο φύλων. Μέτρα όπως ε, τομέας μεταφορών, η πρόληψη των, της εξιστικής διαφήμισης, η υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις γυναίκες μπορούν να προωθήσουν την ισότητα. Θα θέλαμε εσείς ε, ως ε, παλαιά μέλη να δείτε τι αντίκτυπος υπάρχει στις γυναίκες και θα θέλαμε πολύ περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν στον τοπικό προγραμματισμό έτσι ώστε ο τοπικός τομέας, ε, η τοπική αυτοδιοίκηση να αφορά και άντρες και γυναίκες. Επίσης, σε αυτή τη γνωμοδότηση ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εμείς ζητούμε από την Επιτροπή των Περιφερειών να ασχοληθεί με θέματα ισότητας των δύο φύλων. Για την επόμενη θητεία θα θέλαμε η Επιτροπή των Περιφερειών να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να διορίζουν περισσότερες γυναίκες και να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών εισηγητριών. Επίσης, στις ηγετικές θέσεις στο Προεδρείο να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες. Αυτά είναι βασικά βήματα έτσι ώστε η Ευρώπη να γίνει περισσότερο ίση που θα είναι καλύτερη Ευρώπη για όλους μας. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστώ. Έχουμε 15 ομιλητές που έχουν εγγραφεί. Κλείνει ο κατάλογος ομιλητών και θα ήθελα να τηρείτε το χρόνο σας, δηλαδή το ένα λεπτό. Το λόγο ο συνάδελφος ε, Γκαμάρα Ουές. Η συνάδελφος, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ και τον Επίτροπο για την εργασία του έτσι ώστε στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο να αυξηθούν τα προγράμματα για την εκπαίδευση. Υπάρχει βεβαίως αυτό το θέμα της συμμετοχής των νέων στα προγράμματα. Θα ήθελα το πρόγραμμα Erasmus Plus να είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να διευρυνθεί η συμμετοχή των ΑΜΕΑ σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί υπάρχει πολύ χαμηλή συμμετοχή των ΑΜΕΑ μέχρι τώρα. Και αυτό αφορά και τα προγράμματα κινητικότητας. Χρειάζεται προσαρμογή καθώς και περισσότερες εγγραφές στον προϋπολογισμό καθώς και οργάνωση για τη συμμετοχή τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Όμπερσνελ έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, ε, ως δήμαρχος της ΡΙΕΚΑ που το, του χρόνου θα είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του Πολιτισμού γνωρίζω τη σημασία του πολιτισμού ίσως ο πολιτισμός και η εκπαίδευση είναι τα μόνα μέσα κατά της ξενοφοβίας και του λαϊκισμού που είναι πανταχού παρόντες ο πολιτισμός είναι ο τομέας που θα πρέπει να συνεισφέρει για τη διάδοση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ελευθερίας. Εδώ μιλάω για την ελευθερία λόγου και ελευθερία πολιτισμών. Έχει μεγάλη σημασία η αύξηση χρηματοδότησης της δημιουργικής Ευρώπης αλλά και του έρασμου. Μην ξεχνάμε όμως και τα μία συνοχής γιατί πολλά από αυτά έχουν ενταχθεί στην πολιτιστική κληρονομιά. Η Άννα Μαγιάρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όλοι μας εδώ στην Ευρώπη έχουμε μία πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ο καθένας θα πρέπει να αναγνωρίσει τη δική του. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μάλλον διακόπτει Μιλήτρια και λέει ότι το θέμα των μειονοτήτων δεν είναι το ίδιο. Οι μειονότητες έχουν το δικό τους πολιτισμό και αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό για εμάς τους υπόλοιπους. Η πρωτοβουλία των πολιτών ζητά την προστασία των μειονοτήτων. Έχουμε ένα εκατομμύριο υπογράφοντες και μέχρι τώρα δεν έχουν επισυμβεί και πολλά από όσο γνωρίζω. Εάν θέλετε ε, να προωθηθεί, θα μπορέσετε να το κάνετε ουσιαστικά. Βάλτερ Φλέγκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα τέτοιο σημαντικό, και που μιλάμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, για την νεολαία και για την ε, εκπαίδευση στην Ευρώπη. Όταν ξεκινάμε ένα καινούριο πρόγραμμα, θα πρέπει πάντα να διερωτώμαστε ποιο είναι ο απότερο στόχο μα. Εδώ, ο απότερο στόχο μα και τη Ευρώπη και των κρατών μελών είναι να υπάρξει μια ενωμένη Ευρώπη, Ευρώπη μια ευφυή Ευρώπη, μια Ευρώπη με ευφυεί πολίτε. Και προ την κατεύθυνση λοιπόν αυτή θα πρέπει να εξετάσουμε πώ θα πετύχουμε του στόχου αυτού. Ω εκ τούτου, θα πρέπει να επιμείνουμε στην μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την επιστήμη, αλλά και κυρίως να επικεντρωθούμε στη ψηφιακή τεχνολογία και στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Για να προωθήσουμε την πολιτισμό των νέων. Αυτός πιστεύω ότι θα είναι ο δρόμος του μέλλοντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάρθει. Κύριε Επιτροπέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σκληρή δουλειά που έχετε κάνει και θα ήθελα να προσθέσουμε κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των τοπικών αρχών γιατί θα πρέπει να υπάρχουν πιο πολλές πλατφόρμες ανταλλαγής γνώσεων στις ε, πόλεις και στις περιφερειές υπάρχουν ε, μοντέλα βέλτιστων πρακτικών για παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, την προώθηση των σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τι τοπικέ κοινότητες. Επίτροπε, επίσης θα πρέπει να διδραματίσει πιο, πολύ, πιο μεγάλο ρόλο ο θεσμός των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, πολιτισμικών πρωτευουσών και για το Inter-Exit μεγαλύτερη προσοχή και καλωσορίζω την μεγαλύτερη επικέντρωση στο σκέλος του πολιτισμού που έχει μεγάλο ρόλο να παίξει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πολιτισμική ανάπτυξη των πόλεων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιτρόπο Ναύραψη σε όσοι αφορά τι δηλώσει που έκανε για την Ευρωπαϊκή Νεολαία. Να θίξω ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για την νεολαία. Ο πρόεδρος Γιούγκερ κάλεσε και αποκάλεσε μάλλον κάποτε την, ε, εθνική, την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων ως την καλύτερη ε, διαφήμιση από το 1976 λοιπόν ε, είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και πρόκειται λοιπόν ο πρόεδρος της ορχήστρας είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τη σειρά των, με την πάρδο του χρόνου έχει υποκτήσει μεγάλη φήμη και χρησιμοποιείται σε διάφορα εορταστικά περιστατικά, σε εορταστικές εκδηλώσεις και αποτελεί επίσης πολύ, πολύτιμη προϋπηρεσία για τους νέους μουσικούς από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή αυτή αρχίστρα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η τάση και στο μέλλον γιατί αποτελεί σημαντικό, σημαντική πρόθεση του μέλλοντος. Ευχαριστώ κύριε Μπόκα, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αν ε, ξεκινούσα εκ νέου θα ξεκινούσα με τον πολιτισμό. Αυτό είπε ο Ζαν Μονέ, ο θεμελιωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μεγάλη σημασία ο πολιτισμός για τη ταυτοποίηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού από βορρά προς νότο. Το πρόγραμμα πολιτιστικών πρωτευουσών στέφθηκε από επιτυχία. Είχαμε 300, 300 πόλεις οι οποίες έφτασαν στο, στην τελική ευθεία. Θα πρέπει το σχέδιο αυτό της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας και για τους νέους να οδηγήσει σε μια καλύτερη Creative Europe και να αρχίσει και ένα σχέδιο υπέρ των καλλιτεχνών καθώς και της ε, κινητοποίησης των νέων καλλιτεχνών. Ο Φρανσουά Κώστα. Ευχαριστώ. Προέρχομαι από μια περιφέρεια που αύξησε κατά 50% τον προϋπολογισμό υπέρ του πολιτισμού. Η Haute France είναι μια όμορη περιοχή και όλοι οι φορείς πολιτισμού λυπούνται γιατί το πρόγραμμα Interreg έχει μειωθεί δραστικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τον πολιτισμό και τους πολιτιστικούς ε, φορείς, ώστε να μπορούν να συνδράμουν και άλλες περιοχές, στην άλλη πλευρά δηλαδή των συνόρων. Μιλάμε για την εδαφική συνεργασία έτσι ώστε οι δρόντες στον τομέα του πολιτισμού να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα σύνορα και έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένας χώρος πολιτισμού και δημιουργίας. Ο κύριος Καριάνης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη βασίζεται μεταξύ άλλων στην εμπλοκή των πολιτών στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου ή τη περιφέρεια του. Για να είναι όμω δημιουργικοί και παραγωγικοί πολίτε, χρειάζονται πέραν τη επιμόρφωση και χώρου όπου θα καλλιεργήσουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την παιδεία πέστε μας πώς στηρίζετε τη δημιουργία υποδομών όπως βιβλιοθήκες, αίθουσες πολλαπλής χρήσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους οικαστικών τεχνών και εκθέσεων, συνεδριακά κέντρα και πώς θα μπορούσαν όλα, όλες αυτές οι υποδομές να συγχρηματοδοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει και η νεολαία μας πιο δημιουργική. Ευχαριστώ ο κύριος Φλίνκα. Δεν είναι εδώ όμως ο συνάδελφος Τζεριγού. Κύριε Επίτροπε, το Βερολίνο πέρσι έχει συμβάλει στο, στη διατήρηση της ευρωπαϊκού πολιτισμικού έτους. Αυτή η ευρωπαϊκή ταυτότητα και αυτή η κουλτούρα θα πρέπει να διατηρηθεί, θεωρούμε. Αλλά ο πολιτισμός θεωρούμε ότι δεν χρησιμοποιείται επαρκώς ως πόρος για λόγους χρησιμότητας. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν συζητάμε για τον πολιτισμό, γιατί προφανώς είναι σημαντική, σημαντικός ο πολιτισμός σε ό,τι αφορά και την διάσταση της δημιουργικότητας, όχι όμως πάντα με τη λειτουργικότητα ο πολιτισμό δεν θέλουμε να βελτιώσει μόνο την εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα χώρο όπου μπορεί να υπάρξει μια αντιπαράθεση σε ό,τι αφορά ε, πολλά ζητήματα που αφορούν όλες τις, όλα τα επίπεδα του κόσμου. Αυτό θα πρέπει να προωθηθεί μέσω δικτύων, μέσω θεάτρων. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί σημαντικό καθήκον το οποίο θα πρέπει να επιτελέσει το πρόγραμμα Creative Europe. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Σπυρίδων. Ε, αρχικά ήθελα επιγραμματικά να τονίσω την ανάγκη προώθησης δράσεων διαβίου μάθηση και επανακατάρτιση, ώστε οι περιφέρειέ μα αφενόμενα να παραμείνουν ανταγωνιστικέ στο διαρκώ μεταβαλλόμενο παραγωγικό μοντέλο που διαμορφώνεται εν ώψη τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αφετέρου δε να αντιμετωπίσουν τη βαθιά κοινωνική κρίση που πιθανά να επέλθει λόγω τη εξαφάνιση παραδοσιακών θέσεων εργασία. Στην υποχρέωσή μα για δραστική μείωση ανεργία, θα πρέπει οι νέοι να επανεκπαιδευτούν, να αποκτήσουν, να αποκτήσουν ικανότητες, έτσι ώστε η ανεργία η οποία απειλεί σε πολλά κράτη να διαρρήξει τον κοινωνικό ιστό να μειωθεί δραστικά. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι στη χώρα μου στην Ελλάδα οι νέοι έχουν ανεργία 40% όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 20%. Επίση, θα αναφερθώ σε πρωτοβουλίε πρέπει να αναλάβουμε για καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευση, πολιτισμού και αθλητισμού, επαναπροσδιορίζοντα του στόχου μα, ούτω ώστε να αγκαλιάσουμε όλε τι απειλούμενε κατηγορίε πολιτών σε μια Ευρώπη που ο πληθυσμό τη γερνά και δυστυχώ παράλληλα γεννήσει υποχωρούν. Στο σημείο αυτό όμως θέλω να εστιάσω το λόγο που ζήτησα να παρέμβω και να δώσω έμφαση στο πρόβλημα που μέχρι τώρα διαφαίνεται επειδή ό,τι αναφέρθηκα απαιτούνται... Ναι, και αναφέρομαι... Ξεπεράσατε το χρόνο ομιλία σα γι' αυτό λοιπόν θα περάσουμε στο επόμενο ομιλητή. Ο χρόνος ομιλίας σας ε, ολοκληρώθηκε. Σας παρακαλώ καθίστε. Και το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Ιώσεφ Πυρίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επιτροπέ. Ε, κύριε Επιτροπέ, κύριε Τίμπορ, ήδη ο συνάδελφος ε, έκανε το ερώτημα. Θα ήθελα και εγώ να θέσω το θέμα των μειονοτήτων. Πώς βλέπετε το θέμα ενός δεσμευτικού εγγράφου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Τέλος πάντων, έχει τεθεί το θέμα, οπότε να ρωτήσω εσείς πώς θα πάτε, τα παιδιά καλά, η υγεία, τι σκοπεύετε να κάνετε για το μέλλον και δεν ξέρω αν τα 5-7 χρόνια που ήσασταν επίτροπος άλλαξε κάπως η προοπτική που έχετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελευταίος ο συνάδελφος Λουκ Μπράντε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τις ε, προσπάθειές σας ε, να βελτιώσετε την ε, εκπαίδευση και τον πολιτισμό γιατί έχουν κέρια σημασία για την ενότητα της Ευρώπης. Θα ήθελα να υποβάλω μια πρόταση. Στην έκθεσή μου προς τον πρόεδρο Γιούνκερ πρότεινα οι Υπουργοί Πολιτισμού και Παιδείας να βάλουν ε, στην διδακτέα ύλη από τα δημοτικά είδη το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ξέρω βεβαίως πως η παιδεία δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αλλά θα μπορούσατε να αναλάβετε την ε, πρωτοβουλία, να προτείνετε στους υπουργού παιδείας να μπει στην διδακτέα ύλη, όπως σας είπα, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Στο παρελθόν η διαδικασία της Μπολόνιας και άλλες διαδικασίες ε, πήγαιναν προς αυτήν την κατεύθυνση, οπότε νομίζω ότι βεβαίως έχει βελτιωθεί το Εράσμους ε, που είναι μια πάρα πολύ καλή προσδοκία αλλά για να συνδεθούν και ιδιαίτερα οι νέοι μεταξύ τους ε, νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες ε, που λίγο πολύ τήρησαν το χρόνο ομιλίας. Τώρα ο Επίτροπος έχει να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση, να απαντήσει στους 20 ε, παρεμβαίνοντες και νομίζω θα το κάνει με μεγάλη ζωηράδα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος ε, και συγκεκριμένος όπου μπορώ και θα απαντήσω στην κάθε παρέμβαση χωριστά. για να μείνω και στο θέμα. Κύριε Μπορμπόη, με ρωτήσατε για το θέμα των ψηφιακών υποδομών ε, και τον ρόλο της ψηφιακής πρόσβασης ε, για να αποφευχθεί η φυγή των εγκεφάλων ε, και η ερήμωση των περιοχών της Υπέθρου στο ανατολικό τμήμα της Ένωσης. Γι' αυτό υιοθετήσαμε το σχέδιο ψηφιακής εκπαίδευσης πέρσι αρχές του προηγούμενου έτους ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης υποδομών ε, και περιεχομένου. Θα θέλαμε ακριβώς ε, να κινητοποιήσουμε περιφερειακά κονδύλια ή και κονδύλια της συνοχής έτσι ώστε οι περιοχές ε, να φτιάξουν αυτήν την ψηφιακή υποδομή και επιτόπου και στα σχολεία γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε το ότι σύμφωνα με τα δεδομένα μας μόλις 25% των ε, σχολείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Δηλαδή τα τρία τέταρτα δεν ε, έχουν, υστερούν στην ε, ψηφιακή επανάσταση. Επίσης και η εκπαίδευση των διδασκόντων. η κριτική σκέψη και τα λοιπά. Η διδασκαλία προγραμματισμού και λοιπόν ψηφιακών δεξιοτήτων. Όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο του συνασπισμού που έχουμε κάνει με τα κρατη για να τα εφαρμόσουμε. Κύρια Έλερ έθεσε το θέμα της νέας πτυχής του Εράσμους για να γίνει πιο κοινωνικά ευαίσθητο να έχει μια ευρύτερη ακριβώς ε, κοινωνική έκταση και ακριβώς θέλουμε να δώσουμε περισσότερα λεφτά στο Εράσμους σε άτομα που προέρχονται από οικογένειες με λιγότερες ευκαιρίες ε, για να λάβουν μέρος στα προγράμματα Erasmus γιατί κατά την άποψή μου είναι το πιο επιτυχές πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Π.χ. περιθωριοποιημένες ομάδες αλλά και πρόσφυγες ή ανάπηρους ε, το Εράσμος ε, μπορεί να τους στηρίξει πραγματικά και να τους ε, επανεντάξει στην κοινωνία. Ο κ. Σωσότσουκ με ρώτησε για την κληρονομιά μου. Δύσκολη ερώτηση. Να αναφερθώ στο εξής. Ο πολιτισμός και η εκπαίδευση έγινε ένα από τα κορυφαία ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα και τα κράτη-μέλη, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Γκέτεμποργκ, στην κοινωνική σύνοδο κορυφής, ε, ασχολήθηκαν ε, με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και συζήτησαν ε, την σημασία και τον ρόλο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ε, ταυτότητας. Γι' αυτό αναπτύξαμε τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο που είναι ένα σχέδιο χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να αναφέρω κάποια θέματα. Ξεκινήσαμε με την προσχολική εκπαίδευση καταρτήσαμε λεπτομερή σχέδια για τις ξένες γλώσσες, την αμοιβαία αναγνώριση πτυχίων, διπλωμάτων, απολυτηρίων. και το σχέδιο δράσης ε, της ψηφιακής εκπαίδευσης επίσης είναι μέρος αυτού του ευρύτερου σχεδίου. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που θα είναι τμήμα της ε, πολιτικής αυτής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό της Δημιουργικής Ευρώπης. Επίσης ε, αναφερθήκατε στο έτος πολιτιστικής κληρονομιάς ε, και στον αθλητισμό. Ξεκινήσαμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού και τα βραβεία συμπερίληψης που αφορούν ακριβώς αθλητικές ενώσεις και ΜΚΟ που κάνουν κάτι το ουσιαστικό σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συνοχή. Να αναφερθώ τώρα στον μαζικό αθλητισμό, αν μου επιτρέπετε, και τα βραβεία αυτά και την Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού. Συμφωνώ πλήρως πως ε, ο μαζικός αθλητισμό, η πολιτιστική κληρονομιά μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο τοπικό και στο περιφερειακό επίπεδο να ενισχύσουν ε, την ε, τοπική και περιφερειακή ταυτότητα. Ο ρόλος των προπονητών επίσης είναι πάρα πολύ πιο σημαντικός από όσο νομίζουμε Γι' αυτό ακριβώς ε, θα αυξηθεί και ο προϋπολογισμός ε, του Erasmus Plus στο κεφάλαιο του αθλητισμού ε, γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 7 χρόνια για να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για την κατάρτιση προπονητών, την ενημέρωση για τον κοινωνικό ρόλο των προπονητών, γιατί η άτυπη εκπαίδευση, ξέρετε, έχει το ρόλο της, όπως και η επίσημη εκπαίδευση. Ό,τι είναι οι δάσκαλοι είναι και οι προπονητές ε, στον τομέα τους. Η κυρία Φόρντ ε, επεσήμανε την σημασία της ψηφιακής πρόσβασης στην εκπαίδευση. Ναι, νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει έναν καλό τρόπο για να έρθουμε σε επαφή με τους νέους, με τα παιδιά, τους δασκάλους, σε απομακρυσμένες περιοχές, ε, να ψηφιοποιηθεί η διδασκαλία, να υπάρχουν νέες ευκαιρίες, συνεργασία. Μια μεγάλη ευκαιρία για το μέλλον. Γι' αυτό ακριβώς χρηματοδοτήσαμε αυτό το ηλεκτρονικό δίκτυο σχολείων ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη το οποίο φέρνει σε επαφή 500.000 δασκάλους σε διάφορα σχολεία και ελπίζω έτσι να επεκταθεί. Ο κ. Μάρκουλα τόνισε την σημασία της διαβίου κατάρτισης πράγματι. Και αυτό είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου. Κατά την άποψή μου, αυτό δεν αφορά μόνο τους ενήλικες ξεκινάει από την προσχολική εκπαίδευση και τους συνοδεύει σε όλη την ζωή. Πρέπει να ενισχυθεί λοιπόν ο ρόλος της διαβίου κατάρτισης και όλες οι πτυχές ε, του. Συμφωνώ επίση με τις άποψή σας ε, για την εκπαίδευση στις ε, θετικές επιστήμες. Θα θέλαμε να υπάρχει ακόμα εντονότερη συνεργασία των πανεπιστημίων στον τομέα αυτών. Ε, είναι ένας τομέας όπου μπορούμε νομίζω να επιτύχουμε κάποια πράγματα. Μιλάμε για τεχνολογίες εχμής και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αυτών των κλάδων. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και συγχαίρω την ε, Ριέκα μια καλή ευκαιρία για να δείξουμε την ομορφιά της πόλης που την ξέρουμε ήδη πολύ καλά και ταυτόχρονα να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους, ε, νέα μυαλά στην πόλη και να μεταμορφώσουμε την πόλη που έχει μια πλούσια βιομηχανική και εμπορική κληρονομιά αλλά και πολιτιστική κληρονομιά. Να μεταμορφωθεί λοιπόν σε έναν κόμβο ιδεών. Εμείς λοιπόν στηρίζουμε αυτές τις ε, πρωτοβουλίες αλλά δεν πρέπει να παραμελούμε τις πόλεις εκείνες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό αλλά δεν ε, κερδίζουν τελικά. Πέρσι στην Φλωρεντία ξεκίνησε το δίκτυο των ε, Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτεύουσων και υπήρχε και μια άλλη πρωτοβουλία για το δίκτυο των ε, παραλίγο πολιτιστικών πρωτεύουσων δηλαδή των πόλεων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό που έχουν πολύ καλές εμπειρίες μπορούν να μοιραστούν και ελπίζω φέτος να ξεκινήσει και αυτό το δίκτυο. Την έχουμε ένα εργαστήριο ανταλλαγής ε, ιδεών και εμπειριών. Αποκινούμε τις ε, πολιτιστικές πρωτεύουσες. Και βεβαίως Έχουμε του ε, στοχευμένου στόχου για ό,τι αφορά το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και έχουμε να κάνουμε και τις ασκήσεις ε, χαρτογράφησης ε, των συνεργειών μεταξύ των περιφερειακών ταμείων, των ταμείων συνοχής, ε, του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, του Εράσμους. Σε ό,τι αφορά την εταιρική σχέση GRC και εξετάζουμε λοιπόν ευκαιρίες για τα σημεία αυτά εστίασης και συνάντησης. Μία από τις δυσκολίες λοιπόν που αντιμετωπίζουμε είναι οι πολλές ε, διαφορετικέ νομικέ βάσεις για τα προγράμματα αυτά. Καταρχάς, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει μια εναρμονισμένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να συγκεντρώσουμε τα πλέον εκτίματα των προγραμμάτων αυτών και μετά να δούμε το σκέλος της ε, συνεργασίας. Ε, η κυρία Μαγιάρκη και τους Σουφιερή με ρώτησαν για τις προτεραιότητες και της επόμενης επιτροπής. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ μεγάλη και πολύ ε, ευαίσθητη η πολιτική συζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι προφανή πλατφόρμα για τέτοιε συζητήσει. Αποτελεί πολιτικό όργανο και δεν ξέρω πώ ε, θα διαμορφωθεί και πώ θα συμπεριφερθεί η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι στάση θα έχει έναντι της πρωτοβουλίας αυτής, αλλά θα αποτελέσει ορόσημο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όταν τα συλλογικά δικαιώματα, πολιτισμική αυτονομία, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και όλα αυτά τα οποία παραδοσιακά υπάγονται στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης πλέον περάσουν στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εμπειρία από πολιτικής άποψης. Θα είναι σίγουρα έντονη η συζήτηση. Κύριε Μακάρθη και κύριε Φλάγκο, με ρωτήσατε για μια πιο συνεκτική προσέγγιση στον πολιτισμό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο τέτοια δραστηριότητα. Μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία θέσεων απασχόληση, στην ανάπτυξη, στην περιφερειακή προώθηση των περιοχών, ακόμα και στην προώθηση του περιφερειακού τρόπου ζωή, στην ευμέρεια. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε όλε τι πτυχέ αυτέ και όλε τι συνέργειε. Για παράδειγμα, ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο μπορεί να αποτελέσει ε, πολύ σημαντικό φορέα στην ε, τοπική και περιφερειακή οικονομία. Αλλά επίση και κόμβο για την τοπική πολιτισμική ζωή. Θα πρέπει να αναπτύξουμε λοιπόν και να εκμεταλλευτούμε όλε τι συνέργειε, να αξιοποιήσουμε όλε τι ευκαιρίε που έχουμε στη διάθεσή μα για να προωθήσουμε τις ε, δραστηριότητες αυτές. Ο κ. Μακάρθη. Σε ό,τι αφορά το ρόλο της ε, πρωτοβουλίας, ε, είναι πολύ καλή του πολιτισμού. Είναι πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία. Το Κοινοβούλιο ξεκίνησε μια πολύ, ε, πολύ καλή πρωτοβουλία και έχουμε και τις περιφέρειες επιστήμης πλέον. Είναι πάρα πολύ σημαντική και καλή αυτή η πρωτοβουλία Κάνουμε και εμεί κάποιες δραστηριότητε όμως ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Το JRC για παράδειγμα, ταξινόμηση των δημιουργικών πόλεων και περιοχών, περιφερειών. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μιας πιο ευαίσθητη προσέγγιση στην ανάπτυξη πολιτισμού και στην ανάπτυξη δημιουργία ανάπτυξη. Έχουμε και στρατηγικέ εφίους εξειδίκευση. σε ό,τι αφορά τον κλάδο της περιφερειακής ανάπτυξης. Και εδώ θεωρώ ότι ο πολιτισμός είναι στο επίκεντρο αυτής της ευφυούς εξειδίκευσης και θεωρώ ότι στο μέλλον θα υπάρξει μεγαλύτερη εξειδίκευση στον τομέα αυτό και πιο πολλές εξελίξεις. Σύμφωνο απόλυτα μέσα σε, σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες να παραμείνει ζωντανό το σκέλος αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα υπάρξει πλέον επίσημη διαμόρφωση της χρηματοδότησης του σκέλου αυτού. Ο κ. Ντεκώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτό αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς ο πολιτισμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη και πιστεύω πραγματικά ακράδαντα ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα της οικονομικής ανάπτυξης με τη δημιουργία ε, βιομηχανίας ε, του σχετικού κλάδου, ε, με την προώθηση των κοινοτήτων γιατί όσο πιο συνεκτική είναι μια περιοχή, τόσο πιο ανταγωνιστική είναι. Γιατί η συνοχή δίνει αλληλεγγύη, αίσθημα αλληλεγγύης και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει εξαιρετική βάση για ανάπτυξη αλλά και για πλούσια πολιτισμική ζωή, δημιουργικότητα και ούτω καθεξής. σύμφωνα λοιπόν απόλυτα μαζί σας και υποστηρίζω τι φιλοδοξίες σα για μια κουλτούρα διασυνοριακής συνεργασίας. Θα πρέπει να ορίσουμε το πολιτισμικό πλαίσιο, αλλά ένα από τα όνειρά μα είναι να ανοίξουμε ευκαιρίε για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσε πολιτισμού, για διευρωπαϊκές τέτοιες περιοχές. Αυτό θα ήταν, θεωρώ, ένα πολύ καλό παράδειγμα για την ευρωπαϊκή διάσταση των, της, του πολιτισμού και για το πρόγραμμα κινητικότητας. Ο κ. Καραγιάννης έφτασε το ερώτημα του πολιτισμού και των υποδομών για τον αθλητισμό. Δυστυχώς η ανάπτυξη του υποδομών δεν ε, χρηματοδοτείται ιδιαίτερα από το πρόγραμμα Creative Europe είναι μέρος των περιφερειακών ταμείων και των ταμείων συνεχής. Ε, τώρα λοιπόν οργανώ... Ε, εργαζόμαστε για να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε τα όρια μεταξύ των περιφερειακών ταμείων και του Creative Europe. Δεν έχουμε ακόμα πετύχει μεγάλα αποτελέσματα. Ελπίζουμε στο μέλλον για κάτι καλύτερο. ευρωπαϊκές αξίες και η διδαχή αυτών σε ό,τι αφορά και την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση. Πέρσι, το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, το Συμβούλιο Εκπαίδευσης, Παιδείας και Εκπαίδευσης ενέκρινε όλες τις συστάσεις μας προς τα κράτη-μέλη για να εισαγάγουν την δασκαλία ευρωπαϊκών αξίων καθώς και την ευρωπαϊκή ιστορία στα εθνικά σχολικά προγράμματα. Ελπίζω ότι αυτό θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Euh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Όχι μόνο ακούσατε πολύ προσεκτικά, αλλά απαντήσατε σε όλους εξίσου προσεκτικά. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την άκρος αποδοτική συνεργασία. Πριν καλωσορίσω την Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, θα ήθελα να χαιρετήσω την αντιπροσωπεία των 35 δημάρχων από τις Μάρκε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα που βλέπουμε στο βάθος της αίθουσας. Έχουμε 10.000 υπογραφές για τη συμμαχία μας υπέρ της συνοχής, πάνω από 10.000 και αύριο ε, θα προσυπογράψετε την Σύμβαση Δημάρχων υπέρ του κλίματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δέσμευσή σας που αποτελεί αυτό παράδειγμα συνεργασίας. Θα βρείτε και ένα ερωτηματολόγιο ε, το οποίο, με το οποίο θα ξεκινήσουμε κατά την Ολομέλεια του Απριλίου μέσα στα πλαίσια της ε, συνεργασίας έτσι ώστε να έχουμε ένα φόρουμ συνεργασίας και συνοχής καθώς και ένταξης των μεταναστών θα μπορέσετε να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο και επιγραμμικά αλλά και εδώ και να το δώσετε στη γραμματεία ΣΥΒΕΞ που βρίσκεται εκτός της αίθουσας. Και τέλος, με βάση τον ε, εσωτερικό οργανισμό, η Άννα Μαγιάρ είναι γενική εισηγήτρια για να εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Σύνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το οποίο θα εγκρίνουμε αμέσως μετά την επόμενη συζήτηση. Chers collègues, je euh, θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Νταντσίλα, Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, που θα σας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας. Εδώ και ένα χρόνο ο Αντώνιο Κώστα εδώ από πλευράς Πορτογαλίας μας παρουσίασε τις προτεραιότητες της τότε Προεδρίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνδράμουμε από κοινού σε όλα τα επίπεδα για το μέλλον των Ευρωπαίων. Θα θέλαμε να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα μαζί μας. Από Τελεί τιμή για εμάς να σας καλωσορίσουμε για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες ε, της ε, Προεδρίας σας. Είναι η πρώτη σας Προεδρία μετά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για εμάς ε, διότι λαμβάνει η χώρα σε μια κρίσιμη περίοδο στα πλαίσια της έγκρισης του επόμενου ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και την ενδεχόμενη αποχώρηση ενός κράτους μέλους. Συμμετείχατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Ευρωβουλευτής πριν αναλάβετε τη διακυβέρνηση της ε, χώρας σας. Επίσης ήταν, ήσασταν δημοτική σύμβουλος, ξέρετε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και οικοδόμηση της Ευρώπης ε, με βάση τις δεκάδες χιλιάδες πόλεις που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται και για την τοπική δημοκρατία, δηλαδή την τρίτη διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στα πλαίσια μιας κοινή φιλοδοξίας. Μετά από ένα μήνα θα μας υποδεχτείτε στο Βουκουρέστι μέσα στα πλαίσια μιας εκδήλωσης που έχει ενταχθεί στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, βασιζόμαστε στη δέσμευσή σας όπως και εσείς στη δική μας. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ ως προς το μήνυμα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα συνέλθουν στο Σιμπίου το Μάιο για να καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι πόλεις και οι περιφέρειες χρειάζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τις πόλεις. Πρόκειται για ένα θέμα συνοχής, θεμελιωδών δικαιωμάτων, μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις πόλεις και τις περιφέρειες. Αυτό είναι το πρόσταγμα του Συμπίου. Μιλάμε για την συνοχή ως ορόσημο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς ημεριζόμαστε αυτή τη θέση. Δεν υπάρχει εφικτή ένωση χωρίς στεναρή συνοχή. Δεν μπορεί να υπάρχει συνοχή χωρίς τη συμμετοχή των πόλεων και των περιφερειών. Σας δίνω το λόγο, κυρία Πρωθυπουργέ. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, αγαπητά μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε Λάμπερτς, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, για την πρόσκληση να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Oui, ε, Euh, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε Λάμπερτς, καθώς ε, και τα μέλη της Επιτροπής ε, των Περιφερειών για την πρόσκληση να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της Ολομέλειάς σας ε, και ενός οργανισμού ο οποίος αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ τοπικών αρχών, περιφερειακών αρχών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η ατζέντα μας ε, σχετίζεται με πολλαπλές προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσω συνοχής, ενότητας και αλληλεγγύης. Γι' αυτό Το έμβλημά μας είναι η συνοχή, μία κοινή ευρωπαϊκή αξία αντικατοπτρίζοντας ε, τις θεμελιώδεις αρχές οικοδόμησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στα πλαίσια της συνοχής σε όλες τις, τις διαστάσεις πολιτική, συνοχή, οικονομική και εδαφική καθώς και κοινωνική συνοχή. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας με βάση τέσσερους, ε, τέσσερις πυλώνες. Ευρώπη της σύγκλησης, Ευρώπη της ασφάλειας, Ευρώπη ως παγκόσμιο παράγοντα και Ευρώπη των κοινών αξιών. Κυρίες και κύριοι, διανύουμε μια περίοδο όπου θα πρέπει να καταβάλουμε κοινέ προσπάθειες έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να δουν τα ευεργετήματα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος στην καθημερινή του ζωή. Αντιμετωπίζουμε την διαδικασία απόσυρσης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολιετές πλαίσιο, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και άλλες προκλήσεις όπως ε, η μετανάστευση, ασφάλεια και το μέλλον της Ευρώπης. Θα πρέπει να δείξουμε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη στήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών και να φτάσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους πολίτες. Υπό αυτή την έννοια, ο πρώτος πυλώνας του προγράμματος της Προεδρίας αφορά την Ευρώπη της Σύγκλησης. Υπ' αυτή την έννοια, λαμβάνοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οφείλουμε να έχουμε τους κατάλληλους πόρους για να υπάρχει η σωστή εξισορρόπηση μεταξύ πολιτικών ανάπτυξης και σύγκλησης, πολιτικής συνοχής, ΚΑΠ καθώς και πολιτικών που θα πρέπει να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις όπως η μετανάστευση, ασφάλεια και η συνοχή. Υπό αυτή την έννοια η πολιτική συνοχή αποτελεί μια προτεραιότητα στην ατζέντα μας. Χωρίς την πολιτική αυτή οι περιφερειακές ανισότητες θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες. Η πολιτική συνοχής δημιούργησε συνεργατικές σχέσεις μεταξύ θεσμών, περιφερειών και πόλεων της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται στη συνέχεια μια πολιτική συνοχής που να είναι στέναρη και αυτή να είναι η βασική μας στρατηγική επενδύσεων. Η πολιτική συνοχής εξελίχθηκε για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Υπό αυτή την έννοια η πολιτική αυτή χρειάζεται νέα συνοδευτικά μέτρα απλούστευσης και μεγαλύτερων αποδόσεων. Θα συνεχίσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις για την ε, πολιτική συνοχής ε, δυναμικά για να φτάσουμε στο συναφές νομοθετικό πακέτο έτσι οι πολιτικές αυτές θα αντικατοπτρίζουν την ε, καθημερινή ζωή των πολιτών, των πόλεων και των περιφερειών της Ευρώπης. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών για το στεναρό του ε, μήνυμα ήδη από την απαρχή των συζητήσεων για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο έτσι ώστε οι πόροι ε, συνοχής να προωθήσουν τη συνέχεια αυτής της πολιτικής η οποία αγκαλιάζει όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις. Η πρόθεση αυτής της ε, μακροπεριφερειακής πολιτικής μέσα στα πλαίσια της ε, στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια του Δούναβη αποτελεί την απαρχή νέων προκλήσεων για την ε, κατάρτιση μιας μακροπεριφερειακής πολιτικής. Παράλληλα, η Ρουμανία θα ήθελε να εφαρμόσει την Ατζέντα 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε εκπονήσει μια νέα στρατηγική και θα καταβάλουμε προσπάθειες για να καθορίσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές μιας νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί πρόκριμα και για την οικονομική συνοχή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά που να είναι λειτουργική μέσα στα πλαίσια θεμικά του ανταγωνισμού και ε, σε μία λειτουργία απόλυτης διαφάνειας και κινητικότητας. Μία από τις προτεραιότητες αφορά την ε, ε, παγιοποίηση της κινητικότητας των εργαζομένων. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις αναφάκελο καθώς και την αναθεώρηση των κανονισμών συντονισμού της κοινωνικής συνοχής καθώς και την σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Η διασφάλιση της ισότητας ε, και της ισότητας των φύλων και της ισότητας ε, ευκαιριών εργασίας αποτελεί ένα από τα ορόσημά μας. Υπ' αυτή την έννοια Υπάρχει η πρόταση οδηγίας ε, για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των γονέων και κηδεμόνων. Μας ενδιαφέρει άμεσα η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οικονομική ανάπτυξη, η προώθηση επενδύσεων σε μικρο και μακροοικονομικό επίπεδο. Υπ' αυτή την έννοια η Ρουμανική Προεδρία θα προωθήσει τις συζητήσεις σε σχέση με την εμβάθυνση της ΟΝΕ κατά επικοδομητικό τρόπο έτσι ώστε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της συνοχής και της ανθεκτικότητας της πολιτικής αυτής για να αντιμετωπίσουμε τους χρηματοοικονομικούς κλειδονισμούς. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε επίσης για μια Ευρώπη πιο ασφαλή. Πρόκειται για το δεύτερο πυλώνα. Η συλλογιστική της μετανάστευσης αποτελεί κοινό μας μέλημα και μας ενδιαφέρουν όλες οι διαστάσεις διαχείρισής της στα πλαίσια της ψηφιοποίησης και της υπεράσπισης των πολιτών στα πλαίσια της ε, εικονικής πραγματικότητας. Και αυτό αφορά κάθε ψηφιακό μέσο το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Γι' αυτό το όραμά μας αφορά μια Ευρώπη ως παγκόσμιο παράγοντα μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της ΕΕΔ για την ε, ασφάλεια της Ευρώπης. Θα προωθήσουμε όλες ε, τις ε, δυναμικές ασφάλειας μέσα στα πλαίσια και των εργασιών του ΝΑΤΟ. Χρειάζεται μία εμβαθυμένη συνεργασία και στα πλαίσια της προσανατολάς σχέσης γειτονίας μετά από τα πρώτα δέκα χρόνια από την εκκίνηση της ε, σχέσης, της εταιρικής σχέσης με τις ανατολικές χώρες και γι' αυτό θα προσδώσουμε μεγάλη σημασία και στα Δυτικά Βαλκάνη. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο τον τέταρτο πυλώνα των προτεραιοτήτων μας, δηλαδή την Ευρώπη των κοινών αξιών. Εν των ευρωεκλογών θα πρέπει να δώσουμε μία σωστή απάντηση έναντι των λαϊκιστών και των ευρωσκεπτικιστών, προωθώντας μία ένωση πιο δημοκρατική και πιο κοντά στους πολίτες της. Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός αποτελούν κλειδιά για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά την ατομική προοπτική του Ευρωπαίου πολίτη αλλά και υπό το πρίσμα επαγιοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο υπό αυτή την έννοια. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς μπορούν να προωθήσουν μια Ευρώπη πιο συνεκτική, πιο ενωμένη και πιο ασφαλή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εσείς όλοι έχετε να διαδραματίσετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είσαστε ο σύνδεσμος της ευρωπαϊκής πολιτικής και των περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων. Είμαι πεπισμένη ότι η 8η διάσκεψη κορυφής ε, των περιφερειών και των πόλεων που θα γίνει στο Βουκουρέστι το Μάρτιο θα στείλει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δέσμευσης για μια πιο δυνατή Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ε, περιμένουμε στο Βουκουρέστι το Μάρτιο και σας ευχαριστώ πολύ. Merci Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ για την ε, ξεκάθαρη αυτή και ακριβή παρουσίαση σε ό,τι αφορά την Προεδρία σας, σε ό,τι αφορά τους φιλόδοξους στόχους σας και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τα μέλη της Επιτροπής μας. Να σας υπενθυμίσω ότι καταρχάς θα ακούσουμε τις πέντε πολιτικές ομάδες και τους πρώτους αντιπρόεδρους και μετά θα δώσουμε το λόγο σε κάποια μέλη που ζήτησαν να παρεμβούν. Η κυρία Λουκαίδου. Merci, Monsieur le Président. Υπουργέ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εκ μέρους της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στη σημερινή Σύνοδο Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών. Αναφορικά με τα κοινωνικά και οικονομικά θέματα, η πρώτη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει η χώρα σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο εξάμεινο για τους πολίτες και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στο σύνολό του. Οι ευρωεκλογές του Μαΐου, οι οποίες θα καθορίσουν την πορεία της Ευρώπης για τα επόμενα πέντε χρόνια σε συνδυασμό με το επερχόμενο Brexit και τις δυσκολίες που συνεπάγονται αυτού δημιουργούν την ανάγκη μιας ρουμανικής προεδρίας η οποία θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου να αντιληφθεί ο κόσμος την κρισιμότητα και τη σημασία του να ψηφίσει στις συγκεκριμένες εκλογές. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση και έχουν κάνει σημαντική προσφορά τα τελευταία χρόνια στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία θα συνεχιστεί με τη διάσκεψη του Μαρτίου στο Βουκουρέστι. Δεύτερον, δράτω με της ευκαιρίας που είστε γυναίκα να δώσω έμφαση και να σας συγχαρώ για την εισαγωγή στις προτεραιότητες της Προεδρίας τη σημασία της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άντρες καθώς και της σημασίας της μείωσης του χάσματος των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών θέματα που είναι απαράδεκτο να μην έχουν επιληθεί εν έτη 2019. Τρίτον, ένας άλλος σημαντικός τομέας που απασχολεί πολλούς πολίτες είναι η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τα προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτές από την πολιτική εμπορίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κ. Τραμπ οι δύο πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εμπορικές συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ πάνω στην κατάργηση των δασμών για βιομηχανικά προϊόντα και την άρση των μη δασμολογικών φραγμών είναι μια σωστή κίνηση που θα πρέπει να υποστηριχθεί από εσάς. Χαιρετίζω ότι ο ουσιαστικός ρόλος της πολιτικής συνοχής είναι το κεντρικό σύνθημα της Προεδρίας σας. Θα ήθελα ωστόσο να σημειώσω ότι το ΕΛΚ πιστεύει ότι είναι σημαντικό προς όφελος των πολιτών μας να εγκαταληφθεί η συγκεντρωτική πολιτική και να μεταβιβαστούν εξουσίες στις περιφέρειες και τις πόλεις για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες αναφορικά με την ασφάλεια των συνόρων της Ένωσης και τις σχέσεις καλής γειτονίας πρώτον Κύπρια ούσα δεν θα μπορούσα να παραλείψω να πω ότι βασιζόμαστε στη στήριξη της Προεδρίας σας για την προσπάθεια που λαμβάνει η χώρα αυτή την περίοδο ώστε να αναζωογονηθούν οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού. Είναι αναγκαία η εξέβρεση μιας δίκαιης λύσης στη βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας βασισμένη στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Δεύτερον, θα πρέπει αυτή την περίοδο να κάνουμε βήματα μπροστά σχετικά με το μεταναστευτικό, το οποίο θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Είναι σημαντικό να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαίων και ενδυνάμωση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Οι υποχρεώσεις μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να καταλήγουν σε δίκαιη κατανομή βαρών. Ευελπιστώ πως η Ρουμανική Προεδρία θα δώσει έμφαση στην έβρεση συμφωνίας αναφορικά με την πολύ καλή πρόταση για την ενδυνάμωση του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτιοφυλακής με προσωπικό 10.000 ατόμων. Τέλος, η παρουσία σας εδώ σήμερα αποδεικνύει την προθυμία σας να λάβετε υπόψη την φωνή των περιφερειών και των πόλεων και σε αυτό το πλαίσιο θα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στα καθήκοντά σας αναφορικά με την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και το λόγο τώρα έχει η συνάδελφος Ιζαμπέλ Μπουλινό. Κυρία Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και ε, αισθήκαμε την ε, ένταση μεταξύ των χωρών μας σε ό,τι αφορά και την πολιτική συνοχή. Βάλατε λοιπόν στην κορυφή της προτεραιότητας ε, το προτεραιότητα στα θέματα αυτά και αναλάβατε τα ενία της Προεδρίας μια ευαίσθητα στιγμή εν ώψη των κλειπανισμών του Brexit, ε, την στιγμή που πλησιάζουν οι ευρωεκλογέ, ε, τη στιγμή που θέτουμε τις πολιτικές για την περίοδο μετά το 2020. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι και έτσι αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μια ευκαιρία να θέσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στο ύψος των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών, 1,3% του ΑΕΠ σε ό,τι αφορά και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2020-2027. Θεωρούμε ότι η συμφωνία δεν θα είναι ικανοποιητική να περιλαμβάνει καινούριου ε, ίδιου πόρου. Δυστυχώ, από ό,τι ακούμε, δεν προχωράει όμω το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όλε όμω οι μελέτε, όλε οι έρευνε που έχουν γίνει αποδεικνύουν ότι θα ήταν πολύ καλύτερο ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Μα λείπει λοιπόν αυτή η μακροπρόθεσμη διάσταση για να ε, πραγματοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε τα εμπόδια της Ευρώπης και να θέσουμε σε εφαρμογή ένα κοινό όραμα για το κοινό μας μέλλον. Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε πόσο σημαντικό είναι λοιπόν να πετύχουμε μια συμφωνία για το πολιτές οικονομικό πλαίσιο για να αγγιηθούμε τη συνέχιση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προκειμένου οι περιοχές και οι περιφέρειες να συνεχίσουν να επιδιώκουν χωρίς διακοπή την ε, πρόθεση των στόχων μας. Η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τη βασική πολιτική επενδύσεων για τις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης και την καλύτερη έκφραση αν θέλετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί υποστηρίζει όλες τις ε, περιοχές ε, αστικές και υπεθρό. Και επίσης η Ευρώπη ή της αλληλεγγύης που βάζει τον Ευρωπαίο πολίτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι αυτό που επιθυμούμε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο που η χρηματοδότηση των νέων προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ει βάρον των υφιστάμενων ε, προτεραιοτήτων όπω η πολιτική συνοχή και η κοινή γεωργική πολιτική. Θέλουμε λοιπόν να επιμείνει η Ρουμανική Προεδρία σε ό,τι αφορά τι πιο ορατέ πολιτικέ για του πολίτε, για να μην υπάρχει αρνητικό αρνητικός στην ανάπτυξη. Τη στιγμή μάλιστα που οι εθνικοί προπολογισμοί δεν έχουν ακόμα συνέλθει από το σοκ της οικονομικής κρίσης. Θα θέλαμε να πούμε λοιπόν ότι να υπάρξει ο κώδικας διοντολογίας ο οποίος να ενταχθεί στην ε, διευθέτηση και στη ρύθμιση των ε, περιφερειακών ταμείων. Θα πρέπει όλα αυτά να μπουν λοιπόν σε μια ε, νέα ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη που επιθυμούμε σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό για μια καλύτερη περιφερειακή ισότητα, λιγότερες ανισότητες κοινωνικές, προοπτικέ για του νέου. Εδώ ψάχνουμε και αναζητούμε την Ευρώπη για μια φορά ακόμη, λοιπόν, θα θέλαμε να σα ευχαριστήσουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, να ευχαριστήσουμε τη Ρουμανική Προεδρία για το γεγονό ότι έβαλε την πολιτική συνοχή στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων σα και σα ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σα ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει την συνάδελφο Γιάννα Κράμπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να σας καλωσορίσω και εξ ονόματος των φιλελευθέρων αναφερθήκατε στα Δυτικά Βαλκάνια σήμερα ήδη και θα ήθελα λοιπόν να σας υποδείξω το θέμα των διαπραγματεύσεων με την Βορεια Μακεδονία. Όπως ξέρετε πλέον η χώρα αυτή ζήτησε ε, προσχώρηση στο ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ λοιπόν που τοποθετηθήκατε με σαφήνεια αυτό το καλωσορίζουμε. Και καλωσορίσαμε και αυτή την πρόθεση. Επανελειμμένως. Μετά από συναντήσεις με εκπροσώπους στη Βόρεια Μακεδονία, λοιπόν, προκύπτει με σαφήνεια ότι είναι σαφής οι τοποθετήσεις ε, για τα βασικά θεμελιώδη ζητήματα. Οι τοπικές αρχές προφανώς συζητούν τα θέματα αυτά. Όλοι οι φορείς αντιλαμβάνονται ότι η επίλυση του ζητήματος αυτού θα έχει ιδιαίτερη επίπτωση στην ευημερία της περιφέρειας. Και αυτό είναι και ένα σημαντικό βήμα πριν την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίλυση λοιπόν των βασικών ζητημάτων θα εξασφαλίσει την επίλυση των ε, τρεβών εντός της μακεδονικής ε, κοινότητας. Μιλώντας με δημάρχους από την ε, Βόρεια Μακεδονία, παρατηρήσα ότι ζητούν μεταρρυθμίσεις. Αντιλαμβάνονται ότι πολλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν εκ παραλλήλου. Τα τελευταία πέντε χρόνια είμαι μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών και αντιλαμβάνομαι και σημειώνω μεγάλο σκεπτικισμό σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, μακρές συζητήσεις για το θέμα της ονομασίας. Υπάρχουν κάποιες ε, αμφιβολίες που εκφράστηκαν για το κατά πόσο θέλει να προσχωρήσει η Μακεδονία, η Βόρεια Μακεδονία. Αλλά ο κ. Ζάιρ έχει εκφράσει την επιθυμία να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Καλό λοιπόν όλους τους εκπροσώπους ε, των ευρωπαϊκών κρατών μελών και εσάς ε, όλος ιδιαίτερος ω Πρωθυπουργό τη Ρουμανία. Ε, και ασκούσε την Προεδρία να ανοίξουμε την πόρτα για τη διαδικασία αυτή γιατί αν δεν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία θα υπάρξουν περαιτέρω εντάσεις ε. και αυτό θα δώσει μεγαλύτερη επιρροή σε ανατελικές ε, περιοχές στο κομμάτι αυτό των Μαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο θέμα το θέμα των ε, μη δημοκρατικών ηγετών. Οι πιο πολλοί άνθρωποι ζουν σε αστικά κέντρα. Οι δήμαρχοι λίγο πολύ προστατεύουν τα δημοκρατικά δικαιώματα και εμείς ε, προστατεύουμε τη δημοκρατία στις περιφερειές μας. Έχουμε λάβει σημαντικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα αντιδημοκρατικά κινήματα στην περιφερειά μας και δεν έχω άλλο χρόνο να μιλήσω. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την Προεδρία να μας πει πώς η Προεδρία μπορεί να προωθήσει τέτοιες δράσεις σε τοπικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο. Θα ήθελα επίσης να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Σε αυτές τις ε, ταραχώδεις εποχές που περνάει η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ και προσβλέπουμε στα αποτελέσματα που θα πετύχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο τώρα το λόγο έχει ο κ. Γιούγκμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί Πρωθυπουργέ. Εξ ονόματος της ομάδας του ECR θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στην Ολομέλειά μας και να ζητήσω από την Προεδρία σας να βοηθήσει ε, στην επίτευξη που έχει, των στόχων που έχει θέσει η Ρουμανική Προεδρία. Θα ήθελα να εξηγήσω τι εννοώ. σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση τη αγορά, Προσπαθούμε αυτό να ωφελήσει όσο και πολλοί πολίτε γίνεται. Να μην ξεχάσουμε όμω το εξή, να μην πέσουμε στην παγίδα τη δημιουργία ενό κεντρικά διαμορφωμένου συστήματος αναδιανομής. Τέτοια συστήματα έχουν δοκιμαστεί στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη από τα καμονιστικά καθεστώτα και πέρα από τα τραύματα τα οποία δημιούργησαν, απέτυχαν επίση οι τοπικές αρχές γνωρίζουν καλύτερα τις ε, περιοχές τους. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες για επενδύσεις πιο πολύ από ότι τα άλλα επίπεδα διακυβέρνησης και η λήψη αποφάσεων στο τοπικό επίπεδο επίσης βελτιώνει τη δημοκρατικό χαρακτήρα της ε, των περιοχών. Είμαστε επίσης εταίροι στη χρήση των ταμείων. Δεν είμαστε εμπλεκόμενα μέρη. Σε αυτό περιλαμβάνεται και στα διευκρινιστικά κομμάτια του Ταμείου Συνοχής, για παράδειγμα, που είναι στο 1 τρίτο της, ε, των ευρωπαϊκών δαπανών. Το, οι ευρωπαϊκές εξάμεινες, το, ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό εξάμεινο όμως εξακολουθεί να είναι μια δικασία από πάνω προς τα κάτω. Δεν αντιμετωπίζει τις τοπικές αρχές ως εταίρους. Και υπάρχει και σχετική γνωμοδότηση τη Επιτροπή μα για το θέμα αυτό. Και έχω την τιμή να είμαι εισηγητή για το θέμα αυτό και προσβλέπω στη γνωμοδότηση τη ε, Επιτροπή μα για το θέμα αυτό όταν ολοκληρωθεί η γνωμοδότηση τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Κυρία Πρωθυπουργέ, η ομάδα μου ζητά λοιπόν ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση. Ελπίζουμε με τη νέα φετιά να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την ε, προσπάθειά μας για την Ευρώπη, Ευρώπη των πολλών, όχι των λίγων. Και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας για την επιτευχή του στόχου αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα το λόγο έχει ο κ. Μάρκο Μάκουλα. Κυρία Πρωθυπουργέ, να τονίσω εδώ τα βασικά μηνύματα που άκουσα στην ε, δήλωσή σας και διαβάσαμε στα της ε, Προεδρίας σας. Βλέποντας τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα γύρω μας, οι βασικές προκλήσεις είναι οι ίδιες. Αφενός είναι να παραμείνουν οι πολίτες στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μέσω περιεκτικών μεθόδων διακυβέρνησης κάτι το οποίο αφορά ιδίως τους δημάρχους και λοιπούς ερετούς ε, σε τοπικό επίπεδο και από την άλλη εστιάζουμε στην εφαρμογή των ε, στόχων ε, βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ. Για να επανέλθει η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες τονίζουν την ε, ανάγκη τοπικών δραστηριοτήτων. Αυτό είναι σημαντικό για όλους μας και για εμένα και καθώς Φιλανδία θα αναλάβει στην συνέχεια την Προεδρία αναμένω και εγώ την συνεργασία που θα έχουμε και στην ε, Φινανδία και ως ε, Περιφερειάρχης ε, Ελσίνκη και πιθανότατα θα σας ξαναδώ και θα συνεργαστώ και με τους υπουργούς σας. Εμείς, η Επιτροπή των Περιφερειών, συνιστούμε την προώθηση της καινοτομίας γενικώ και της κοινωνικής καινοτομίας για να αυξηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και η συνοχή στην Ευρώπη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο προτεραιότητες σας. Πρώτα, την μακροπεριφερειακή στρατηγική και την εμπειρία των όσων έχουμε κάνει στην περιοχή της Βαλτικής για να βοηθηθεί και η περιφέρεια, η μακροπεριφέρεια του Δούναβη και της ε, Μαύρης Θάλασσας. Μικρές εταιρείες, έξυπνη εξειδίκευση κτλ. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο ήδη έχετε τονίσει, τα Δυτικά Βαλκάνια, πώς μπορεί να σημειωθεί πρόοδος ε, εκεί, είναι σημαντικό για εμάς από τον Βορρά, τον Νότο ή την ε, Ανατολή, την Δύση. Είναι σημαντικό για όλους μας λοιπόν. Γι' αυτό ακριβώς ε, όλα αυτά και υπό το φως ε, της εφαρμογής της Συμφωνίας ε, των Πρεσπών. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε την Ευρώπη για όλους. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο Εμίλ Τζραγκίτσι. Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα να αποτανθώ ενώπιον σας και να σας χαιρετήσω από πλευράς των φιλελευθέρων ως πρωθυπουργό της χώρας μου και μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τας και της εντολής σας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε να προωθήσουμε συγκεκριμένα νομοθετήματα, διότι το 75% των ε, νομοθετικών πράξεων εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο που βρίσκεται πολύ κοντά στο πολίτη. Άρα μετά από σχεδόν έναν αιώνα προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα μελήματα των πολιτών, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγροτικές περιοχές προαπαιτούν προγράμματα συνοχής διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις υποδομών και τρόπου ζωής μεταξύ αγροτικών περιοχών και μεγάλων άστεων. Ξεκινώντας από αυτή την ιστορική διάσταση και δυνάμει του άρθρου 8 της συνθήκης της ε, Λισαβόνας για να υπάρχουν σχέσεις καλής, ε, ε, καλής γειτονίας θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσονται οι σχέσεις μας και με τη δημοκρατία της Μολδαβίας με προγράμματα ειδικής συνεργασίας έτσι ώστε οι Ρουμάνοι πολίτες αλλά και οι Μολδαβοί να μπορέσουν να προωθήσουν μια συνεργασία γιατί μην ξεχνάμε ότι το ίμιση του το ίμιση του πληθυσμού της Μολδαβίας έχει ρουμανική υπηκότητα αλλά και βουλγαρική, ιταλική και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε τις σχέσεις ε, καλής γειτονίας και των προτιμησιακών σχέσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Λάμπερτς γιατί προώθησε τις ε, τοπικές ε, ε, συνεταιριστικές σχέσεις και σας περιμένω μαζί με τον κύριο Μάρκουλα στο Βουκουρέστι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρωθυπουργέ για το δυναμικό σας λόγο. Η Μαριάννα Γκασού έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη μας χαρά να χαιρετήσουμε την παρουσία σας στα πλαίσια των θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων όπου επιθυμούμε να προωθήσουμε μια Ενωμένη Ευρώπη. Ξέρουμε ότι για τη Ρουμανία αυτό αποτελεί και πρόκληση αλλά και ευκαιρία. Γιατί πρόκληση, γιατί το εργατικό δυναμικό αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Είναι μια ευκαιρία, κυρία Πρωθυπουργέ, που δεν μπορούμε να τη χάσουμε. Η παρουσία στο Βουκουρέστι για διασκέψεις κορυφής, σεμινάρια και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστούμε γιατί η 8η διάσκεψη θα γίνει στο Βουκουρέστι και θα συμμετάσχουν 500 τοπικές αρχές αλλά και 100 ε, οργανώσεις νέων. Ολόκληρη η Ρουμανία, το Κλούσνα Πόκα, το Σιμπίου, ε, η Μπάια Μάρε, το Βουκουρέστι, όλες αυτές τις πόλεις ε, μπορείτε να τις επισκεφτείτε. Να δείτε τις ομορφιές της πατρίδας μου και τον πολιτισμό και τις παραδόσεις των Ρουμάνων. Παράλληλα μπορούμε να πούμε ότι θα προωθήσουμε τις οικονομικές, ε, το οικονομικό μέλλον των νέων. Κυρία Πρωθυπουργέ, τα προβλήματα και οι προτεραιότητες είναι πολλές. Εσείς ως ε, Ρουμάνα πολίτης θα μας ε, εκπροσωπήσετε σωστά. Θα ήθελα αυτό το εξάμεινο να προωθήσετε και το θέμα των θεωρήσεων ε, για το χώρο του Σέγγεν. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μας να προσχωρήσουμε στο χώρο Σέγγεν και ευχαριστώ πολύ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών. Σας περιμένουμε με μεγάλη αγάπη για να δείτε τις αξίες και τις παραδόσεις του ρουμανικού λαού. Ελπίζω λοιπόν να συμμετάσχετε σε αυτή τη διάσκεψη όπου θα συμμετέχει και η Δημοκρατία της Μολδαβίας και θα αποτανθείτε και στις τοπικές αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας όπου εμείς θα πρέπει να συνδράμουμε για να προσχωρήσει η Μολδαβία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε δίπλα σας ενότητα από τη διαφορετικότητα αλλά μέσω ένωσης έρχεται και η δύναμη σας ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ το λόγο έχει τώρα κύριος Καμίνης Είναι εδώ ο κύριο Καμίνη, ε, Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε. La parole est maintenant... Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Γκίντεβολφ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερος ε, θετικό και ευχαριστώ και την Ρουμανική Προεδρία που αναλαμβάνει καθήκοντα για να διατηρήσει την συνοχή της Ευρώπης. Θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο για να έχουμε κάποια φιλοδοξία να εγκριθεί και φέτος. Σας παρακαλώ λοιπόν να προσπαθήσετε να επιτύχετε κάποια πρόοδο και επιπλέον ε, να διατηρήσουμε τις αρχές μας, ε, την αρχή του κράτους δικαίου, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της διαφθοράς, πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Η παράκλησή μου είναι να λάβετε υπόψη τις αντιρρήσεις ε, της ε, Κομισιόν ε, και της Επιτροπής της Βενετίας για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που κάνετε στη χώρα σας. Δεν είναι ανάμειξη στα εσωτερικά μιας χώρας. Πρόκειται για εμπιστοσύνη, γιατί χωρίς αυτήν δεν υπάρχει συνοχή της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Τώρα τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Χλίνκα. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να εξετάζουμε και να κάνουμε διαπραγματεύσει για το θέμα αυτό τη πολιτική συνοχή ε, μετά το 2020. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε το εξή, πώ η Ρουμανική Προεδρία σκοπεύει να ενθαρρύνει την όλη διαδικασία αυτή, να δώσει κίνητρα και η συνεργασία με την Επιτροπή Κορίνα Κρέτου πώς θα δημορφωθεί και με τη σχετική γενική διεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μακάρθουρ, έχετε λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτον, οι πηγές ε, χρηματοδότησης ε, των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να κατευθύνονται στις περιφερειές και πρέπει να στείλουμε το σχετικό μήνυμα στα κράτη-μέλη. Πρέπει να κοιτάμε προς το μέλλον, διδασκόμενοι από το παρελθόν, να δούμε την καινοτομία, τις νέες μεθόδους επενδύσεων, να επενδύσουμε στην οικονομική ανάπτυξη, ακόμα και σε μικρές περιφερειές. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ένα σχέδιο δράσης για τις ε, πόλεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολλά καλά παραδείγματα. Αλλά πρέπει να αναπτυχθούν ε, περαιτέρω στις πόλεις. Με την Συμμαχία για την Συνοχή, Επιτροπή των Περιφερειών μας έχει δείξει πώς μπορούμε ακριβώς να πούμε μια... να αναπτύξουμε ένα φύγημα για τα διαφορετικά ταμεία. Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν τα μηνύματα τα οποία θέλω να σας επευθύνουν ε, τα μέλη της Επιτροπής μας και σας δίνω το λόγο με χαρά για να απαντήσετε στα σχόλια αυτά, κυρία Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα λεχθέντα, τα προβλήματα τα οποία αναγνωρίσατε, καθώς και τις προσδοκίες που έχετε από τη Ρουμανική Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Για την κυρία Λουκαίδου από το ΕΛΚ, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και για τις εκτιμήσεις σας. Έχετε δίκιο. Οι ευρωεκλογέ του Μαΐου θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο για το μέλλον της Ευρώπης. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται συνοχή μεταξύ θεσμικών οργάνων και όλων εκείνων που μπορούν να προωθήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες ε, αποτελούν προαπαιτούμενο. Η παρουσία μου και εδώ και στην ΕΟΚΕ δείχνει ότι έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους, σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν την Ευρωπαϊκή Οδό. Για μας δεν έχει σημασία ποιο πολιτικό κόμμα θα κερδίσει αλλά θα πρέπει να κερδίσει η Ευρώπη κατά των ευρωσκεπτικιστών και των αντιευρωπαϊκών δυνάμεων. Αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου εν ώψη των ευρωεκλογών. Η ισότητα των δύο φύλων στη συνέχεια. Αυτό το θέμα ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να περάσουμε από τις ε, δηλώσεις από το δηλωτικό λόγο στα συγκεκριμένα μέτρα. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό και στις 31 ε, Μαρτίου θα οργανώσουμε μία διάσκεψη για την ισότητα των δύο φύλων και ελπίζουμε να παρευρεθείτε και εσείς στη διάσκεψη αυτή. Τώρα, ο ρόλος της συνοχής ε, έχει μεγάλη σημασία για τη Ρουμανική Προεδρία. Γιατί δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι διχασμένη, ότι υπάρχουν πολλές αποκλίσεις και πιστεύω ότι η συνοχή θα πρέπει να μας απασχολήσει, όπως είπα και στην αρχή. Μας ενδιαφέρει η πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνιστόσα. Γι' αυτό η συνοχή είναι η ατμομηχανή της Ουμανικής Προεδρίας. Ε, κυρία Μπουτίν, ελπίζω να μην κάνω λάθος τα ονόματα, να μην τα προφέρω λάθος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, προκλήσεις τις οποίες δεν είχαμε μέχρι τούδε και που θα πρέπει να απαντηθούν από κοινού. Προκλήσεις που σχετίζονται με το Brexit αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit. Θα πρέπει να οριοθετήσουμε τα πλαίσια λειτουργίας μας. Στις 9 Μαΐου στο Συμπίου θα προσπαθήσουμε να δούμε και το θέμα των προκλήσεων του ΠΔΠ εν ώψη και των ευρωεκλογών και τις νέες προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την χορήγηση ασύλου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις παραδοσιακές μας πολιτικές επίσης, δηλαδή την ΚΑΠ και την πολιτική συνοχής. Το ΠΔΠ εκπροσωπεί ένα από τα βασικά μελήματα της Ρουμανικής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις εδώ ξεπερνούν τις ε, συνήθεις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα στα πλαίσια της εκπεριτροπής προεδρίας είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις συζητήσεις. Η Ρουμανία πρότεινε να προωθήσουμε τις ε, συζητήσεις με βάση τις διαπραγματεύσεις για να φτάσουμε σε ρεαλιστικές επιλογές έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια συνένεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά το φθινόπωρο του 19. Ως προς τις πολιτικές αλληλεγγύης θα πρέπει να μας διέπουν, να διέπουν τις εργασίες μας. Γι' αυτό μίλησα και για την κοινωνική αλληλεγγύη που θα πρέπει να προωθηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η υποστήριξη των περιφερειών και πόλεων. Συζήτησα το θέμα με τον πρόεδρό σας έτσι ώστε να βρούμε τα καλύτερα, να φτάσουμε στα καλύτερα αποτελέσματα με βάση την απτή μας πραγματικότητα. κυρία Γκράβνεκ. Τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν μία προτεραιότητα για την Προεδρία μας μαζί με την Ανατολική Εταιρική Σχέση ως προς τις διαπραγματεύσεις για τη Βόρεια Μακεδονία αποτελούν προτεραιότητα για εμάς και γι' αυτό αυτό χαιρετίζουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών η οποία ανοίγει νέους δρόμους ε, για μια νέα για μια άλλη χώρα για να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συνδράμει σε όλα αυτά αλλά και κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ε, τύχει υποστήριξης ιδιαίτερα για τις χώρες ε, για τις οποίες θα πρέπει να ανοίξουν νέα κεφάλαια. Μιλώ για τις υποψήφιες χώρες. Θα υποστηρίξουμε τις υποψήφιες χώρες προς αυτή την κατεύθυνση. Με ρωτήσατε για την αναχέτηση των μη δημοκρατικών δυνάμεων και των αντιευρωπαϊστών. Νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές ε, πολιτικές πλησιάζουν τον πολίτη. Θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τον πολίτη και να ενημερώνουμε τους πολίτες ε, για τα μέτρα που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην Ευρώπη γιατί έχουμε να κάνουμε με μια Ευρώπη των πολιτών. Αυτή την οδό θα πρέπει να ακολουθήσουμε αν θέλουμε να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες. Και έτσι θα υπερισχύσουμε εκείνων που είναι αντιευρωπαϊστές και δεν δέχονται τις ε, δημοκρατικές διαδικασίες. Ο κύριος ε, ε, Γιόγκμαν από το ECR μου υπέβαλε μία ερώτηση. Νομίζω ότι μπορούμε να ορίσουμε καλύτερα τις επενδυτικές ανάγκες. Έχουμε πολλούς δημάρχους εδώ και νομάρχες οι οποίοι τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά γιατί προσέλκυσαν επενδύσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και έτσι η αποκέντρωση είναι ένα νέο ε, δυναμικό βήμα. Αρχίσαμε την αποκέντρωση από πέρσι στη, χώρα μου, στη χώρα μου και θα επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία, λέει η Πρωθυπουργός χωρίς μικρόφωνο και είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή η οδός λαμβάνει υπόψη τις κοινέ αρχές και ανάγκες που διέπουν τις περιφέρειες. Κύριε Πρώτε Αντιπρόεδρε, βεβαίως η Φιλανδία ακολουθεί της Ρουμανίας στην Προεδρία. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά και με εσάς και με την Κροατία και θα οριοθετήσουμε το πρόγραμμα για τους επόμενους 18 μήνες. Θα κλείσουμε τη στρατηγική ατζέντα 14-19 και θα ανοίξουμε τη στρατηγική ατζέντα 2019-2024. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία μεταξύ Ρουμανίας, Φιλανδίας και Κροατίας. Είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο αν θέλουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και στο τέλος της θητείας και είμαι πεπισμένη ότι όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η Επιτροπή Περιφερειών και Πόλεων οι Εθνικές Επίτροπες θα προωθήσουν αυτή τη στρατηγική ατζέντα όπως ίσχυε μεταξύ 14 και 19. Παράλληλα θα σκιαγραφίσουμε τη νέα στρατηγική ατζέντα και ο στόχος για τους επόμενους 18 μήνες είναι να ορίσουμε ένα κοινό πλαίσιο δράσης με τη Φιλανδία και την Κροατία. Ο κύριος Δρακίτσι υπέβαλε μία ερώτηση. Η διάσκεψη με τη συμμετοχή της Μολδαβίας είναι πολύ σημαντική. Όπως ξέρετε, η Ρουμανία είχε μία κοινή συνεδρίαση με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Υποστηρίζουμε τη Δημοκρατία της Μολδαβίας για να ε, γίνει υποψήφια χώρα για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένους στόχους για τους ε, φίλους μας ε, πέρα από τον ποταμό Προύτ. Αυτός είναι ένας ε, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προωθήσουμε αυτούς τους κοινούς στόχους. Ε, για τη Μαριάννα Γκάζου. Μαριάννα, μίλησες ε, πολύ πατριωτικά υπέρ της ε, Ρουμανίας και είμαι σίγουρη ότι μετά την επίσκεψη των μελών θα δείτε όλοι τι έχουμε καταφέρει. Τώρα, σε σχέση με τις θεωρήσεις και το χώρο του Σέγγεν. Από το 11 και μετά η Ρουμανία πληρεί όλους τους όρους προσχώρησης και αυτό το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς η απάντηση και η απόφαση είναι πολιτικής υφής. Εμείς προσπαθήσαμε να προωθήσουμε τη δική μας υπόθεση γιατί πληρούμε όλους τους όρους. Θα θέλαμε λοιπόν να προσχωρήσουμε στο χώρο Σέγγεν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και πιστεύω στις δηλώσεις του Ζαν claude Juncker, ο οποίος είπε ότι σε αυτό το στάδιο θα πρέπει η Ρουμανία να προσχωρήσει στο χώρο Σέγγεν και το ίδιο έγινε και από τον Αντώνιο Ταγιάννη, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω να ληφθεί αυτή η απόφαση πολιτικής υφής γιατί μιλάμε για ενότητα και συνοχή και δεν μπορούμε να απεκδηθούμε των ευθυνών μας. Ο κύριος μίλησε για το κράτος δικαίου. Ε, επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει πολλές φορές. Στη Ρουμανία τηρείται το κράτος δικαίου και αυτό είπα και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε οποιοδήποτε κράτος τα δικαιώματα των πολιτών θα πρέπει να την χάνουν σεβασμού και αυτό αφορά και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Εγώ ως Πρωθυπουργό έχω λάβει υπόψη όλες αυτές ε, τις πτυχές και το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτών καθώς και η καταπολέμηση της διαφοράς διαφθοράς αποτελούν για μένα προτεραιότητα. Σε σχέση με την Επιτροπή της Βενετίας θα ήθελα να πω ότι η Ρουμανία, η δημοκρατία της Ρουμανίας ε, ποτέ δεν αθέτησε αποφάσεις του δικαστικού και δεν έχουμε παρέμβει στον δικαιοδοτικό τομέα πάντα στηρίζαμε τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Όλες αυτές οι κατηγορίες κατά της ρουμανικής κυβέρνησης, όλες αυτές οι κατηγορίες είναι αβάσιμες. Κύριε Μακάρθη, προτείνεται ένα πρόγραμμα δράσης για τις μικρές και μεγάλες πόλεις και ε, μιλάτε και για την υποστήριξη της πολιτικής συνοχής. Ήμουνα ευρωβουλευτής για εννέα χρόνια και συμμετείχα και στην Περιφερειακή Επιτροπή. Είχα υποβάλει πολλές τροπολογίες υπέρ της πολιτικής συνοχής. Για μένα η πολιτική συνοχής καθώς και η ΚΑΠ είναι στρατηγική σημασίας και ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση και χαίρομαι διότι στην Επιτροπή Περιφερειών συγκλίνετε και εσείς και ακολουθείτε αυτή την κατεύθυνση καθώς ε, ε, και διαβλέπω μία υποστήριξή σας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει η κατάλληλη χρηματοδότηση έτσι ώστε να προωθήσουμε τη συνοχή μεταξύ ε, Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης και ιδιαίτερα των περιφερειών που είναι λιγότερο αναπτυγμένες. Και αυτό αφορά και τη συνεργασία κοινοτήτων και πόλεων. Η συνοχή είναι ύψης της σημασίας θα πρέπει να υπάρχει ε, ουσιαστική σύνοχη και αυτό ακριβώς θα προωθήσει η Ρουμανική Προεδρία μέσα στα πλαίσια της εκπεριτροπής ε, προεδρίας της. Εμείς επίσης θα είμαστε ε, αμερόληπτος διαμεσολαβητής όπως ε, επιβάλλεται για όλες τις προεδρίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να λάβετε υπόψη ότι στη Ρουμανική Προεδρία στο πρόσωπό μας δεν έχετε μόνο έναν φίλο αλλά και μία δύναμη υπέρ της Ευρωπαϊκής Συνοχής και Οικοδόμησης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρωθυπουργέ για τις απαντήσεις που μόλις δώσατε όσον αφορά τις διάφορες παρεμβάσεις που έκαναν τα μέλη μας. Με μεγάλη χαρά ήδη προετοιμαζόμαστε να έρθουμε 14 με 16 Μαρτίου στην, ε, ε, στο Βουκουρέστι για την διάσκεψη κορυφής. Θα μου επιτρέψετε τώρα να συνοδεύσω την ε, κυρία Πρωθυπουργό και βεβαίως σας αφήνω στα έμπειρα χέρια του αντιπρόεδρου μας ε, ε, Μάρκουλα. Και βεβαίως ακόμα έχουμε πολλή δουλειά, έχουμε αργοπορήσει, είμαστε πίσω κατά δύο γνωμοδοτήσεις. Right, uh, ladies Κυρίες και κύριοι αξιότιμα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών έχουμε πολλές νομοδοτήσεις για το απόγευμα θα πρέπει να γίνει και μια αλλαγή στη σειρά θα εξετάσουμε τώρα την νομοδότηση που θα βλέπουμε στις 6 κανονικά βέβαια της Άννα Μάγιαρ είναι εδώ και η Ρομπέρτα Μετσόλα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό και μετά θα δούμε τις δύο γνωμοδοτήσεις για το ΣΕΝΤΕΞ του Γιάννος ε, Καρασόνη και της Ούλρη και Χίλερ και μετά έχουμε συμφωνήσει με τον Μάικαλ Σέλερ ότι ε, Σέφερ μάλλον ότι η δική του Ονομοδότηση θα εξεταστεί αύριο. Κατά τα λοιπά, δεν θα αλλάξει κάτι στη μέση διάταξη. Με τη σειρά Μπιργκίτα Σακρεντέου, Γιάνν Τρέαη, Όλγερ Γκέμπλεβιτ αργότερα σήμερα. Με τη σειρά, όπω το λέμε στη μέση διάταξη. Λοιπόν, εφόσον συμφωνείτε, και σα ευχαριστώ που συμφωνείτε, να καλωσορίσω την Άννα Μάγκιαρ Λοιπόν, μόλις είναι έτοιμη η Άννα μπορεί να ξεκινήσει με μια σύντομη εισαγωγή και μετά την παρουσίασή σας θα έχουμε και τη συνεισφορά της Ρομπέρτα Μετσόλα. Άννα, έχεις το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μπορέσω να σας μιλήσω σήμερα για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και τον σχετικό κανονισμό διότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και σε περιφερειακό επίπεδο, όχι μόνο σε εθνικό. Είναι σημαντικό δηλαδή σε περιφερειακό επίπεδο να δούμε πώς οι ε, παραμεθόριες περιοχές ε, ε, διαχειρίζονται τη φύλαξη των σύνορων για να εξασφαλίσουμε ότι τα εσωτερικά μας σύνορα μπορούν, μπορούμε συνέχεια να τα διαβούμε ελεύθερα για να συμβεί αυτό πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Βεβαίως η Frontex είναι εδώ για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια. Το έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την Frontex για να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματική ε, στην προσπάθειά της αυτή ε, φύλαξης ε, των εξωτερικών συνόρων. Έχουμε λοιπόν αυτή την γνωμοδότηση και εγώ προσπάθησα εδώ να δώσω ε, ιδιαίτερη έμφαση στην κατανομή των ρόλων, των αρμοδιοτήτων ε, και βεβαίως τονίζω τη συνεργασία που είναι απαραίτητη μεταξύ των ε, διαφόρων εμπλεκομένων φορέων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε μια σειρά από εξουσίες, αρμοδιότητες στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στην Frontex. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να καταλάβουμε ότι η Frontex και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πολιτικά όργανα. Δηλαδή θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ουδέτεροι θεσμοί. Εφόσον δοθούν εξουσίες στην Frontex, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εδώ έχουμε μία εικόνα ατελή. Έχουμε ένα κενό, διότι υπάρχει ο τεχνικό σκέλος και το πολιτικό σκέλος. Και αυτό βεβαίως αποτυπώνεται στην γνωμοδότησή μου. Προσπάθησα λοιπόν να ενσωματώσω τις ε, τροπολογίες τις πιο σημαντικές στη γνωμοδότηση αναφέρομαι σε τέσσερις κατηγορίες και όχι τρεις κατηγορίες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μέτσολα για τη συνεργασία. Έχω ενσωματώσει αυτή την πρόταση ε, στην γνωμοδότηση. Θα ήθελα να πω ακόμα κάτι. Ήταν πραγματικά μια πολύ καλή εμπειρία η συνεργασία με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στο γραφείο ε, της Frontex στη Βαρσοβία. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Αυτά για τη γνωμοδότηση σε γενικές γραμμές. Το τελευταίο κομμάτι έχει και ένα πολιτικό ε, σκέλος, ένα μια πολιτική δήλωση. Ευχαριστώ Άννα, ευχαριστώ πολύ και τώρα η Ρομπέρτα Μέτσολα έχει το λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μάγιαρ. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ιστορία αυτή για ένα θέμα που μας αφορά όλους. Το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία ε, δεν γνωρίζουν σύνορα από τη μία χώρα στην άλλη, από τη μία ήπειρο στην άλλη. Και βεβαίως ε, υπάρχει το θέμα τη μετανάστευση που είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα αυτής της γενιάς, που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αν το δούμε σφαιρικά. Είτε μιλάμε για τις ΗΠΑ, ε, είτε μιλάμε για την Αφρική και την Ευρώπη. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνο με μια σφαιρική παγκόσμια προσέγγιση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε απλά να μιλάμε χωρίς να παίρνουμε αποφάσεις. Αποφάσεις σε βάθος χρόνου και όχι ε, σπασμωδικές αντιδράσεις. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα της μετανάστευσης από μια μέρα στην άλλη. Στην Ευρώπη, εάν θέλουμε να είμαστε ένα παράδειγμα για τον κόσμο, αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η δική μου θέση ως εισηγήτρια για το θέμα αυτό, αλλά και ως ε, συντονίστρια του ΕΛΚ στην Επιτροπή Ελευθεριών του Κοινοβουλίου, είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της μετανάστευσης σφαιρικά και ισορροπημένα. Θα πρέπει δηλαδή να ενσωματώσουμε, να λάβουμε υπόψη μας και τις ηθικές υποχρεώσεις που έχουμε και τους ε, θεμητούς φόβους για την ασφάλειά μας. Άνθρωποι είμαστε το κάτω-κάτω. Πρέπει να φανούμε δίκαιοι απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται προστασία. Πρέπει όμως να είμαστε και σκληροί απέναντι σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τους πιο ευάλωτους. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με αυτή τη νομοθεσία, την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και φυλακή είναι ακριβώ αυτό η πρόταση αυτή έχει φτάσει στο Κοινοβούλιο, προχωράει η εξέτασή της. Ο στόχος είναι να ενισχύσουμε την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και να επιταχύνουμε την επιστροφή των μεταναστών που δεν χρήζουν προστασίας. Μετά ε, το σχέδιο εξέτασης, ε, σχέδιο γνωμοδότησης τον, τον Νοέμβριο στο Κοινοβούλιο στην Επιτροπή είχαμε ε, πάρα πολλές ε, τροπολογίες. Προφανώς πολλά μέλη από όλες τις πολιτικές ομάδες ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, παρακολουθούν την πρόοδο που έχει σημειωθεί επί αυτής της νομοθετικής έκθεσης. Πάντως συνεχίζονται οι εργασίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην φάση της ολοκλήρωσης των ε, συμβαστικών τροπολογιών και σε τεχνικό και σε πολιτικό επίπεδο για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή στο Στρασβούργο. Και βεβαίως σας διαβεβαιώ ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική νομοθεσία και γι' αυτό ε, την αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα προσοχή. Έχουμε υποβάλει μια σειρά από τροπολογίες που ελπίζουμε να συμπεριληφθούν στην νομοθεσία. Ακούμε τη λένε και οι υπόλοιποι όμως. Ακούμε και την Επιτροπή των Περιφερειών αλλά και άλλους εμπλεκόμενους φορείς που επίσης έχουν υποβάλει τροπολογίες που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην νομοθεσία. Ελπίζουμε να μπορέσει αυτή η νομοθεσία να τελεσφορήσει πριν τις επόμενες ευρωεκλογέ. Θέλουμε να δώσουμε την απαραίτητη ευελιξία έτσι ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε δυνάμεις ε, σε, μία, σε κάποια σύνορα που βρίσκονται υποπίεση. Έχει σημειωθεί πρόοδος το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν συνεισέφεραν όμως ούτε σε ανθρώπινους πόρους ούτε σε εξοπλισμό ε, έχει οδηγήσει ε, στο να μην είναι αρκετά αποτελεσματικές οι κοινέ επιχειρήσεις του, της Frontex Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των συνοριοφυλάκων, της ακτοφυλακής και να έχει μια ενισχυμένη ε, εντολή αυτή η δύναμη θα πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τα εξωτερικά μας σύνορα και να εξασφαλίσουμε την επιστροφή όσων έρχονται στην Ευρώπη για να έχουμε ενισχυμένη ασφάλεια στην Ευρώπη. Προτείνουμε μια σειρά από αλλαγέ, δίνοντας στον οργανισμό αυτό ε, το δικό της επιχειρησιακό βραχίωνα με εκλεστικές εξουσίες ε, για τις δραστηριότητε τους για να μπορούν να υποστηρίξουν πραγματικά ε, τα κράτη-μέλη. Αυτό το σώμα δεν πρέπει να αυξηθεί μόνο ποσοτικά. Πρέπει να έχει τις απαραίτητες δυνατότητες, τις αρμοδιότητες να παρέμβει όποτε χρειάζεται για να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα, για να μπορέσουμε να προλάβουμε δευτερογενείς μετακινήσεις και να εφαρμόσουμε στην πράξη την ε, ε, επιστροφή των παράνομων μεταναστών. Είναι το πρώτο ζήτημα η ασφάλεια. Αυτό λένε οι συμπολίτε μα. Αυτό μα λένε στα κράτη-μέλη. Είναι το πρώτο στοιχείο ανησυχία. Θα πρέπει λοιπόν αυτή την ανησυχία εμεί ε, να την καλύψουμε για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τη Σέγγιν και την ελεύθερη κυκλοφορία ε, στο εσωτερικό τη Ένωση. Χρειάζεται αμοιβαία εμπιστοσύνη λοιπόν μεταξύ κρατών μελών και γι' αυτό πρέπει να ασφαλίσουμε, να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά μα σύνορα. Αυτό που συνέβη το 2015 με τη Συριακή κρίση ε, ε, ήταν η συνειδητοποίηση ότι ορισμένε φορέ ένα κράτο μέλο ε, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο του μια κατάσταση. Τώρα μπορεί να παρέμβει όμω αυτή η συνοριοφυλακή είτε κατόπιν αιτήματο ενό κράτου μέλου, είτε εφόσον οι αρχέ επιβολή του νόμου αξιολογήσουν ότι πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο, με τη σύμφωνη γνώμη του κράτου μέλου βέβαια, ότι πρέπει δηλαδή να συμβεί κάτι, να υπάρξει μια επέμβαση. Με τη νέα πρόταση ε, εδώ γεφυρώνουμε αυτές τις δύο ε, προϋποθέσεις. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι επειδή η Συρία και η Εμένη δεν είναι κοντά μας, δεν σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνη ή ότι δεν μας αγγίζει. Γιατί ο κόσμος ορισμένες φορές είναι μικρότερος από ό,τι νομίζουμε. Ε, μεταξύ των συμπολιτών μας, στα κράτη-μέλη, υπάρχει φόβος και θα ήταν λάθος να τα γνωρίσουμε όλα αυτά. Ο χώρος Σέγγεν μεταξύ των κρατών μελών πάει χέρι-χέρι με την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Τελειώνοντας, να πω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Στη συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση, είτε την νόμιμη είτε την παράτυπη, ε, αμέσως κυριαρχεί το συνέστημα ε, διότι ε, αφορά άμεσα τους ανθρώπους. Είναι εύκολο να κατηγορήσει κάποιον βέβαια τον ξένο για τα πάντα, αλλά πρέπει να δούμε πίσω από τη φτηνή αυτή η πολιτική εκμετάλλευση αυτών των ζητημάτων. Και βεβαίως ε, είναι καθήκον μου να υπογραμμίσω πάνω απ' όλα ότι η μετανάστευση πάνω απ' όλα είναι ένα ανθρώπινο ζήτημα. Μιλάμε για γυναίκες και άντρες δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι για κάθε στατιστικό στοιχείο που βλέπουμε, για κάθε αριθμό που βλέπουμε στις ειδήσει, από πίσω υπάρχει μια ζωή, μια ελπίδα, όνειρα για μια καλύτερη ζωή. Να μην ξεχνάμε ποτέ αυτό. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Πρόκειται για πολύ σημαντικό θέμα. Πράγματι θα έχουμε λοιπόν και άλλες παρεμβάσεις από τα μέλη μας. Έχω στη λίστα μου Γιάννος Αργίλαν κλπ. Μπορείτε να λάβετε και άλλοι τον λόγο. Ας αρχίσουμε με τον Γιάννο Σαργυράν. Έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Πρώτα, εξετάζοντας την πρόταση, θεωρώ ότι δείχνει με ποιον τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε πιο αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα. Αν εξετάσουμε πιο προσεκτικά, Νομίζω ότι καλούμαστε να αποφασίσουμε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε την μετανάστευση και πώς θα μεταφερθεί η σχετική αρμοδιότητα από εθνική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η μεταφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, αμφισβητείτε διότι έχει καθυστερήσει πολύ να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ την συνάδελφό μας Συγγετρία η οποία προσπάθησε να ξεκαθαρίσει την διαδικασία που είναι πολύ συγκεντρωτική. Αλλά όπως έχει τώρα η πρόταση δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει δεκτή. Ευχαριστώ. Βιντσέντσο Βιάνκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ ε, ε, με συγκίνηση μιλάω για το θέμα αυτό, γιατί ακριβώς στις 4 Φεβρουαρίου του 2001 δηλαδή ακριβώς 18 χρόνια πριν αν δεν κάνω λάθος, όταν ήμουν υπουργό Εσωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας σε μια συνάντηση με τον αρμόδιο επίτροπο, τον Αντώνιο Βιτορίνο από την Πορτογαλία, ξεκινήσαμε, ρίξαμε την ιδέα της δημιουργίας μιας σύγχρονης ε, ε, ευρωπαϊκής αστυνομίας των συνόρων. Πέρασαν 18 χρόνια. Με μεγάλη πικρία λοιπόν διαπιστώνω ότι ε, κάθε χώρα μεμονωμένα τα τελευταία αυτά χρόνια αναγκάστηκε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει που θα είχαν αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη ευκολία εάν υπήρχε ήδη αυτή η αστυνομία των συνόρων. Χειροκροτώ λοιπόν αυτό το κείμενο, αυτόν, αυτή την πρόταση, αυτόν τον κανονισμό και ζητώ από την Επιτροπή Περιφερειών να δείξει θάρρος έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή αστυνομία. Στην γνωμοδότηση της συναδέλφου βρίσκω κάποια θετικά στοιχεία. Ωστόσο βρίσκω και έλλειψη θάρρους, βρίσκω και μεγάλο βαθμό δηλίας ε, για να ε, ενστερνιστούμε αυτήν την έννοια της πραγματικής ε, ευρωπαϊκής αστυνομίας η ψήφος μου θα εξαρτηθεί από την τύχη που θα έχουν οι υποβληθείς τροπολογίες. Θα πρέπει και μέσω των τροπολογιών να ενισχύσουμε την ιδέα ότι μαζί από κοινού θα πρέπει να ε, ε, αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και το θέμα των πλοίων ε, όπως του Sea-Watch ας πούμε δεν θα πρέπει να είναι μεμονωμένης χώρας πρόβλημα. Η Ευρώπη σαν σύνολο θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και δυστυχώς Πρόεδρε με μεγάλη πικρία. Θα καταψηφίσω εάν χρειαστεί. Ευχαριστώ κύριο Φράγκο Γιάκοπ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στην Επιτροπή ΣΥΒΕΞΕ είχαμε συζητήσει για το κατά πόσον η Επιτροπή Περιφερειών θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει όσον αφορά αυτή την πρόταση κανονισμού που εκ πρώτη όψεω αφορά αρμοδιότητα αποκλειστικά των κρατών μελών. Ωστόσο, διάφορε σκέψεις μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε ε, να ε, συζητήσουμε το θέμα αυτό γιατί και εμείς θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μέρο του προβλήματος αλλά και γιατί ω τοπικές περιφερειακές αρχές αλλά και γιατί θα πρέπει να είμαστε ε, συνεκτικοί με προηγούμενες προτάσεις ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να κινηθούμε ταυτόχρονα ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το χρονοδιάγραμμά του. Ε, και επομένως στην ουσία στην Επιτροπή Σύβεξε κάναμε μονάχα μια γενικής φύσεως συζήτηση αλλά δεν μπορέσαμε να υποβάλλουμε τροπολογίες ή να υποβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Σε σχέση με τη γνωμοδότηση της συναδέλφου Μαγιάρ, την οποία θα θέλαμε βεβαίως να ευχαριστήσουμε για την εργασία της, ε, βρίσκουμε ε, κάποια σειρά ε, γενικών παρατηρήσεων τις οποίες δεν μπορούμε να συμμεριστούμε, διότι η ουσία των τροπολογιών ε, στην ουσία θέλει να μειώσει ε, την ε, λογική της προσπάθειας έτσι ώστε να περιοριστούν σε πιο εθνικά επίπεδα. Αυτό δεν μπορούμε να το συμμεριστούμε τη στιγμή που η συζήτηση που κάνουμε είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε και αυτή είναι η συζήτηση που κάνουμε να δημιουργήσουμε λέω έναν κοινό χώρο ευρώ, εντός του οποίου θα γίνεται και μια κοινή διαχείριση της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Ε, ε, ε, αντιθέτως βλέπουμε ενίσχυση θεμάτων όπως είναι το κλείσιμο των συνόρων, η μείωση των μεταναστευτικών ροών, η πίεση επί των μεταναστευτικών. Τον Δεκέμβριο του 2018 είχαμε την έκθεση Μπόσμαν η οποία ακριβώς έλεγε ότι δεν θα πρέπει να βασιστεί η πολιτική για τους μετανάστες μονάχα σε θέματα ε, ασφάλειας ή να είναι μονάχα εθνικά, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια ενσωμάτωση ε, των ε, μεταναστευτικών πολιτικών. Ε, e. επίσης πρέπει να σας πω ότι η σοσιαλιστική ομάδα θα καταψηφίσει την ίδια τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ ο Κριστόφρου Γιόν. Oui, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αργήσαμε πολύ όσον αφορά την πρόσταση των συνόρων. Επανειλημμένα έχω πει ότι κάποιε χώρε και πολιτικέ ομάδε ε, ε, είχαν εκφράσει την ανησυχία τη διασφάλιση των ε, συνόρων έτσι ώστε να προστατευτούν από την άφηξη παρανόμων μεταναστών. Τώρα βλέπουμε ε, ότι μιλάμε για 10.000 ε, συγγνώμη, ε, ακτοφύλακες και συνοριοφύλακες και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι εκεί απλώς για να δώσουν έτσι μια χαριτωμένη νότα στα σύνορα, είναι εκεί για να δουλέψουν. Υπάρχουν κάποιες αρχές βεβαίως δημοκρατικές ε, τις οποίε είναι προσφυλή σε κάθε χώρα, αλλά βεβαίω θα πρέπει και αυτοί ε, οι αστυνομικοί να έχουν την δυνατότητα ε, να δράσουν και βεβαίω θα πρέπει να υπάρξει και συντονισμό σε Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένω σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω εμεί θα αντιταχθούμε σε οποιαδήποτε γνωμοδότηση ή οποιοδήποτε κείμενο που δίνει μονάχα ρόλο κομπάρσου σε αυτού του συνοριοφύλακε και ακτοφύλακε. Τρει ακόμη παρεμβάσει από David Simmons, Φρανσουά Ντεκοστέρ και Σπέργερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει δεσμευμένο στην στήριξη των ευρωπαϊκών προσπαθειών για την διαχείριση και προστασία των συνόρων μας. Σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση, η συγγήτρια έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην εξέβρεση ισορροπίας πράγματι σε ένα ευαίσθητο θέμα. Σημαντικό είναι το θέμα αυτό για μας εδώ την Επιτροπή Περιφερειών, διότι οι περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις είναι εκείνες οι οποίες καλούνται να πληρώσουν το τίμημα όταν δεν προστατεύονται επαρκώς τα εξωτερικά σύνορα των χωρών μας. Η πρωτοβουλία αυτή η οποία θα προσφέρει περισσότερη στήριξη σε μια εθνική αρμοδιότητα είναι σωστή. Είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο μεταναστευτικό μετακινούνται γεωγραφικά και αλλάζουν και κατά την φύση τους. Έτσι λοιπόν, μία χώρα μέλος προσπαθεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή, χρειάζεται να έχει πρόσβαση και στους σχετικούς πόρους. Νομίζω τελικώ είναι σημαντικό να το δούμε αυτό μέσα στο πλαίσιο και του υπολείπου έργου που διεξάγεται εδώ στην Επιτροπή Περιφερειών. Και διμερές, και γνωρίζω ότι πολλοί από του συναδέλφου μα στην Γαλλία που εκπροσωπούν λιμάνια έχουν ε, πολύ δουλέψει για το θέμα αυτό και συζητούμε με τις γειτονικές μας χώρες για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η συνεργασία μας στο μέλλον. Από την άποψη λοιπόν της ομάδας του ECR και του Ηνωμένου Βασιλείου χαιρόμαστε για την έκθεση και θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε συνολικά και να αποτελέσει βάση για τις περαιτέρω εργασίες μας στο μέλλον. Φρανσουά Ντεκοστέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαγιάρ, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πρώτα την εισηγήτρια, διότι το θέμα βεβαίως είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Προσπαθούμε δηλαδή να οικοδομήσουμε μια πιο αποτελεσματική Ευρώπη. Εδώ και χρόνια άλλωστε εγώ ακούω να μιλούν για την ανάγκη ε, δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής διότι αυτό θα δείξει και αποτελεσματικότητα. Ε, εκφράζω την εκκλησία μου σήμερα, διότι για να δημιουργηθεί αυτή η αποτελεσματική Ευρώπη, αναζητούμε πρώτα την απεικοδόμησή τη, την αποδόμησή τη. Για να γίνει μια, για να φτιαχτεί μια αποτελεσματική Ευρώπη, ωστόσο πρέπει να τη διατεθούν πλέον αποτελεσματικά ευρωπαϊκά μέσα. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι υπάρχει μια λογική στην έκθεση της ε, κυρίας Μαγιάρ, μια λογική όμως που δεν επιθυμώ να ακολουθήσω διότι η αποτελεσματικότητα θα σήμαινε να υιοθετήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ ανοίγοντα τον δρόμο για την αποδόμησή της σημαίνει ότι στερούμε από τους πολίτες τη δυνατότητα χρήσης ενός αποτελεσματικού μέσου ενώ η αποτελεσματική προστασία των συνόρων τη χρειάζεται. Γι' αυτό προτείνω στην συνάδελφό μας Μαγιάρ να αποσύρει την 2R, 9R και 14R τροπολογίες για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε έτσι και εμείς υπέρ της εκθεσής της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο Φραντ Σάουσπεργκερ. Δεν θα ήθελα ακόμη να μπω στις λεπτομέρειες των τροπολογιών. Θα ήθελα να πω κάτι, ας πούμε, επί της αρχής. Και πρώτα συγχαίρω την Άννα Μαγκιάρ που νομίζω ότι πραγματικά κατέβαλε προσπάθεια για να συντάξει μια καλή γνωμοδότηση που αποτελεί και την βάση για μια αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων καθώς και μια ε, αποτελεσματική ε, ε, πολιτική επιστροφών. Είναι καλά αιτιολογημένα αυτά. Δυστυχώς οφείλω να πω όμως ότι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει δεν είναι απολύτω λογικό σε όλα τα σημεία, διότι αν όλοι είμαστε υπέρ της αποτελεσματική προστασίας των εξωτερικών σύνορων και αν θέλουμε να ε, γίνει σωστή και λογική πολιτική επιστροφών, χρειαζόμαστε ισχυρή Frontex. Δεν βοηθεί κανένα να προστατεύσουμε τα εσωτερικά μας σύνορα, αλλά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί χρειαζόμαστε πραγματικά έναν αποτελεσματικό Frontex. Και επισημαίνω επίσης ότι η Αυστριακή Προεδρία, η οποία μέχρι τέλους κατέβαλε προσπάθειες για την εξέβρεση δίσως ώστε ήδη από το 2020 να έχουμε τους 10.000 συνεργάτες της Frontex για τον αποτελεσματικό έλεγχο και προστασία των συνόρων. Δεν μπόρεσε βέβαια να καταστεί δυνατόν αυτό στο Συμβούλιο Υπουργών. Δεν μπόρεσε δηλαδή να εξευρεθεί η αναγκαία πλειοψηφία ή ομοφωνία. Συμφωνώ με τις αιτιολογίες που προτείνει στην έκθεσή της η Άννα Μάγκερ. Θεωρώ όμως ότι θα έπρεπε να καταλήγει σε άλλο συμπέρασμα. Αυτό θα τα συζητήσουμε και ε, λεπτομερώς, αλλά θεωρώ και θέτω και το ερώτημα, αν όντω είναι σκόπιμο, σε μια γνωμοδότηση να επισέλθουμε μέχρι και τις τελευταίες λεπτομέρειες για το πόσο θα πρέπει να απασχοληθεί ο συγκεκριμένος ε, συνεργάτες του Frontex και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να πούμε δηλαδή τι θέλουμε ως αρχή, ως βασική αρχή και μετά να παραπέμψουμε το όλον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στις τροπολογίες και η συγκήτρια να τοποθετηθεί επί ορισμένων αλλαγών, εφόσον χρειάζεται αν τι θέλατε να αντιδράσετε αμέσως. No, οκ. Α, ναι, θα ήθελα τώρα να πω κάτι, λέει η κυρία Μαγιέρ. Ορίστε λοιπόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αντιδράσω έτσι εν συντομία σε αυτά που ακούστηκαν. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους για τις συνεισφορές σας Νομίζω ότι κατέστατε σαφές ότι το θέμα αυτό είναι δύσκολο. Είναι ιδιαίτερο και σημαντικό για όλους μας. Ε, κύριε Αγγιλάν, να σας πω ότι δεν νομίζω ότι το κείμενο αυτό είναι αδύναμο. Προσπάθησα να επικεντρωθώ στα πιο σημαντικά στοιχεία και νομίζω ότι η Frontex πρέπει να έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει να υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά ε, την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Σε ό,τι φορά τώρα στη συνεργασία προσπαθούμε να εργαστούμε ακριβώς σε αισθήματα συνεργασίας ε, σε αυτό το κείμενο. Νομίζω ότι όλοι έχουν ένα ρόλο να παίξουν. Αναφέρομαι στο Συμβούλιο, ε, στην Κομισιόν και στη Frontex το κείμενο, στην αρχική πρόταση δεν γίνονταν αναφορά στο Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι η συνεργασία είναι αυτό που μετράει εδώ. Εγώ έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να επικεντρωθώ ακριβώς σε αυτό το ζήτημα της συνεργασίας. Κύριε Καπούρ τώρα, κύριε εμείς ε, δεν δίνουμε, δεν μοιράζουμε αρμοδιότητες και εξουσίες. προσπαθούμε να ενισχύσουμε την Frontex χωρίς να στρεβλώσουμε τις αρμοδιότητες που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Διατηρούμε την ίδια κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων. Θέλουμε απλώς να δώσουμε μεγαλύτερη υποστήριξη στη Frontex για να αντιμετωπίσει τεχνικά ζητήματα. Δεν μιλάμε όμως εδώ για τις, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες ε, της αρχής αυτής. Κάποιος αναφέρθηκε στην εθνική κυριαρχία. Βεβαίως και είναι σημαντική η εθνική κυριαρχία, όπως και η συνεργασία. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει η Frontex εδώ ε, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ο κύριος Σίμενς αναφέρθηκε προηγουμένως ε, στις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα σε περιφερειακό επίπεδο ως περιφερειακοί πολιτικοί άρχοντες ε, με το θέμα των συνόρων τότε το συζητούμε ε, με την κυβέρνηση της χώρας μας. Εάν όμως ε, ε, οι αρμοδιότητες αυτές ε, είναι και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε απευθυνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν τις αρμοδιότητες αυτές αναλάβει όμως η Κομισιόν τελικά, τότε μπαίνει θέμα επικουρικότητας. Κύριε Ντεκώστα, ε, δυστυχώς δεν μπορώ να αποσύρω τις τροπολογίες μου τις τροπολογίες μου ως εισηγήτριας οι τροπολογίες αυτές δείχνουν ότι προσπάθησα να βρω ε, στοιχεία από τις δικές τροπολογίες και να τις να, τα ενσωματώσω στο κείμενο και ε, απομακρύνθηκα από τις αρχικές μου τροπολογίες και διατυπώσεις. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα των διαφορών αρχών. Ε, δέχτηκα λοιπόν αυτά που πρέπει αλλά όχι πλήρως. Αυτό είναι και το νόημα μια συμβαστική τροπολογία. Οπότε δεν μπορώ τώρα να αποσύρω ε, τις τροπολογίες αυτές. Νομίζω δεν έχει νόημα να εγκρίνουμε την πρόταση της την αρχική της Κομισιόν ως έχει. Να ευχαριστώ και τον, τον κύριο Σάουσμπεργκερ για την υποστήριξη. Νομίζω ότι θα εξετάσουμε ε, τα διάφορα σημεία και θα δούμε τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα περνάμε στην ψηφοφορία επί των τροπολογιών. Η πρώτη τροπολογία υπαριθμών 1 έχει αποσυρθεί. Ο κύριος Μιλάνο, ναι για το 2, για το 2 πρόεδρε, για το 2 θέλω να μιλήσω εγώ, για την τροπολογία 2. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Ε, περνάμε λοιπόν στην επόμενη τροπολογία 2R του εισηγητή, εφόσον εγκριθεί τη 2 και η 11 και η 4 αλλά και η 10 καταπίπτουν. Ε, κύριε Μιλάνο. Ευχαριστώ. Εδώ έχουμε μια πρώτη, ένα πρώτο υπόδειγμα τροπολογίας ε, άρα που δεν λαμβάνει υπόψη ναι, τα όσα ε, υπόθηκαν ε, στην τροπολογία 2 του συναδέλφου Μπιάνκο. Στην ουσία δηλαδή έπανα υποβάλει το κείμενο της εισηγητρίας. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση και διαμεσολάβηση ας πούμε. Ε, εδώ με αυτήν την πρόταση βλέπουμε οπισθοδρόμηση ενώ εμείς πρέπει να εμπλουτίσουμε την ε, γνωμοδότηση. Δηλαδή αν περάσει η τροπολογία της εισαγητρίας αποδυναμώνουμε το κείμενο. Επομένως κάνω μία έκκληση Όπω και ο συνάδελφο από την, από την Άλντε. Δηλαδή να αποσύρει η συγγήτρια αυτήν την τροπολογία. Εάν δεν ε, αποσύρει την τροπολογία η συνάδελφος ε, ε, η συγγήτρια, θα προτείνω να ψηφίσω, στου συναδέλφου προτείνω να ψηφίσουν την τροπολογία Μπιάνκο. Εντάξει, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Μαγιάρε, κυρία εισηγήτρια, παρακαλώ ένα σχόλιο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να διατηρήσω αυτήν την ε, ε, τροπολογία. Είναι μια τροπολογία που έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμεσολάβησης και επομένως θεωρώ ότι είναι συμβιβαστική. Ε, γιατί θα πρέπει το κράτος υποδοχής να έχει αυτές τις αρμοδιότητες. Ωραία, να ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ, υπέρ του 2R. κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό you can start voting. άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 2R της ηγετρίας Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Επομένως έχουμε τροπολογία κατά και επομένως απορρίπτεται η τροπολογία 2R. And uh, then we vote. Προχωράμε λοιπόν. Ε, ψηφίζουμε την τροπολογία 2. Η υπέρ της τροπολογίας 2 παρακαλώ ψηφίστε. Υπέρ. Σας ευχαριστώ κατά. Η τροπολογία είναι υπέρ και επομένως εγκρίνεται η τροπολογία 2. Τροπολογία 3. Υπέρ. Ψηφίστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ψήφι κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 4. Υπέρ. Κατά. εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθμών 5 υπέρ κατά απερίφθη. Τροπολογία 6 υπέρ Thank you. Σας ευχαριστώ. Ψήφι κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας. Η τροπολογία, η τροπολογία εγκρίνεται μια και την υπερψήφισαν οι περισσότεροι. Τροπολογίες 7 και 8 είναι ταυτόσιμες, επομένως ψηφίζονται από κοινού. Υπέρ. Ευχαριστώ. Ψήφι κατά. Η πλειοψηφία είναι υπέρ. Επομένως εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ναι, η συγκήτρια ζητάει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Επομένως ψηφίζουμε 7 και 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τις τροπολογίες 7 και 8. Πέρας της ψηφοφορίας. Η τροπολογία γίνεται δεκτή αφού η πλειοψηφία υπερψήφισε. Τροπολογία 9 άρα εάν υπερψηφιστεί οι τροπολογίες 10, 11, 12, 16 καταπίπτουν 9 R και 14R υπέρ. Thank you against. Κατά. Ναι. The majority is... Η πλειοψηφία καταψηφίζει, αλλά τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε χωριστά. Η 9 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 10 να ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ της 10 κατά εγκρίνεται η τροπολογία αυτή τροπολογία 11 υπέρ Ζητώ συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος η τροπολογία 11 καταπίπτει από τη στιγμή που εγκρίθηκε ήδη η τροπολογία 10. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 12. Δεν ψηφίσουμε την 11. 12 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 12. Okay, we close the vote. Πέρα ψηφοφορίας, η πλειοψηφία είναι κατά του κειμένου αυτού, επομένως απερίφθη. Τροπολογία υπερθμών 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 14, όχι, ναι, ναι. Την ψηφίζουμε τη 14. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 14 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία εγκρίνει. Είναι υπέρ. Επομένω εγκρίνεται. Α, αυτή η τροπολογία είναι ταυτόσιμη με την επόμενη, άρα ψηφίζουμε την 17. 17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20R. Εάν εγκριθεί η 20 καταπίπτει. Ψηφίστε παρακαλώ για την 20R. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επ' αυτού. Πέρας της Με μία ψήφο διαφορά η πλειοψηφία είναι υπέρ και επομένως εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 22 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 23 έχει αποσυρθεί. Άρα ψηφίζουμε την τροπολογία 24R. Εάν εγκριθεί θα καταπέσει η τροπολογία 24. Ψηφίζουμε λοιπόν την 24R υπέρ κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 24R. Μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. Πέρασε. Η τροπολογία, ε, συγγνώμη, η πλειοψηφία είναι κατά, επομένω ε, δεν έγινε δεκτή η τροπολογία. Άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 24 υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος ψηφίζει κατά. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 24. Πέρας της ψηφοφορίας. Η τροπολογία, η ψηφοψηφία συγγνώμη είναι υπέρ, άρα η τροπολογία γίνεται δεκτή. Τροπολογία 25R της εισηγητρίας. Ψηφίστε παρακαλώ για την 25R. Κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία και επομένως καταπέ... καταπίπτει η τροπολογία 25. Τροπολογία 26 υπέρ κατά εγκρίνεται η τροπολογία 26 Τροπολογία 27, άρτηση συγγετρίας, εάν εγκρίθει καταπίπτει η τροπολογία 27, ψήφι υπέρ της 27R. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 27R. Ψήφισαν όλοι, πέρα της ψηφοφορίας. Η τροπολογία απορρίπτεται. Άρα ψηφίζουμε την τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Η τροπολογία εγκρίνεται. Τροπολογία της συγκεντρίας 28 28R υπέρ κατά Εγκρίνεται, επομένως καταπίπτει 28 τροπολογία υπαριθμών 29, εάν εγκρίνεται η, καταπίπτει η τροπολογία 30 υπέρ της τροπολογίας 29, κατά η, ε, τροπολογία εγκρίνεται, επομένως η 30 πίπτη. ψηφίζουμε την τροπολογία 31, όχι, έχει αποσυρθεί, δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Η τροπολογία της εισηγήτριας υπαριθμών 32R. Ψηφίζουμε πρώτα αυτήν την τροπολογία της εισηγήτριας υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 34 υπέρ κατά εγκρίνεται τελική ψηφοφορία επί του συνόλου της τροποποιημένης γνωμοδότησης ψηφίζουμε ποιοι είναι υπέρ της γνωμοδότησης σας ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Α, έχουμε εδώ δύο αποχές. Διαφορετικά θα ήταν ομόφωνη η έγκριση. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν η τροπολογία αυτή. Ε, δούλεψε σκληρά η συγγήτρια αλλά και αυτοί που ε, υπέβαλαν τις ε, προτάσεις τροπολογιών. Συγχαρητήρια σε όλους. Ε, Uh, uh, Τώρα ακολουθεί η επόμενη γνωμοδότηση. Γιάννος Καρασόνη. Παρακαλώ να έλθεις εδώ, επάνω. Thank Oops.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 Right. Ο πρόεδρος. Ε, Καλώ λοιπόν. Ε, καλά το λέω το όνομά σα. Γιάννος Καραξόνη. Έχετε το λόγο για να μπορέσετε να κάνετε την εισαγωγή στην ε, εισήγηση, στη γνωμοδότησή σας μάλλον. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να απευθύνω τον λόγο σε εσά έχοντας συντάξει τη σημαντική αυτή γνωμοδότηση για λογαριασμό της ε, Επιτροπής Περιφερειών. Ήταν άλλωστε και μεγάλη πρόκληση η σύνταξη της ε, παρούσας γνωμοδότησης διότι συζητεί δύο σημαντικά έγγραφα. Το ένα είναι για την ε, τη δημιουργική Ευρώπη και το άλλο είναι εκείνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα πολιτισμού. Χρειάστηκε λοιπόν να συντάξω ταυτόχρονα. Σα παρακαλώ να σεβαστείτε τον ομιλητή, λέει ο πρόεδρο. Συνεχίστε και ελπίζω να γίνει κάπω ησυχία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την σημασία της συνεργασίας αλλά δεν νομίζω ότι, δεν, ότι μπορεί να αποφύγει κανείς να τονίσει τη μεγάλη σημασία των περιφερειακών και ε, ε, δημοτικών αρχών. Πρέπει οι άνθρωποι που ζουν και μακριά από τα αστικά κέντρα να έχουν επαρκή πληροφόρηση για τις δυνατότητες που ανοίγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προγράμματά της κλπ. Και να μπορούν και οι ίδιοι να εμπλέκονται στις λήψεις αποφάσεων. Για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη έχω ορισμένες σκέψεις γράψει στο χαρτί που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ο τομέας του πολιτισμού προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για την περίοδο 2021 έως ε, 27. Θα είναι ένα standalone program το οποίο θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για όλους τους δημιουργούς του καλλιτεχνικού τομέα. Για τον προϋπολογισμό νομίζω ότι η μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη και η ξεκάθαρη δέσμευση υπέρ της στήριξης των πολιτιστικών σημαίνουν ότι το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται θα πρέπει να αυξηθούν σε τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν εξετάσουμε τους τρεις διαφορετικούς τομείς, θα ήθελα να εκφράσω κάποιες ανησυχίες σχετικά με την, με την αναλογία των προτεραιοτήτων στον πολιτιστικό τομέα. Η το καινούργιο θεματολόγιο πολιτισμού αποτελεί τη βάση και επίσης θα ενισχύσει και εταιρικέ σχέσεις και συνεργασίες με εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάνει και τη σύνδεση και με άλλους τομείς όπως της παιδείας. Η ανακοίνωση τονίζει τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων καθώς και το ζήτημα της αποκατάστασης πολιτικής κληρονομιάς για να υπάρξει αύξηση της ανάπτυξης και άλλα σχετικά. Είναι αναγκαίο να περιλάβουμε σε αυτά και το θέμα της κινητικότητας. Μην το λησμονείτε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Μπορούμε να περάσουμε αμέσω στην ψηφοφορία των τροπολογιών. Ας ε, το κάνουμε λοιπόν. Ε, ε, μαζί ένα και δύο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Κανεί εγκρίνονται λοιπόν. Υπάρχουν τρία. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Η ε, πλειοψηφία είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τέσσερα. έχει αποσυρθεί. Δεν ψηφίζεται. Υπαριθμόν πέντε ψήφι υπέρ. Κατά. Εδώ θα χρειαστεί ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ναι, εδώ στο 5 το παρόν κείμενο λέει έως το Δεκέμβριο του 2020. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος προγράμματος, τα κράτη-μέλη χρειάστηκαν να σε επιμέρους περιπτώσεις ε, χρηματοδότηση, οικονομική υποστήριξη. Τον Οκτώβριο το κείμενο που εγκρίθηκε περιλάμβανε κάποια αντιφατικά στοιχεία. Γι' αυτό το λέω αυτό τώρα. Μάλιστα, θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα υπέρ κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία όμως, έτσι άρχιτη ψηφοφορία. Okay, we close the vote. The... Πέρας ψηφοφορίας υπερψηφίζεται. Η τροπολογία 5 εγκρίνεται 6R του εισηγητή. Ψηφίζουμε υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται η 6R. Οπότε καταπίπτει η 6. 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8. R του εισηγητή. Έτσι εάν εγκριθεί 8 και 9 καταπίπτουν. Υπέρ της 8R. Κατά. Κανείς. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 8 και οι 9. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική ψηφοφορία νομίζω θα χρειαστεί, διότι πολλοί δεν ψήφισαν καθόλου Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας η ψηφία ε, υπερψηφίζει εγκρίνεται λοιπόν τροπολογία 11 υπέρ κατά Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Άρχιτη ψηφοφορία. Can we close the vote? Πέρας ψηφοφορίας. Ε, Ορισμένε φορέ είναι δύσκολο έτσι να είμαστε βέβαιοι. Λοιπόν, υπερψηφίζεται εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ εντάξει δεν είναι σαφέστερα τα πράγματα κακά εκατά, εγκρίνεται συγγνώμη τροπολογία 13 υπέρ κατά εγκρίνεται η 13 14 υπέρ κατά εγκρίνεται 15 υπέρ κατά εγκρίνεται 16 υπέρ κατά εγκρίνεται 17 του εισηγητή 17R υπέρ κατά εγκρίνεται καταπίπτει 17 18 έως 22 από κοινού υπέρ κατά εγκρίνονται λοιπόν αυτές τις τροπολογίες 18 έως 22 και τώρα έχουμε μια νέα συμβαστική τροπολογία του εισηγητή ναι σας ακούμε Ναι, για αυτή την τροπολογία θα ήθελα να αναφερθώ στους που ανησυχούσαν ε, σε ό,τι αφορά το αρχικό κείμενο. Πρόκειται για το 36 και είναι έτοιμοι λόγω αυτού του σημείου να απορρίψουν το σύνολο της νομοδότησης. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε, όπως βλέπετε και στην οθόνη. Θα ήθελα να ακούσω όμως και εδώ ποια είναι ποιο είναι το πρόβλημά σας με αυτό το σημείο του κειμένου. Μιλάμε για το 36, έτσι. Εδώ είναι, μιλάμε για μια σύσταση Μιλάμε για την κοινωνική διάσταση, έτσι. Προωθούμε το, την πολιτική κληρονομιά της Ευρώπης, μιλάμε για την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα και πρέπει να υποστηρίξουμε την προστασία και το σεβασμό της ευρωπαϊκής θρησκευτικής κληρονομιάς και των κοινών αξιών με βάση το άρθρο 2 του Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επ' αυτού έχετε να μας πείτε κάτι. Εγώ είμαι ανοιχτός, όπως βλέπετε, σε συμβασμούς. Ναι, παρακαλώ, ο κύριος Αντρετσεύσκη και μετά η κυρία Καριολάινεν. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια εξαιρετικά ποιοτική γνωμοδότηση. Εδώ λέμε ότι οι Ευρώπη έχουν, ε, οι Ευρωπαίοι έχουν ρίζες χριστιανικές, ευρωχριστιανικές. Αυτή είναι η βάση στην οποία βασίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αντενάουερ, ο Σούμαν, ο Ντεγκάσπερι δημιούργησαν την Ευρώπη επ' αυτών των βάσεων. Και εμεί να το σεβαστούμε αυτό. Μόνο αν το σεβαστούμε αυτό θα μας σεβαστούν μετά και άλλοι. Βεβαίω, η θρησκευτική διαφορετικότητα και ποικιλομορφία είναι ένα στοιχείο ε, και αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης. Δεν είναι όμως αυτό το καλύτερο επιχείρημα κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι ε, από άλλες υπήρους που φτάνουν στην Ευρώπη. Εάν λοιπόν φτάνουν αυτοί με τη δική τους ταυτότητα πρέπει και εμείς να διαφυλάξουμε τη δική μας. Δεν μπορούν αυτοί να ενσωματωθούν σε κάτι που δεν υπάρχει στο κενό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε εμείς μια ταυτότητα για να ενταχθούν στη δική μα ταυτότητα. Λοιπόν, θα έλεγα να μην ακολουθήσουμε αυτή την οδό του να παρνηθούμε δηλαδή την ταυτότητά μας, να σεβαστούμε το παρελθόν μας. Η κυρία Κάρια Λάνεν έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καρατσόνη για την έκθεσή του, την νομοδότησή του. Μιλάμε τώρα για την τροπολογία 23, 24 και 25 όλες αφορούν ουσιαστικά το ίδιο σημείο και είχαμε συζήτηση από αυτού και στην Επιτροπή και σήμερα και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την τροπολογία αυτήν. Εμείς, η πολιτική μας ομάδα μπορεί να τη δεχτεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πλέον έχουμε μια διατύπωση η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Ο κύριος Κούπερ έχει το λόγο. Ναι, θυμάμαι η Τζο Κόξ, ε, η Αγγλίδα βουλευτής που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του Brexit, είχε πει ότι είναι πιο πολλά αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Και όταν μιλάμε για χριστιανοεβραϊκές αξίες εδώ δεν είναι σαν να μην βλέπουμε την κοινωνία στην οποία ζούμε μουσουλμάνοι, χριστιανοί, χριστιανοί εβραίοι όλες αυτές τις θρησκείες μιλούν για την ειρήνη, μιλούν για τη συνεργασία δεν θέλουν να μας χωρίσουν πρέπει λοιπόν να διαβάσουμε ε, να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές όταν βλέπουμε τροπολογίες που μιλούν για την κληρονομιά μας να δούμε πού μας οδηγεί αυτός ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος μας οδηγεί στην τρέλα και δεν μπορούμε να τον υποστηρίξουμε. Πρέπει να υποστηρίξουμε μια ενωμένη και μια Ευρώπη και μια Ευρώπη διαφορετικότητα στην οποία εγώ θα ήθελα να παραμείνω κιόλα. Ο κύριος Γκέσιγκ έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Øh, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Βλέπω τον συμβασμό που προτείνει ο εισηγητής και θεωρώ ότι είναι εύλογος συμβιβασμός και δείχνει τον σεβασμό μας απέναντι στις θρησκευτικέ πεπιθήσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει εκπρόσωπος από την Σλοβενία. Χαίρομαι που βρήκατε ε, με συμβαστική λύση είχαμε μια έντονη συζήτηση και πλέον υπάρχει μια συμβαστική λύση που αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκές αξίες που προωθούμε βασίζονται ε, και στην ποικιλομορφία και στην ακαιρεότητα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προωθήσουμε στο μέλλον η, η κουλτούρα μας ε, βασίζεται σε κάποια ιστορικά γεγονότα ε, όταν τονίζουμε ένα από αυτά πρέπει να τονίσουμε και τα υπόλοιπα Είναι δύσκολο να μπουν όλα αυτά σε μια διατύπωση. Εμεί πάντω θα υποστηρίξουμε αυτή την τροπολογία. Παρακαλώ, επόμενος ομιλητής. Ακούστε, στα πρακτικά αυτά ζητήματα πρέπει να προσπαθούμε να φτάσουμε στην, πραγματικ... στην αλήθεια. Ε, μιλήσαμε για την εκπαίδευση, για την παιδεία. Πώς όμως θα μεταφέρουμε στις μελλοντικέ γενιές αυτό το οποίο θέλουμε να του μεταφέρουμε. Θέλουμε να έχουμε ε, μια καλή σχέση με τους γείτονές μας, με τους αδερφούς μας, ε, με τους άλλους, ε, ακόμα και με αυτούς που πιστεύουν σε άλλα πράγματα. Μπορεί εμείς να έχουμε πανέμορφες πόλεις και καθεδρικούς ναούς. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή πρέπει να μπορούμε να ε, θαυμάζουμε την κληρονομιά μας και να αποδοχούμε και την διαφορετικότητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε με την ευκαιρία αυτή για ένα θέμα το οποίο κρίνεται από διάφορου τρόπου. Θέλω να ευχαριστήσω όμω εξ ονόματο τη ε, ομάδα μου, τον κύριο Καρατσόνη, για την τροπολογία που έχει καταθέσει. Η γνωμοδότησή του είναι σημαντική και άπλεται σημαντικών θεμάτων. Δεν είναι μια γνωμοδότηση ε, για, που αναφέρεται σε ιστορικέ φιλοσοφικέ αξιολογήσει. Αυτό το ξεκαθάρισε με την τροπολογία του. Και εμείς καλούμεθα να επικεντρωθούμε στα βασικά θέματα. Αυτό το συζητήσαμε σήμερα το πρωί στην πολιτική μας ομάδα και μάλιστα σε βάθος. Νομίζω ότι πρόκειται για μια πορεία συνεργασίας αυτή που επιλέγει ο κ. Καραζόνη και αυτό τον ευχαριστώ ρητά. Ορίστε κύριε Καραζόνη, εσείς και μετά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Όσον αφορά την, ε, ε, το, ε, τον συμβιβασμό επετέφθη την τελευταία στιγμή έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και μια ενωτική γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειών. Πριν δεκτώ τον προφορικό συμβιβασμό θα ήθελα να αναφέρω τα λόγια του Αντώνιο Ταγιάννη, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή η κληρονομιά, η οδεοχριστιανική, είναι <clears throat> πάρα πολύ σημαντική. Στο Στοκόλμη, στη Μάλτα, στο Ελσίνκι, στη Ρώμη, στο Βερολίνο. Ο Σταυρός είναι ε, η ε, διασύνδεση. Ε, έχουμε κοινή κληρονομιά και κοινή ταυτότητα ο, η κληρονομιά μας δεν είναι να είμαστε ο ένας εναντίον του άλλου αλλά πρέπει να ξέρουμε και ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Okay, uh, now we go to the vote. The rapporteur's amendment uh, covers these 23, 24, 25 and that's the compromise that we have seen on the screen. Those in favor of that vote now. Against. Ε, Εγκρίνεται. Επομένως, οι τροπολογίες 23, 24 και 25 καταπίπτουν. Ε, ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε επί του συνόλου της τραποποιημένης γνωμοδότησης υπέρ. Σας ευχαριστώ. Ψήφι κατά. Αποχές, δύο αποχές, καμία ψήφος εναντίον. Επομένως η πλειοψηφία ε, υπερψήφισε και επομένως εγκρίνεται η έκθεση και συγχαίρω τον εισηγητή. Now, next. Περνούμε τώρα στην επόμενη γνωμοδότηση της ε, κυρίας Ουλρίκε Χίλερ. Κυρία Χίλερ, παρακαλώ, ελάτε εδώ μαζί μας. Eh?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 Ωραία λοιπόν είναι ενδιαφέρον το ε, αντικείμενό σας είναι ο Ερασμός έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα αυτό με τον Επίτροπο κ. Ναύρατιτς τώρα η κυρία Χίλερ θα κάνει τη σχετική ε, εισαγωγή στην ε, γνωμοδότησή της παρακαλούμε το μικρόφωνο της ομιλητρίας σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα είμαι σύντομη διότι ο χρόνος αρχίζει και πιέζει κάπως. Ε, θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου γιατί ήταν και μεγάλη τιμή για μένα που μου αναθέσατε την σύνταξη της γνωμοδοτήσεως κάτι βεβαίω το οποίο ποτέ δεν μπορεί να φέρει εις πέρας μόνος του ή μόνη της πολλοί με βοήθησαν από το γραφείο της ΣΥΝΤΕΚ από τα άλλα επίσης αλλά και από την δική μου ομάδα και βεβαίως και ο εμπειρογνώμων μου που ε, κάθεται δίπλα μου. Όλα τα πρόσωπα αυτά έκαναν μεγάλη προσπάθεια, όπως και εσείς βεβαίως, με τις τροπολογίες που καταθέσατε και που εν μέρει είναι σημαντικές συμπληρώσεις και τις οποίες σας ευχαριστώ. Μιλήσαμε και σήμερα για τον έρασμο. Πρόκειται τώρα για το πρόγραμμα που διαδέχεται το πρώτο πρόγραμμα και θα ισχύει από το 2021 έως 2027 και έχει κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διεξήχθησαν διάφορες ακροάσεις και στις Βρυξέλλες αλλά και στην Βρέμη, την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Έχουμε λάβει πολλές άλλες παρεμβάσεις, έχουμε ανταλλάξει εμπειρίες με εμπειρογνώμονες οι οποίοι εργάζονται στο πρακτικό πεδίο. Προσπαθήσαμε να τα περιλάβουμε όλα αυτά στη γνωμοδότηση και τώρα έχετε μπροστά σας το αποτέλεσμα. Ο έρασμος ε, είναι, έχει τρία σημαντικά σημεία. Δεν υπάρχουν σύνορα στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό. Και αυτό είναι σωστό. Πρέπει να ε, καταργηθεί κάθε σύνορο που ε, αποτελεί εμπόδιο για την εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Εκεί χρειάζεται να υποστηρίξουμε τις αξίες μας, είτε πρόκειται για την αλληλεγγύη είτε πρόκειται για τον ανθρωπισμό. Αυτό που πρέπει να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο πριν είναι οι αξίες αυτές τις οποίες ε, διαδίδουμε και με το πρόγραμμα Έρασμος. Ε, η, παιδεία θα πρέπει να είναι κοινό αγαθό. Όλοι θα πρέπει να, πρέπει να, έχουν, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ανεξαρτήτως οικογενειακού, ε, ιστορικού κλπ. Τώρα, για τα πιο σημαντικά σημεία της γνωμοδοτήσεως. Ήδη τα είπα αυτά το πρωί. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο εμφανίστηκε κατ' επανάληψη στις διαβουλεύσεις που διεξαγάγαμε είναι μεταξύ των σπουδαστών αλλά και των πρόσωπων που ε, ακολουθούν μια κατάρτιση χρειαζόμαστε για όλους αυτούς επιχειρήσεις που να τους ε, λάβουν στις τάξεις τους και επομένως θέλουν όλο και οι περισσότερες, και περισσότερες επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή ήδη και μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και μικρές επιχειρήσεις, όχι μόνο αυτές που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Με κάποιο τρόπο πρέπει να τις προσελκύσουμε. Εμείς προτείνουμε μεγαλύτερη συμμετοχή της ιδιωτικής οικονομίας, ιδίως στον τουρισμό και στην κινητικότητα, διότι μας διακατέχει η ανησυχία ότι άλλος πολλά χρήματα που διατίθεται για τον έρασμο θα εισρεύσουν ε, προς τα εκεί, αλλά δεν θα δοθούν αρκετές δυνατότητες σε πολλούς 18χρονους ε, να ε, εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα. Τώρα για τον αθλητισμό, κυρίως μας ενδιαφέρει να ανοίξουν οι δυνατότητες ώστε και μικρές αθλητικές εκδηλώσεις να μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα έρασμο. Και γι' αυτό είναι σημαντικό για μας αυτό το όριο που υπάρχει, το ότι πρέπει να είναι κατελάχιστον 10 χώρε μέλη, να καταργηθεί. Να είναι δυνατόν δηλαδή και με, λιγότε, και με συμμετοχή λιγότερων χωρών μελών να γίνονται τέτοιε ευρωπαϊκέ αθλητικέ εκδηλώσει που να χρηματοδοτούνται από τον Εράσμο. Για τα δίκτυα των σχολών, αυτό μα ικανοποιεί πολύ. Ήδη γίνονται πολλά πράγματα, αλλά δεν θα πρέπει να περιοριστούν στι πρωτεύουσε, θα πρέπει να ενισχυθεί και η περιφερειακή διάσταση και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή για την οποία είμαστε εμείς αρμόδιες και αρμόδιοι στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι αναγκαίο να υπάρξει εντονότερη διαβούλευση η οποία να λάβει υπόψη και να μπορεί και να εκπροσωπήσει το τοπικό επίπεδο και να συνεργάζεται και με τους εθνικούς θεσμούς. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία νομίζω. Ε, αν θέλετε τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα όντως στις ψηφοφορίες. Στην πράξη έχουμε πολλές προτάσεις. Η συγκίτρια έχει και δικές της τροπολογίες, αλλά είναι και υπέρ όλων των υπολείπων εκτός από μία. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν σύντομα. Λοιπόν, 1. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά, εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 3. Ρο. Υπέρ κατά εγκρίνεται 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 6 ρο της εισηγήτριας δηλαδή υπέρ κατά εγκρίνεται 7 Α, 7, 8 εκπίπτουν. 9 έχει αποσυρθεί. 10 ρο της συγητρίας υπέρ κατά εγκρίνεται η 10 εκπίπτει 11 υπέρ κατά εγκρίνεται 12 ρο υπέρ κατά εγκρίνεται 12, 13, 14 εκπίπτουν 15 έως 22 όλες μαζί Ψηφίστε υπέρ. Κατά εγκρίνονται 23. Τροπολογία της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Κάνει εγκρίνεται. 23 εκπίπτει. 24 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. τη εισηγήτριας 26 ρο υπέρ κατά εγκρίνεται 27 υπέρ κατά εγκρίνεται της εισηγήτριας 28 ρο υπέρ κατά εγκρίνεται προχωρώ στην 29 υπέρ κατά εγκρίνεται 30 ρο της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται 30-31 εκπίπτουν 32 υπέρ κατά εγκρίνεται 33 υπέρ κατά εγκρίνεται 34 ρο της ηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται ακολουθεί 36 ορό της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται 37 υπέρ κατά εγκρίνεται 38 υπέρ κατά εγκρίνεται 39 ρο υπέρ κατά εγκρίνεται 40 υπέρ κατά εγκρίνεται 49 η εισηγήτρια είναι κατά ψήφι υπέρ ουδής κατά η πλειοψηφία λοιπόν είναι κατά απορρίπτεται 42 υπέρ κατά εγκρίνεται 43 ρο υπέρ κατά εγκρίνεται 44 υπέρ κατά εγκρίνεται 45 ρο της ηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται το σύνολο της νομοδοτήσεως τώρα ας ψηφίσουμε σας ευχαριστώ πολύ κατά κανείς αποχές κανείς άρα ομόφωνη υποστήριξη. Είμαστε όλοι υπέρ του έρασμου. Ωραία, έχουμε ακόμα τέσσερις γραμμοδοτήσεις. Μπριγίτε Σακρεντέους, παρακαλώ, έλα. Where do we have Birgit? Ah, η Μπιργκίτε είναι εδώ, έρχεται. On this as introduction. So good Είχαμε, έγινε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μελών ε, διαφόρων και της ε, εισηγητρίας και επομένως έχουμε κάποιες προτάσεις ε, από πλευράς της εισηγητρίας και μάλλον μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα αλλά βέβαια πρώτα να μας κάνει μια εισαγωγή η Μπυργίτε Σακρεντέους και θα της δώσω αμέσως λοιπόν το λόγο. Καλό είναι να ανοίξεις το μικρόφωνο πάντως πριν μιλήσεις Μπριγκίτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι τόσο αργά ε, και αναφέρομαι βέβαια σε όλους όσοι είναι ακόμα παρόντες για να ακούσετε για ένα θέμα το οποίο μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Ε, όλοι μπορούμε ε, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας και η έρευνα και η καινοτομία βεβαίως είναι κάποια, κάποιοι θετικοί τρόποι της κοινωνίας στο νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία ε, προσφέρονται πολλές ε, δυνατότητες σε όσους εργάζονται ε, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Πλέον σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο υπάρχουν τρόποι δράσης για την πρόθεση της κοινωνίας. Εδώ δεν αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε κάποια περιφέρεια. Εδώ γίνεται λόγος για την κοινωνία στο σύνολό της. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να καταδείξω την μία ή την άλλη περιφέρεια. Εγώ πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε και οφείλουμε να δημιουργήσουμε, να οικοδομήσουμε ε, την, μια βιώσιμη κοινωνία, ε, μια κοινωνία ε, η οποία θα περιέχει όλα τα στοιχεία της προστασίας του περιβάλλοντος ε, ε, και προστασία της κοινωνίας γενικότερα. Μπορούμε να, πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα έτσι ώστε να βελτιωθεί και η ίδια η έρευνα και να προκύψει καινοτομία αυτό που μας λέει η Κομισιόν είναι ότι πρέπει να εξευρεθούν συνέργειες, δηλαδή τα διάφορα προγράμματα, ε, τα διάφορα, οι διάφοροι πόροι, τα διάφορα ταμεία ε, θα πρέπει να συνενωθούν έτσι ώστε να προκύψουν ε, όσο γίνεται μεγαλύτερες συνέργειες και έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο. Η έρευνα και η καινοτομία είναι σημαντικές για την οικονομία φυσικά, αλλά όχι μόνον. Η έρευνα και η καινοτομία είναι σημαντικές για την κοινωνία των πολιτών, για, τις, ε, ε, για τα ε, πανεπιστήμια. Και αυτό είναι ένα ταξίδι το οποίο θα ξεκινήσουμε μαζί με την Κομισιόν. Θα αναρωτιέστε ίσως γιατί εγώ θα δείτε το όνομά μου μεταξύ των ε, ε, συναδέλφων που έχουν υποβάλει τροπολογίες. Θέλαμε να ε, έχουμε τους ίδιους ορισμούς. Γι' αυτό έχω προσυπογράψει πολλές τροπολογίες. Γιατί είναι αρκετοί αυτοί που έχουν υποβάλει τροπολογίες για τους ορισμούς. Είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρες οι έννοιες. Ε, τροπολογία 23. Στην τροπολογία 23 ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός λεπτομέρειας. Γι' αυτό λοιπόν θα σας ζητούσα να μην υπερψηφίσετε την τροπολογία αυτή. Αντιθέτως, όσον αφορά την τροπολογία 26, θα θέλαμε να, ε, το, να την προσυπογράψουμε όπως και τα σημεία 32, 33 και 36 Ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσίασή σας και για την εργασία που κάνατε. Ο κύριος Μακάρτιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτήν την ε, γνωμοδότηση γιατί πραγματικά η έρευνα, η καινοτομία μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένε βελτιώσεις, σε προστασία των οικοσυστημάτων, περιβάλλοντος κτλ. Πολλά συζητήθηκαν ε, κατά τη διάρκεια της ε, ε, συζήτησης αυτής και κυρίως το θέμα που αφορά το GRC, το κοινό κέντρο ερευνών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης θέματα όπως είναι η μεταφορά ενέργειας, ε, οι πλατφόρμες ανταλλαγής ε, στοιχείων και καινοτομιών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και χαίρομαι που έχουν συμπεριληφθεί. Επίσης, ε, Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο και τα προγράμματα ε, Interreg έτσι ώστε να, ε, να ξαναδούμε επίσης ε, και τα προγράμματα δράσης, τη δυναμική τους έτσι ώστε να δημιουργηθούν αυτές οι συνέργειες. Θα πρέπει να πω επίσης ότι το είχαμε πρόσφατα την απονομή του ε, βραβείου ε, Icap ε, και λυπήθηκα που δεν μπορέσαμε να έχουμε πραγματικά τους ανθρώπους που θα θέλαμε να το έχουν κερδίσει. Εν πάση περιπτώσει Um, να περάσουμε λοιπόν τώρα στην στις ε, τροπολογίες Ένα, δύο, τρία να ψηφιστούν από κοινού υπέρ, κατά εγκρίνονται τροπολογία 4 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά εγκρίνεται Άρα καταπίπτει η 6. Ε, τροπολογία από κοινού για τις τροπο... Ε, ψηφοφορία από κοινού για την 7, ε, 8 και 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά εγκρίνεται Τροπο, ψηφίζουμε από κοινού 12, 13, 14 υπέρ κατά εγκρίνονται. Έχουμε συμβιβασμό για τη 15 Κυρία εισηγήτρια, θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό. Έχετε διαγράψει κάποιες ε, από τις ε, ε, λέξεις, τέλος πάντων κάποια στοιχεία της διατύπωσης. Ναι, όντως λέει η εισηγήτρια. Στην τροπολογία γίνεται πρόταση να γίνει μείωση ανισοτήτων ε, κτλ. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να προκύψουν συνέργειες. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Η είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι θα πρέπει να ελέγξουμε η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν επί της τροπολογίας 16. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 16. Από κοινού ψηφίζουν την τροπολογία 17 έως 22. Να ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Τροπολογία 23. Η εισηγήτρια είναι κατά, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 23. Πέρας της ψηφοφορίας ε, ε, καταψηφίστηκε η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται τροπολογία 25 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται η συγκήτρια. Έχει υποβάλει τροπολογία 26R υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Επομένως, τροπολογίες 26, 32, 33, 36 καταπίπτουν. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Από κοινού 29 μέχρι 31 ψηφίζουμε υπέρ κατά εγκρίνονται. Τροπολογία 32, ο μάλλον η 32 έχει καταπέσει και η 33 ψηφίζουμε από κοινού για τις τροπολογίες 34 και 35 υπέρ κατά εγκρίνονται Τροπολογία 37. Ψηφίζουμε την 37 υπέρ κατά καμία ψήφος κατά εγκρίνεται λοιπόν η τροπολογία αυτή. Ψηφίζουμε τώρα την τροποποιημένη γνωμοδότηση υπέρ κατά Κανείς δεν ψηφίζει κατά, κανείς δεν απέχει και επομένως εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια κυρία Σακρεντέους για τη γνωμοδότησή σας. Right, do we have Jan Λοιπόν, είναι εδώ ο Γιάνν Τρέι, παρακαλώ. Ελάτε και μετά από αυτή την νομοδότηση μας μένουν ακόμα δύο. Όλγιαρτ Γκεμπλέβιτς και Γιώζεφ Ρίμπανη. Την επόμενη φορά πρέπει θα ζητήσω ο εισηγητής ήδη να έρχεται όταν ψηφίζουμε για την προηγούμενη τροπολογία. Έτσι να επιταχύνουμε, να κερδίζουμε και λίγο χρόνο να προλάβει και να φάει όποιος θέλει να φάει να κάνει τίποτε άλλο όπως το βράδυ, όπως περιπτώσει. Γιάν Τρέι. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Εδώ έχουμε μια γνωμοδότηση πρωτοβουλία της Επιτροπή των Περιφερειών που αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη. Με βοήθησε ο εμπειρογνώμονα μου ο κύριος Σέλ από την, ε, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Ταλίν ε, είναι και επικεφαλής του project για το πρώτο ε, λεωφορείο χωρίς οδηγό στο Ταλίν είναι προφανές ότι η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει ριζικά το πώς ε, είναι ο κόσμος που ζούμε Καλό είναι λοιπόν να υπάρχει μια χρωμάτωση πρωτοβουλία ε, από την πλευρά μα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλωστε έχει ασχοληθεί με το θέμα. Εμείς ως περιφέρειες και τοπικές αρχές θέλουμε να τονίσουμε ποιες είναι οι δυνατότητες και στο δικό μας επίπεδο σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό από το από πλευρά ε, τοπικών αρχών και τοπικών, τοπικής παροχής υπηρεσιών. Ε, μεταφορά χωρίς οδηγό, ε, έξυπνες πόλεις, αυτοματοποιημένες λύσεις ε, και το πώς αυτό συνδέεται με το κράτος πρόνοιας, τις, τις ε, υπηρεσίες περίθαλψης και υγείας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στον τομέα της παιδείας ε, αλγόριθμοι παραδείγματος χάρη ε, που ε, εγγράφουν τα παιδιά στα σχολεία ανάλογα με το που μένουν Ποια είναι τώρα τα κεντρικά μηνύματα αυτής της νομοδότησης Επανακατάρτιση είναι προφανές ότι η τεχνητή νοημοσύνη ε, στο άμεσο μέλλον θα αντικαταστήσει μια σειρά από θέσει απασχόληση. Δηλαδή θα χαθούν θέσει απασχόληση. Θα δημιουργηθούν όμω άλλε. Και αυτό σημαίνει ότι αυτές οι νέες εργασίες ε, για να, οι θέσεις εργασίας για να μπορέσουν να πληρωθούν θα χρειαστούν επανακατάρτιση, εκπαίδευση και εδώ οι περιφέρειες έχουν ένα ρόλο να παίξουν. Πρέπει εδώ να είμαστε ευέλικτοι ε, σε επίπεδο χρηματοδότησης ε, στον τομέα της εκπαίδευσης να απομακρυνθούμε ε, σε μια προσέγγιση που βασίζεται σε αυτή διάφορα project θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο μακριά στο μέλλον και θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι σημαντικό να υπάρξει και ένα συντονισμό των στρατηγικών για την τεχνητή νοημοσύνη ε, στι εθνικέ στρατηγικέ των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμεί έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εργασία στην Εσθονία για την τεχνητή νοημοσύνη και προσπαθούμε να συντονίσουμε το τι κάνουμε εμείς με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές. Είναι σημαντικό να υπάρξουν πιλωτικά προγράμματα σε τοπικό επίπεδο για μια σειρά από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Να μην αφήσουμε τις τοπικές αρχές δηλαδή ε, απ' έξω από αυτήν την προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσεχές μέλλον θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδότηση για τέτοιου είδου project τεχνητής νοημοσύνης και γιατί όχι να προβλέψουμε ένα μέρος της χρηματοδότησης ε, για αυτό το ζήτημα στο άμεσο μέλλον. Επενδύουμε τρεις φορές λιγότερο ε, από τους Κινέζους στον τομέα αυτόν. Τέσσερις φορές, λιγότερο από τους Αμερικανούς. Ε, έχουμε μείνει πίσω. Εγώ υποστηρίζω την ιδέα να δημιουργήσουμε μια σφαιρική πλατφόρμα για την τεχνητή νοημοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συμμετοχή και εκπροσώπων από τις περιφέρειες και φορέων τοπικών που θα μπορέσουν και αυτοί να συνεισφέρουν από το δικό τους πρίσμα, από τη δική τους οπτική γωνιά. Και βεβαίως χρειάζεται και ένα νομικό πλαίσιο πρέπει να πλαισιώσουμε νομικά την τεχνητή νοημοσύνη και γιατί μπαίνουν και ζητήματα ηθικής, θα πρέπει όλα αυτά να συνάδουν με τη χάρτη θεμελιών δικαιωμάτων ε, και βεβαίως υπάρχει το θέμα της ασφάλειας το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε καθώς και της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας της. Όσο πλησιάζουμε προς ψηφιακές λύσεις, τόσο πιο ευάλωτες, ε, αυτά τα στοιχεία τη ιδιωτική ζωή και τη ταυτότητά μα τελικά. Η εφαρμογή τη τεχνητή νοημοσύνης στην Ευρώπη ε, πρέπει να περιλαμβάνει και τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Υπάρχουν συνεισφορέ. Όχι. Θα ακούσουμε περισσότερο για τεχνητή νοημοσύνη όταν έρθει και η Φιλανδική Προεδρία. Λοιπόν, πρώτα θα ψηφίσουμε από κοινού τις τροπολογίες 1 έως 5. Παρακαλώ, υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Πολύ ωραία, εγκρίνονται. Τροπολογία 6, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Διότι πολλοί δεν ψηφίζουν, κάποιοι μάλλον είναι για καφέ. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά παρακαλώ. All right, let's close the vote. Πέρας ψηφοφορίας υπερψηφίζεται αυτή η τροπολογία. Τώρα από κοινού 7 έως 9 ψηφίζουμε υπέρ κατά εγκρίνονται αυτές τις τροπολογίες και τώρα το σύνολο της νομοδότησης υπέρ κατά αποχές πολύ ωραία ομόφωνα λοιπόν εγκρίνεται η νομοδότηση συγχαρητήρια κύριε Τρέι Ma sooviksin veel tänada eh, Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλη την ομάδα που με βοήθησε, τον εμπειρογνώμονά μου. που συνέβαλαν στην επιτυχή κατάληξη αυτής της νομοδότησης να πω και δύο λόγια έτσι διαφημιστικά αν θέλετε η Εστονία προωθεί ψηφιακές λύσεις όπως ξέρετε και αυτή τη στιγμή και στις Βρυξέλλες ε, υπάρχει ένα λεωφορείο χωρίς οδηγό που προέρχεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Εσθονίας, το Ταλίν και μπορείτε να το δείτε αύριο στην αντιπροσωπεία μας. Ελάτε να το δείτε. right. Uh, Πολύ ωραία. Η επόμενη γνωμοδότηση τώρα, Όλγερ Γκέμπλεβιτς, αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Να δώσω τον λόγο ευθύς αμέσως ε, για την εισαγωγή. Okay. you, Mr. Ε, Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Αυτή η ιστορία της παραπληροφόρησης μας απασχολεί εδώ και από, πολύ, από πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα με την εξέλιξη του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων η παραπληροφόρηση έχει γίνει τελικά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος που απειλεί την σύγχρονη δημοκρατία. Πολλοί ανεξάρτητοι θεσμοί έχουν επιληφθεί του θέματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλωστε πέρσι τοποθετήθηκε σχετικά διότι αντιλαμβανόμαστε πλέον όλοι ότι τίθεται σε κίνδυνο οι ελεύθερες εκλογές. Δημοσίευσε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς ως Επιτροπή Περιφερειών προβαίνουμε σε γνωμοδότηση διότι η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης είναι κοινό καθήκον όλων μας. Στη γνωμοδότησή μου περιλαμβάνω πολλά παραδείγματα. Παραδείγματα εκστρατιών παραπληροφόρησης. Αναγράφω επίσης ότι υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις στις οποίες εμείς οι ίδιοι δημοσιεύουμε εσφαλμένες πληροφορίες. Έχει διαπιστωθεί από μελέτε ότι μια ψευδής πληροφορία έχει 70% περισσότερες πιθανότητες να διαδοθεί από μια αληθή πληροφορία. Άρα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα των εκλογών. Από την άλλη μεριά χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια υπεύθυνη κοινωνία. Για να μπορέσει να γίνει αυτό χρειάζεται λήψη μέτρων σε πολλά επίπεδα. Στην δε γνωμοδότησή μου εγώ υποστηρίζω τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν τέσσερα ουσιώδη στοιχεία για την καταπολέμηση παραπληροφόρηση. Πρώτον, περισσότερη διαφάνεια σχετικά με τις πηγές των ψευδών πληροφοριών. Θα πρέπει δηλαδή να είναι γνωστό ποιος δημοσιεύει τις ε, παραπληροφορίες, ποιος χρηματοδοτεί την δημοσίευση αυτή. Επίσης πρέπει να υπάρξει έλεγχος της παραπληροφόρησης. Σημαντικό αυτό. Και χρειαζόμαστε και προγράμματα κατάρτισης για να έχουμε έτσι ενσυνείδητους πολίτες. Όσο γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έλθει σε συμφωνία με τις ε, πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και έχει αναπτύξει και σχέδιο ε, δράσης για τα επόμενα χρόνια. Ως εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Περιφερειών θέλουμε και εμείς την ευθύνη να αγωνιστούμε κατά της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων. Πρώτα, θεωρούμε ότι η παιδεία παίζει ρόλο κλειδί για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Οι τοπικές αυτοδιοίκησεις είναι αρμόδιες για την παιδεία. Για το λόγο αυτό πρέπει ε, να αναλάβουμε ευθύνες, τις ευθύνες μας για τη δημιουργία ενός συνειδητού πολίτη, ο οποίος δεν θα πέφτει στις παγίδες που του στείνει η παραπληροφόρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή. Δεν πρόκειται μόνο για τη δημιουργία της κοινωνίας τις πληροφορίες όπως λένε κυρίως αυτό που μας απασχολεί είναι η συνειδητοποίηση για τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και αυτό αποτελεί καθήκον πολλών οργανώσεων και όχι μόνο των μη κρατικών οργανώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων που καταπολεμούν την παραπληροφόρηση. Είναι σημαντικοί οι οργανισμοί αυτοί, οργανώσει μάλλον αυτέ, και χρειάζονται υποστήριξη. Χρειαζόμαστε επίση υποστήριξη για τοπικούς ε, στόχους τοπικής εμβέλειας δηλαδή και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Εδώ πρέπει να παίξουμε ένα ρόλο εμείς γιατί βλέπουμε ότι βρίσκονται πλέον σε φάση άμυνας ε, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης τα οποία, ε, τα οποία δρούν υπεύθυνα, δεν δημοσιεύουν ανώνυμα άρθρα. Άρα πρέπει να υποστηρίξουμε τα μέσα αυτά ενημέρωση, ώστε να επιτύχουμε στα αυτιά των πολιτών να φτάνουν υπεύθυνε πληροφορίε. Θέλω να ευχαριστώ πολύ τον εμπειρογνώμονά μου κύριο Μπίλεβιτ, καθώς και, και όλα τα πρόσωπα εκείνα που έχουν συντάξει τροπολογίες. Προσπάθησα να τις λάβω υπόψη όλες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την θαυμάσια ε, εισαγωγή σας. Α, κύριε Αρμάου δεν επιθυμείτε να κάνετε παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή η πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί ακριβώς ε, προωθεί την πολιτική κοινωνία προς ε, την κοινωνία της τεχνολογίας. Θα ήθελα ε, να πω δύο λόγια όσον αφορά τις τροπολογίες μου σχετικά με την ανοιχτή διακυβέρνηση. Εάν καταφέρουμε να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα των τοπικών αρχών στην, ε, στις πληροφορίες γενικά θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτά τα fake news, οι ψευδείς ειδήσει ε, φτάνουν ε, μέχρι όλους αλλά και πολύ γρήγορα και μάλιστα δεν διαφέρουν στην ουσία από τα, τις κανονικές ειδήσει. Γι' αυτό λοιπόν τοπική περιφερειακή διοίκηση θα έπρεπε έπρεπε να έχουν ανοιχτά στοιχεία έτσι ώστε ε, ένας πολίτης ο οποίος αμφιβάλλει για μία είδηση να μπορεί να την ελέγξει. Ναι, γιατί ξέρετε ε, μπορεί ας πούμε να ε, του λένε για ένα στοιχείο και αν έχει αμφιβολία να μπορεί να το ελέγξει στο site ας πούμε της ε, τοπικής ή περιφερειακής διοίκησης. Λέω ότι η καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων περνάει και μέσα από το Open Government, από την εύκολη ανοιχτή προσβασιμότητα που δίνει την δυνατότητα στον πολίτη να ε, επιβεβαιώσει αν πρόκειται για ψευδή είδηση, για fake news. Ευχαριστώ. Στο Παλέρμο ε, στην ε, Σικελία θα έχουμε και μία συνεδρίαση του ΣΕΝΤΕΚ για την ψηφιοποίηση. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τον λόγο. Ε, είμαι από την Δανία, Περιφερειακός Σύμβουλος. Δεν συμφωνώ με αυτήν την ε, πρόταση και όχι γιατί δεν έχει δουλέψει καλά ο εισηγητής, ε, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να δοθούν χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου από πλευράς Κομισιόν για τέτοια πράγματα τα οποία είναι αρκετά ασαφή. Απ' την άλλη πλευρά δεν θέλουμε κανένα περιορισμό όσον αφορά την ελευθεροτυπία, τη δυνατότητα έκφρασης. Δεν λέω ότι δεν είναι πρόβλημα η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση. Θα συμφωνήσω πάντως με τον προηγούμενο ομιλητή ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτή διακυβέρνηση και βεβαίως την αντίστοιχη παιδεία, συμπληρώνω εγώ, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε και να, υπερασπι... να προασπιζόμαστε τους εαυτούς μας από τα fake news. Όταν εφευρέθη ε, ε, το ραδιόφωνο φοβόταν ο κόσμος για τον τρόπο με τον οποίο ε, θα επηρεάσει την κοινωνία. Η ευρωπαϊκή κοινωνία όμως είναι πιο έξυπνη από ό,τι νομίζετε. Γι' αυτό να μην δαπανούμε χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου για τέτοια πράγματα Ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος, δεν ε, έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Προχωράμε λοιπόν στην τροπολογία. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία αρ. Τροπολογία του εισηγητού υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επομένως καταπίπτει 2, τροπολογία 3 υπέρ κατά. Εγκρίνεται 4 υπέρ κατά. Εγκρίνεται 5 υπέρ κατά. Υπερψηφι... Α, απορρίφθηκε. Ε, τροπολογία 6 κατά απερίφθη τροπολογία 7 υπέρ κατά υπερψηφίστηκε εγκρίνεται λοιπόν τροπολογία 8 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά εγκρίνεται 11 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 13 άρα του εισηγητού υπέρ κατά εγκρίνεται. Εγκρι... Ε, καταπίπτει 13, τροπολογία 14 άρτου εισηγητού υπέρ, κατά. Εγκρίνεται, καταπίπτει λοιπόν η 14, τροπολογία 15 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται, τροπολογία 16 άρτου εισηγητού υπέρ, κατά. Εγκρίνεται επομένως καταπίπτουν οι 16 και 17, τροπολογία 18 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία του εισηγητού υπαριθμών 19R υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και επομένως καταπίπτουν οι τροπολογίες 19 και 20. Τροπολογία 21R του εισηγητού υπέρ κατά εγκρίνεται καταπίπτουν οι 21, 22, 23 και 24 δεν έχουμε άλλες τροπολογίες ψηφίζουμε λοιπόν επί του συνόλου της τροποποιημένης γνωμοδότησης υπέρ κατά μία ψήφος κατά δύο αποχές καμία αποχή εγκρίνεται έτσι όπως την τροποποιήσαμε. Λοιπόν, την εγκρίναμε την γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα περνάμε στην τελευταία γνωμοδότηση για απόψε. Γιώζεφ Ριμπάνη. Οδική ασφάλεια και αυτοματοποιημένη κινητικότητα.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 Ωραία λοιπόν για τη γνωμοδότηση αυτή έχουμε μια προφορική συμβαστική τροπολογία και κάποιες αλλαγές που θα τις δούμε όμως όταν θα προχωρήσουμε. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στον εισηγητή μας κύριο Ριμπάνη. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Η παρούσα γνωμοδότηση χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο είναι η επανεξέταση της οδηγίας 2018, μετά αναφέρεται στη στρατηγική και το τρίτο είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κινητικότητα. Για την αναθεώρηση τώρα της οδηγίας κατατέθηκαν 17 τροπολογίες, 19 μάλλον τροπολογίες, 19. Το πιο σημαντικό είναι πάντως να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας είναι προφανές ότι χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών και μετά να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί, να τονιστεί ο ρόλος των ε, ε, δικτύων TNT, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Σε ορισμένες περιφερειές μπορούμε να αναπτύξουμε τέτοια δίκτυα μεταφορών. Αλλά αυτό χρειάζεται τα αναγκαία κονδύλια για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Εγώ με ικανοποίηση πάντως είδα ότι μπορέσαμε να αποφασίσουμε και βασικές οδούς θα ακολουθήσουμε για την τοπική και περιφερειακή συνεργασία. Σε ορισμένες ε, περιφέρειες έχουμε ήδη πρωταρχικούς, ε, πρωταρχικής σημασίας δρόμους, αλλά σε άλλες όχι. αυτοκινητοδρόμους ας πούμε. Και αυτά, αυτοί οι αυτοκινητοδρόμοι μπορούν να βοηθήσουν τις περιφερειές να αναπτυχθούν πολύ ταχύτερα. Αυτό που χρειάζεται βέβαια είναι να κάνουμε και αξιολόγηση των οδικών αρτηριών και να έχουμε και επαρκή χρόνο για να γίνει η αξιολόγηση αυτή. Χρειαζόμαστε επίσης θέσπιση σαφών κανόνων σε αυτή την πολυσχηδή και πολυφωνική Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για την στρατηγική της αυτο, αυτοματοποιημένης κινητικότητας. Αυτό βέβαια συγκίνησε πολλούς, είδα και τις τροπολογίες. Πάντως, για, την, ε, για το μέλλον ανοίγεται μια μεγάλη ε, ευκαιρία και ιδίως για αεροκατοικημένες περιοχές, διότι σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μεταφορές αυτού του είδους για να προσεγγίσουν πιο εύκολα αστικά κέντρα και να διεκπαιρεώσουν υποθέσεις τους. Υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό της ε, κινητικότητας. Η κινητικότητα δηλαδή θα γίνει εν τέλει παροχή υπηρεσίας. Και αυτό θα αλλάξει όλη την φύση της κυριότητας των αυτοκινήτων. Της ιδιοκτησίας αυτοκινήτων δηλαδή και θα σημαίνει ότι θα απαλλαγούν από την κυκλοφορία αυτοκινήτων καθώς και από πάρκινγκ κλπ σημαντικά τμήματα των αστικών κέντρων μας. Εμείς χρειάζεται να εναρμονίσουμε βέβαια τα δίκτυα των οχημάτων που θα κινούνται με αυτόματο τρόπο αλλά ως τοπικές αυτοδιοίκησεις είναι σημαντικό για μας ε, να ξεκινήσουμε τεστ, δοκιμασίες, καθώς και πιλωτικές διαδρομές για να μπορέσει η κινητικότητα να γίνει πιο αποτελεσματική και επομένως και λιγότερο δαπανήρη, πιο φτηνή. Πιο φτηνή κινητικότητα σημαίνει βέβαια ότι θα αυξηθεί η κυκλοφορία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την αύξηση. μέσα στα αστικά κέντρα πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε και να προετοιμάζουμε την αντιμετώπιση των διαφορών προκλήσεων. Χρειαζόμαστε ευφύ οχήματα που να κινούνται μέσα στα αστικά κέντρα. Ενώ στην Ήπεθρο μας χρειάζονται ευφυείς δρόμοι. Να δούμε τώρα και τον τρίτο πυλώνα του εγγράφου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κίνηση. Ευρωενώ δηλαδή την ανακοίνωση της Επιτροπής. και με ορίζοντα το 2050. Βλέπουμε να δημιουργείται, το ενδεχόμενο να δημιουργείται ηλεκτρονικό σμόγ στις πόλεις και δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την αντιμετώπιση του. Δεν γνωρίζουμε ποιε θα είναι οι συνέπειε στην υγεία των ανθρώπων, για παράδειγμα. για τις ευφυείς μεταφορές αυτές σημαίνουν και μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Με την χρήση δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εναλλακτικές πηγές ενέργειας και μάλιστα με τρόπο αποτελεσματικό. Ένα τελευταίο θέμα τώρα σε σχέση με το κείμενό μου. Όπως σας είπα έχω 19 τροπολογίες. Από αυτές τις 19 τροπολογίες οι 12 είναι δικές μου και άλλες τρεις τις οποίες θα αποσύρω. Διότι σε πολλά σημεία γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τροποποιήσουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής σε αυτά τα τμήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Παρεμβάσεις. Ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να υποστηρίξω μέγα μέρο τη γνωμοδότηση, αλλά βρίσκω ότι έχει ένα πρόβλημα. Στη γνωμοδότηση και ορισμένε τροπολογίε, κατά τη γνώμη μου, ε, με περιττό τρόπο προβάλλεται το επιχείρημα της επικουρικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που λέει είναι ότι θα πρέπει να καθορίσουμε ε, ε, βασικές αρτηρίες και primary roads πέρα από τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και να εξετάσουμε τα πράγματα μέσα στην οδηγία για αυτοκινητοδρόμους και βασικούς δρόμους. Το πρόβλημα κατά την εξέταση της γνωμοδότησης προκύπτει από την παραπομπή στην, ε, στον ευρωπεριφερειακό, στην ευρωπεριφερειακή βάση δεδομένων που είναι κάτι όπως η Ευρωστάτ ίσως να μην την έχετε ακούσει όλοι πρόκειται για βάση δεδομένων που τη φτιάχνουν οι εθνικοί φορείς ε, κτηματολογίων και χαρτογράφησης. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων που προκύπτει από τα δεδομένα που παρέχουν εθνικοί φορείς και θα πρέπει να απηχεί τις απόψεις αυτών των εθνικών φορέων. Με ορισμένες από τις τροπολογίες υπάρχει ένα πρόβλημα ε, που προκύπτει επειδή κάτι έχει συμβεί σε μια συγκεκριμένη χώρα μέλος. Και απευθύνομαι στους Δανέζους, στους Δανούς μάλλον συναδέλφους μου, διότι αυτό που συνέβη στη Δανία είναι ότι υπήρξε μια μετακίνηση ορισμένων από τους δρόμους από την αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης σε τοπικές αρχές. Σε ό,τι αφορά λοιπόν πάντως τους Δανούς, αυτό τους προκαλεί ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την οδηγία που ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τους βασικούς δρόμους πέραν των αυτοκινητοδρόμων. Ίσως λοιπόν να υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα αυτό πρέπει να επιληθεί σε εθνική βάση και όχι ε, σε γενική ευρωπαϊκή βάση. Ε, δεν λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε εναρμόνιση, αλλά αυτό που λέω ότι αν εξετάζουμε την οδική ασφάλεια και εν ώψη της κυκλοφορίας, της κίνησης δηλαδή διευρωπαϊκά των ε, Ευρωπαίων πολιτών, θα πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία σε ζήτηματα ασφαλεία, αλλιώ θα αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οδηγία είναι να δημιουργήσει αυτή την κοινή βάση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλεια. Αυτή η ε, τράπεζα δεδομένων δεν χρησιμοποιείται παντού σε όλη την Ευρωπη... Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και το πιο κοντινό που έχουμε στο ανάλογό του που είναι η Ευρωστάτ. Υπάρχουν ορισμένε τροπολογίε οι οποίε εγώ θα αντιταχθώ, αλλά διότι οι τροπολογίε αυτέ κινούνται προ μια θέση επικουρικότητας που νομίζω ότι εν προκειμένου θα έπρεπε να αποφύγουμε. Θέλει να σχολιάσει ο εισηγητής. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ ένα σχόλιο. Συμφωνώ κύριε Μπορ. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το θέμα αυτό. Είναι δύσκολο λέει, να βρεθεί μια κοινή λύση. Εμείς είμαστε όμως εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών φορέων. Πρέπει λοιπόν να προτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα. και θα πρέπει να συμμετάσχουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην ανάπτυξη αυτών των υποδομών των οδικών. Υπάρχουν περιφερειακά project. Και αυτά τα project χρειάζονται συγκεκριμένες υποδομές. Η Άννα Μάγκιαρ, παραδείγματο χάρη από το ΕΛΚ, υπέβαλε μια τροπολογία, τροπολογία 4. που καταδεικνύει αυτό που σας είπα πάει προς αυτή κατεύθυνση νομίζω πρέπει να υποστηρίξουμε τέτοια πράγματα ευχαριστώ ο κύριος Άντερσεν έχει το λαό. ευχαριστώ πρόεδρε ο Άλμπερ Μπόρα μας παρουσίασε σαφέστατα ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μου και θέλω να αντιδράσω. Νομίζω ο εισηγητής μας λέει ότι με αυτήν την ευθύνη ε, για τους ε, δρόμους είμαστε υπεύθυνοι και για την ασφάλεια και θέλουμε να το διατηρήσουμε αυτό αυτό θέλουμε να πούμε είναι δική μας η ευθύνη. Αυτό λέμε στην πρόταση τροπολογίας μας. Θέλουμε να παραμείνει αυτό στις δικές μας τοπικές αρχές, την Δανία. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς θέλει το λόγο, όχι να περάσουμε στις τροπολογίες. Λοιπόν, τροπολογία παρθυμών 1. Εφόσον αγκριθεί η 1, τότε θα, θα ψηφίσουμε μόνο για το όρο others στο 2. Λοιπόν, παρθυμών 1, υπέρ, Ευχαριστώ. Κατά. Εντάξει, απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπάρχει εδώ μια προφορική τροπολογία, προφορική συμβαστική τροπολογία. Είναι θέμα βεβαίως και γλωσσικών εκδοχών εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε στα αγγλικά, όπως το βλέπετε στην οθόνη. Αυτή θα είναι η, η γλωσσική εκδοχή αναφοράς, η αγγλική, εφόσον εγκριθεί η συμβαστική αυτή τροπολογία. Ο κύριος Μπόρ θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ναι, προσπαθώ να διαβάσω βεβαίω τι λέει στην οθόνη, δεν βλέπω και πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπω ε, κάτι που με ενοχλεί. Να καθορίσουμε ποια τμήματα δρόμου. Τι λέμε εδώ, ότι υπάρχουν κάποια τμήματα του δρόμου που θα υπόκειται στην οδηγία και κάποια άλλα τμήματα του ίδιου δρόμου πιο κάτω ε, ε, δεν θα υπόκειται στην οδηγία. Ε, είναι αυτή η διατύπωση κάπως ε, χαλαρή και προβληματική. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά έτσι όπως είναι διατυπωμένο εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ και θα το καταψηφίσω. Δεν ξέρω αν ο κύριος συγκητής μπορεί να το εξηγήσει κάπως καλύτερα. Ακούστε, δεν βλέπω κι εγώ πολύ καλά. Θα μιλήσω ουγγρικά, που έχω και το ουγγρικό κείμενο. Ίσως να μην είναι καλή η αγγλική μετάφραση. Δεν ξέρω, έχετε κάποια πρόταση κύριε Μπόρ εσείς επί της διατύπωσης. Ναι, χρησιμοποιούμε, έχουμε συνηθίσει ο κύριος Μπόρ να μας ε, βρίσκει τη σωστή αγγλική διατύπωση που να διευκρινίζει τα πράγματα διότι και εμένα μου φαίνεται ότι κάτι πρέπει να αλλάξει δεν είναι καλή η αρχική αυτή η εκδοχή. Πρόεδρε, να προσπαθήσω να σας βοηθήσω και σας και τον εισηγητή. Στην τελευταία, η τελευταία φράση δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, θέλετε να συμμορφώνετε με την πρόταση, με, την αρχή, με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας πρόταση της Κομισιόν. Ωραία. Η προηγούμενη φράση όμως, εκεί έχετε βγάλει ε, το μέρος του δρόμου που καλύπτεται. Ε, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Όμως εδώ έχετε βάλει road section, τμήμα του δρόμου. Το τμήμα του δρόμου είναι ε, ένα τμήμα α έως β, ας πούμε, από την πόλη α στην πόλη β. Αυτό το τμήμα καλύπτεται από την οδηγία και μετά από την πόλη αυτή δεν καλύπτεται. Να φύγει ο όρος section τότε, λέει ο πρόεδρος. Τμήμα. Συμφωνεί ο εισηγητής να φύγει ο όρος section είναι κάπως καλύτερα έτσι τα πράγματα. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν επί της προφορικής αυτής ε, συμβαστικής τροπολογίας. Έχει φύγει ο όρος section, τμήμα. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται 5. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. εγκρίνεται 6 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά εγκρίνεται η 9 αποσύρεται και του, του, του εισηγητή υπαριθμών 10 άρα έχει αποσυρθεί 10 λοιπόν απλή 10 θέλει να πει κάτι ο κύριος Πεντεράντερς ναι αν κατάλαβα καλά η, η 8 εγκρίθηκε οπότε αποσύρεται η 10 πολύ ωραία εντάξει είναι σαφέστερα τα πράγματα έτσι απορρίφθηκε ε, μάλλον αποσύρθηκε και η 10 11 υπέρ Ευχαριστώ. Κατά. Πολύ ωραία, εγκρίνεται. 12 ...12R του εισηγητή αποσύρεται. Και η 12 τώρα. Ψηφίζουμε επί της 12. Ε, κατά. Η πλειοψηφία είναι κατά, όπως βλέπετε, οπότε απορρίπτεται. Του εισηγητή 13R υπέρ κατά εγκρίνεται καταπίπτουν οι 13 και οι 14 15 υπέρ κατά λοιπόν για να το ξαναδούμε 15 ε, υπέρ κατά Μάλιστα, ηλεκτρονική ψηφοφορία για να το επαληθεύσουμε. Κάποιοι το σκέφτηκαν από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, για να δούμε. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται για μία ψήφο. 16 υπέρ κατά εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά ξανά υπέρ Κατά. Η πλειοψηφία είναι κατά. Απορρίπτεται για μία-δύο ψήφους. Για μισή ψήφο. 18 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε επί του συνόλου της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές όχι πολύ ωραία ομόφωνη έγκριση ευχαριστώ κύριε Σιγητά πολύ ωραία εργαστήκαμε σκληρά συνεχίζουμε αύριο το πρωί Καλό βράδυ. Πέρα στη συνεδρίαση συνεχίζουμε αύριο στις 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ. Τέλος για σήμερα. Γεια σας και από εμάς.